η έναρξη της Συνόδου, η οποία σταμάτησε στις 18 Ιουλίου τρέχοντος. Έχω κάποιες ανακοινώσεις. Μία που με, μου προκάλεσε μεγάλη θλίψη. Πέθανε ο Αντρέι Μπράτφορντ από την Πορτογαλία, ευρωβουλευτής. Χάσαμε το ζήλο του, εμείς, το κόμμα του, η χώρα του. Πολύ νέος, 48 χρονών μόλις. Αφιερωμένη η ζωή του ήταν στην υπεράσπιση της δημοκρατίας, στην αξιοποίηση της πολιτικής αυτονομίας της, στις Αζόρες και όλοι τον ήξεραν ως ένα πολύ ευγενικό άνθρωπο, πάρα πολύ εφραδή, πάρα πολύ καλλιεργημένο και ακέραιο ηθικά. Εξελέγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα και αντιμετώπισε μια νέα πρόκληση, πολύ σημαντική, εκφράζω την προσωπική μου θλίψη για το χαμό του Αντρέ απέναντι στην οικογένειά του, στους σοσιαλιστές, στους οποίους ανήκε και σε ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει και ακόμη μια δύσκολη ανακοίνωση που πρέπει να κάνω. Την περασμένη εβδομάδα έγιναν σοβαρότατες πλημμύρες στην Ευρώπη. Ε, χτύπησαν ένα μεγάλο κομμάτι του κέντρου της Ισπανίας και του, της νότιας ανατολικής Ευρώπης. Και ξεχύλισαν πάρα πολλοί ποταμοί στο Αλικάντε, στην Βαλένθια, στην Μούρθια, Γρανάδα, ε, στη Μαδρίτη. Έχασαν κάποια άτομα τις ζωές τους. Κάποια άτομα χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τι ε, οικίε τους. Δεκάδες χιλιάδες εξ ονόματος του Ευρωκοινοβουλίου θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μας και τα συλληπιτήρια για τα θύματα στις οικογένειε τους και την απόλυτη δέσμευσή μας και αλληλεγγύη μας για τους πλημμυροπαθείς. Θα ήθελα να αναγνωρίσω επίσης την αέναη και ακάματη δουλειά που κάνουν οι σωστικές υπηρεσίες, τα ειδικά σώματα, οι εθελοντές, οι οποίοι συμμετέχουν στην ζώνη αυτή και στις εργασίες διάσωσης. Εξ ονόματος του συναδέλφου και των θυμάτων της Ισπανίας και για να δείξουμε το πόσο κοντά είμαστε στις οικογένειές τους, θα ήθελα να σηκωθείτε όλοι και να τηρήσουμε ενός λεπτού Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Πύρη ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Ή συνάδελφος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ανταλλαγή φυλακισμένων ανάμεσα, κρατούμενων ανάμεσα στην Ουκρανία και την ε, Ρωσία. Ε, απελευθερώθηκαν 24 ε, πεζοναύτες από την Ουκρανία. Νομίζω όμως ότι συμφωνούμε ότι αυτή η ανταλλαγή δεν θα πρέπει να είναι η βάρος ε, της δικαιοσύνης για τα θύματα του ΜΗ-17. Το ότι παραδόθηκε ο κύριος Τέμαχ στη Μόσχα ήταν επώδυνο όχι μόνο για τα θύματα αλλά και για τις οικογένειες. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ότι φυσικά είμαστε αλληλέγγυοι απέναντι στην Ουκρανία. Περιμένουμε όμως να ανταποκριθεί στο ψήφισμα του, ε, των Ηνωμένων Εθνών και να ε, βρει αυτούς που βρίσκονται πίσω από την κατάρριψη του αεροσκαφους μη Mi-17. Ευχαριστώ. Τα πρακτικά της 16ης ε, Ιουλίου τα έχουμε μοιράσει. Έχετε παρατηρήσει από αυτόν, πάνω στην τελευταία δηλαδή ολομέλεια. Ο κύριος Παπαδάκης παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή η Κύπρος βρίσκεται περικυκλωμένη από τον πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας. Την ίδια στιγμή έχουν εγκαταστήσει πλατφόρμες για ανακάλυψη υδρογοναθράκων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου που είναι και ευρωπαϊκή. Ταυτόχρονα ο κύριος Τσαβούσογλου απειλεί καθημερινά με επικισμό της πόλης της αμχώστου όπου προστατεύεται από ψηφίσματα των ηνωμένων εθνών και του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο οφείλει να πράξει. το ευρωπαϊκό συμβούλιο έχει αποφασίσει τη λήψη κυρώσεων κατά της τουρκίας οφείλει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Ε, Υπάρχουν παρατηρήσεις για τα πρακτικά. Αυτό είχα ρωτήσει. Εάν όχι, τα πρακτικά εγκρίνονται. Εν συνεχεία, μετά το θάνατο του κυρίου Μπράτφορντ και το διορισμό του κυρίου Γκαλτιέρη ως Υπουργό Οικονομικών της ε, Ιταλίας, ε, χειρεύει η θέση του από τις 19 Ιουλίου μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου του, χείρεψε μάλλον, μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου του 19. Οι αρμόδιες αρχές της Δανίας, άλλη ανακοίνωση, μου είπαν ότι ο κύριος Μαριάν Δίν αντικαθιστά τον Ιέπε Κόφορντ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις 2 Ιουλίου του 2019. Και οι αρμόδιες αρχές της Πορτογαλίας μου ανακοίνωσαν την εκλογή του Ευρωβουλευτή της Ιζαμπέλ Καρβάης που αντικαθιστά το κύριο Μπράτφορντ από τις 3 Σεπτεμβρίου του 2019. Κατοσορίζω τους νέους συναδέλφους και έχουν κάθε δικαίωμα να απολαμβάνουν όλων των προνομίων του Κοινοβουλίου. Η νομική υπηρεσία ε, εξέτασε τον κύριο Άντσο και τον Αρία Σατσεβερία και επικύρωσε την, το διορισμό τους από τις 4 Απριλίου και 21 Μαΐου του 2019 μέχρι το τέλος ε, της τελευταίας ε, κοινοβουλευτικής Υπάρχουν αντιρρήσεις. Πολύ ωραία, επικυρώνονται όλες αυτές οι, όλοι αυτοί οι διορισμοί. Εν συνεχεία, το ΕΛΚΑ, οι σοσιαλιστές, οι πράσινοι, ID, ECR, καθώς και οι μη εγγεγραμμένοι, μου ζήτησαν να, να αναφέρω κάποιες αποφάσεις ό,τι αφορά τους διορισμούς στις ε, αντιπροσωπείες και επιτροπές. Αυτές οι αποφάσεις θα μπουν στα πρακτικά της σημερινή συνεδρίασης και θα τεθούν σε ισχύ την ημερομηνία την ίδια. Οι Γιούρι και Τραν ε, τροποποίησαν κάποια κείμενα με βάση το 241.4 του κανονισμού αυτές οι τροποποιήσεις εγκρίνονται εκτός και αν μέσα σε 24 ώρες από την ανακοίνωση μία πολιτική ομάδα ε, ή ένας αριθμός ε, ευρωβουλευτών ε, που φτάνει στο κατώτατο όριο του κατοφλίου ζητάει το αντίθετο. Οι τροποποίησεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας και θα αναφερθούν και στα πρακτικά της τρέχουσας συνόδου. Επίσης, η Επιτροπή Πολιτισμού αποφάσισε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις διαθεσμικές πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου με βάση το άρθρο 42 του κανονισμού. Οι θέσει του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση είναι η εντολή για αυτές τις διαπραγματεύσεις και υπάρχει στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας και όλα αυτά θα δημοσιευτούν στα πρακτικά της σημερινής συνόδου. Άλλη ανακοίνωση αφορά την εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Στις 30 Αυγούστου του 19 δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα μία πρόσκληση για να υποβληθούν υποψηφιότητες για να εκλεγεί ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Η προθεσμία για αυτές τις υποψηφιότητες είναι η 30 Σεπτεμβρίου του 19. Στις 4 Σεπτεμβρίου λάβατε από μένα ένα email με περαιτέρω ε, πληροφορίες με βάση το 231 παράγραφος 2 του κανονισμού κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να υποστηρίζεται από τουλάχιστον 40 ευρωβουλευτές που, είναι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη. Κάθε ευρωβουλευτής θα μπορέσει να στηρίξει μόνο μία υποψηφιότητα. Αν ένας ευρωβουλευτής ε, στηρίξει περισσότερους υποψήφιους, η, υποψηφι... η στήριξη του αυτή είναι άκυρη αυτή τη στιγμή η υποψηφιότητα πάει στον Πρόεδρο, δεν μπορεί να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε υπογραφέ στήριξη. Όταν ολοκληρωθεί η προθεσμία για την ε, παρουσίαση των ε, υποψηφιοτήτων, θα εγκρίνουμε την, ε, την ισχύ των υποψηφιοτήτων και θα πάει στην Επιτροπή Αναφορών που θα γίνουν σχετικές αναφορές αρχές Δεκεμβρίου. Μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ευρωβουλευτές. Η εκλογή του νέου διαμεσολαβητή προβλέπεται για την Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Και τώρα περνάμε στην ημερήσια διάταξη. Η οριστική ημερήσια διάταξη εγκρίθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου από τη διάσκεψη των Προέδρων με βάση το άρθρο 157 και έχει μοιραστεί. Ας δούμε κάποιες αλλαγές. Μετά από τις διαβουλέσεις με τις πολιτικές ομάδες, θα ήθελα να σας παρουσιάσω την εξής πρόταση τροποποίησης του σχεδίου μερίσιας διάταξης που αφορά την Τρίτη. Ο τίτλος της δήλωσης της Κομισιόν για την κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη της Νόδου Κορυφής του ΟΗΕ για τη δράση για το κλίμα στη Νέα Υόρκη θα πρέπει να αλλάξει και να γίνει προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής για τη δράση για το κλίμα και τη Συνόδου για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Νέας Υόρκης. Αντιρρήσεις. Εάν δεν υπάρχουν, αυτές, αυτή η τροποποίηση εγκρίνεται. Πάντα για την Τρίτη, η Πράσινη και η Γκουε ζήτησαν η συζήτηση για τη δήλωση του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δασικές πυρκαγιές στην Αμαζονία να ολοκληρωθεί με ένα ψήφισμα που θα ψηφιστεί το πρωί της ε, Πέμπτης. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Λάμπερτς, πρόεδρο Λάμπερτς, για να παρουσιάσει το αίτημα αυτό εξ ονόματος των πράσινων. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Συνάδελφοι, αυτό που συμβαίνει στον Αμαζόνιο δεν τον και είναι, μιλάμε για εναιστώτα χρόνο, είναι μαζικές ε, εκτεταμένες πυρκαγιές. Είναι τεράστιο πρόβλημα πανκοσμίας εμβέλειας. Είναι απόλυτα θεμητό εμείς να συζητήσουμε και να τοποθετηθούμε. Αυτό που φοβώ, φοβάμαι είναι ότι αν απλώς συζητήσουμε την κατάσταση, χωρίς να φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα, βλέπω ήδη κάποια άτομα τα οποία βρίσκονται εκεί στην Αμαζονία και κάνουν ε, big business ε, θα τρίβουν τα χέρια του και θα λένε η Ευρώπη ένα τίγρη, ο οποίο δεν δαγκώνει. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση με ένα ψήφισμα, έτσι να τελειώσουμε, που θα λέει ποια είναι η άποψή μα και τι συνέπειε τι οποίε θεωρεί ότι υπάρχουν ε, κατά την άποψή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η Βραζιλία δεν κάνει τίποτα, μείνει αδρανή. Δηλαδή, αν συνεχίσει να λέει δεν υπάρχει κανένα απολύτω πρόβλημα και ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ασχολούνται με τα δικά του θέματα. Νομίζω ότι το θέμα του Αμαζονίου δεν είναι μόνο πολιτιστική κληρονομιά, ε, μας αφορά όλους, είναι βασικό στοιχείο για την ε, καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής και δεν μπορούμε να μην κάνουμε τίποτα. Σας ζητώ λοιπόν να ψηφίσουμε την Πέμπτη ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο θα λέει ξεκάθαρα ποιε είναι οι συνέπειε που θέλουμε, ε, που βλέπουμε ότι υπάρχουν από την κατάσταση σήμερα. Υπάρχουν ε, αντίθετε απόψει. Λέει ο Πρόεδρο. Κάποιο που θέλει να πάρει το λόγο για να υποστηρίξει την αντίθετη θέση. Όχι, δεν βλέπω κανένα. Άρα ψηφίζουμε το αίτημα με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Όχι, όχι, δεν ψήφισαν όλοι. Φρένο. Τώρα όμως ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Επομένως, δεν αλλάζει η μερίσια διάταξη. Πάντα για την ε, τρίτη, η ΓΚΟΕ και ID. Ποιο είναι το πρόβλημα? Κυρία Κρέτου, ποιο είναι το πρόβλημά σας? Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Μικρόφωνο. Με μικρόφωνο κατά προτίμηση. Πολύ ωραία το καταγράφουμε. Για την τρίτη. Οι ομάδε ID και GUE ζήτησαν η συζήτηση και ψηφοφορία για την έκθεση του κυρίου Γκουαλτιέρη για το διορισμό του, της Προέδρου του Ευρωπαϊ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ να αναβληθεί στην πρώτη ολομέλεια του Οκτωβρίου, ούτω ώστε να μπορέσει η κυρία Λαγκάρντ να παραστεί. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπάι για να παρουσιάσει το αίτημα εξ ονόματος της ομάδας ID. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση και η ψηφοφορία προβλέπεται μαζί με την κυρία ε, Λαγκάρντ αύριο. Δεν ε, το κανονίσαμε χθες. Ε, το, το ξέραμε εδώ και πολύ καιρό. Η κυρία Λαγκάρ τελευταία στιγμή μα είπε ότι έχει υποχρεώσει ανηλυμένε στη Ουάσιγκτον και δεν θα είναι παρούσα. Ορισμένοι λένε ότι αρκεί η ακρόαση τη ενώπιον τη ε, Επιτροπή ΕΚΟΝ. Δεν αρκεί φυσικά αυτό. Πολύ συχνά θεωρείτε ότι εδώ πέρα έρχεται και καταγράφεται οι απόψει σα. Οι αποφάσει λαμβάνονται αλλού και με κάθε διαφάνεια. Σήμερα προτείνουμε και την ταπείνωση προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το μοναδικό θεσμικό όργανο το οποίο είναι νόμιμο γιατί εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία. Φυσικά η διακυβέρνηση της ΕΚΤ είναι εκ των όνων κάνευ θέμα. Είναι πολύ σημαντικό η πολιτική καταπολέμηση του πληθωρισμού ενό ε, ισχυρού ευρώ είναι σημαντικό για τις εξαγωγές Ευρώπης, είναι σημαντικό για την οικονομία και βεβαίω θα θέλαμε η κυρία Λαγκάρτ τουλάχιστον έχει την ευγένεια να έρθει εδώ και να συζητήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί. Και ζητάμε ακριβώς γι' αυτό ε, επειδή θα μπορέσει να έρθει αύριο, να αναβληθεί η συζήτηση αυτή και η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος ο οποίος θέλει να πει κάτι αντίθετο. Όχι. Ο κ. Λάμπερτ ζήτησε το λόγο. Πρόεδρε, δεν συμφωνώ σε καμία περίπτωση με τα επιχειρήματα του κ. Μπέι. Αναφέρει τη διαδικασία. Να υπενθυμίσω ότι η διαδικασία προβλέπει μία ακρόαση της υποψηφίου από την αρμόδια επιτροπή που είναι καθήλυνα αρμόδια. Έτσι. Δηλαδή της Επιτροπής ΕΚΟΝ έγινε αυτή η ακρόαση, ήταν στη διάθεση ε, της Επιτροπής αυτής, συζήτησε επί ώρες μαζί μας, επομένως σεβαστήκαμε τους κανόνες και εν συνεχεία θα πρέπει να ε, γίνει η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Σας τονίζω επίσης το εξής, ότι η κυρία Λαγκάρτ είπε ότι καταρχά δεν είχε κανένα πρόβλημα να έρθει στην Ολομέλεια. Δεν την υποχρεώνει όμω ο κανόνα να έρθει ντε και καλά στην Ολομέλεια. Εγώ νομίζω ότι αν θέλει να υποφεληθεί το Κοινοβούλιο να βελτιώσει το προφίλ του και να κάνει με μία συζήτηση με την υποψήφια της έκτη είναι πολύ σωστό. Νομίζω όμως ότι η κυρία Λαγκάρτ είχε πολύ ε, θεμητούς λόγους να είναι στη Ουάσιγκτον. Ε, δεν θεωρώ ότι είναι έλλειψη σεβασμού προς εμάς. Αν όμως αύριο η συζήτηση δεν γίνει παρουσία της, δεν έχει νόημα να γίνει. Για τελείως διαφορετικούς λόγους λοιπόν από του κυρίου Μπέι, νομίζω ότι θα έχει νόημα, αλλά μόνο και μόνο αν γίνει συνενετικά εντός του Κοινοβουλίου, να κάνουμε την συζήτηση και την ψηφοφορία τον Οκτώβριο, στην πρώτη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Εάν θέλετε όμως να το παρουσιάσετε ως ε, μία πράξη αντίσταση απέναντι στην κυρία Λαγκάρτ δεν συμφωνώ. Ο λόγο που το κάνουμε είναι για το στάτου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το να κάνουμε συζήτηση για το διορισμό τη κυρία Λαγκάρτ χωρί την κυρία Λαγκάρτ δεν έχει κανένα νόημα. Αν θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση για την ε, νομισματική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Αυτή η, αυτό το αίτημα δεν υποβλήθηκε στη διάσκεψη των ε, Προέδρων και δεν υπάρχει αυτό το αίτημα ενώπιον μα σήμερα. Δεν είναι αυτό το θέμα μα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ομπρή επίσης θέλει να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Γκουε Επίση, το άρθρο 130 του κανονισμού που λέει ότι ο διορισμός της, του Προέδρου της ΕΚΤ θα πρέπει να γίνει δύο μήνε μετά την ακρόαση. Η ακρόαση τη έγινε στι 4 Σεπτεμβρίου. Έχουμε μέχρι τι 4 Νοεμβρίου, λοιπόν, για να διορίσουμε τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχουμε δύο ακόμα ολομέλειε τον ε, Οκτώβριο που θα μπορούσαν να μα επιτρέψουν να κάνουμε μια συζήτηση ήρεμη, σωστή, υγιή με την κυρία Λαγκάρντα. Τι, τι μπορούμε να περιμένουμε ω νέα νομισματική πολιτική από τη νέα πρόεδρο τη ΕΚΤ. Θυμάμαι ότι στην ακρόασή τη είπε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα άκουγε επί χρόνια τις αγορές. Καιρό είναι, λέει, να ακούσει ε, τους ευρωπαϊκούς λαούς. Εδώ εκπροσωπούμε εμείς τους ευρωπαϊκούς λαούς. Είναι και καινή ώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μα ακούσει και εμά. Επί καιρό άκουγε μόνο τι αγορέ. Δεν μπορώ να φανταστώ, φίλοι και φίλε και συνάδελφοι, ότι λέτε όχι σε μια συζήτηση παρουσία της κυρίας ε, όταν ξέρουμε ότι ο διορισμός της είναι πάρα πολύ σημαντικός ε, για μια πολύ σημαντική πολιτική, για τον πλανήτη κτλ. Σας ενθαρρύνω λοιπόν να γίνει μια συζήτηση παρουσία της κυρίας Λαγκάρντ. Ε, παρουσιάστηκε το αίτημα, εντάξει, θα πρέπει να ψηφίσουμε με ονομαστική κλίση. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Επομένως, δεν αλλάζει η μερίσια διάταξη. Υπάρχει ένα ηλεκτρονικό πρόβλημα. Έσβησε η οθόνη με τις α, ψήφους, λέει ο πρόεδρος. Με τον αριθμό των ψήφων. Ήθελα να διαβάσω το αποτέλεσμα. Παρακαλώ. Sul tabellone principale i voti ε, Δεν κατάλαβαν οι βουλευτές γιατί οι αντίθετες ψήφοι, ε, οι ψήφοι κατά δηλαδή, εμφανιζόταν ως αποχές πάνω στην οθόνη. Λοιπόν, υπέρ 175. Κύριε Μπούλμαν, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Υπάρχει η εντύπωση στην αίθουσα ότι υπήρξε ηλεκτρονική σύγχυση όσον αφορά το αίτημα των πρασίνων ε, σχετικά με το ψήφισμα. Δεν ήταν σαφές εάν το αποτέλεσμα αντιστοιχούσε στο πραγματικό αποτέλεσμα. Παρακαλούμε να επαναλάβετε την ψηφοφορία, διότι ε, δεν επιτρέπεται τεχνικά προβλήματα να αλλάξουν το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα για τη συζήτηση για την έκθεση Γκουαλτιέρη είναι υπέρ 175 κατά, για κατά 2,74 ε, και 10 αποχές. Ψήφι κατά 274. Επομένως, δεν αλλάζει η μερίσια διάταξη. Σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα για το αίτημα, για τη συζήτηση για την Αμαζονία, έχουμε υπέρ 194, κατά, κατά 228 και 13 εποχές. Για την Τρίτη, η ομάδα Renew ζήτησε το ψήφισμα που ολοκληρώνει τη συζήτηση για τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Κομισιόν για τις παρεμβάσεις και παρεμβολές ε, ξένων σε εκλογές και την παραπληροφόρηση σε δημοκρατικές ε, εθνικές εκλογές ή ευρωπαϊκές εκλογές να γίνει την πρώτη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Θα δώσω το λόγο σε όποιον θέλει να υποστηρίξει αυτό το αίτημα. Παρακαλώ, ποιος είναι. Ποιος θα μιλήσει υπέρ. Ουδής. Η κυρία Ίνθελτ Um, είναι αρκετά σαφές. Ε, μπορούμε να έχουμε τη συζήτηση κατά τη γνώμη μας. Ε, το σχέδιο ψηφίσματος όμως απαιτεί περισσότερο χρόνο διότι είναι επίμαχο και δέστη το θέμα. Ε, ας έχουμε λοιπόν συζήτηση και να έχουμε ψήφισμα στην επόμενη σύνοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ιντβελτ. Ποιος θέλει να τοποθετηθεί με την αντίθετη θέση. Πολύ χαίρομαι που βλέπω μεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο που θέλει να τεθεί το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη, διότι ήταν αίτημα του S&D. Θα πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε ενωμένοι και μπορούμε, εάν έχουμε ειδική επιτροπή την επόμενη εβδομάδα, να βάλουμε το θέμα αυτό. Ελπίζουμε όμως το αποτέλεσμα να μην είναι να ε, ξεχαστεί το θέμα. Συζήτηση αύριο λοιπόν και ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα. Ακούσαμε λοιπόν τις δύο απόψεις, υπέρ και κατά. Θα ψηφίσουμε λοιπόν το αίτημα τώρα με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Όχι, συγγνώμη, διανατάσσεως χειρός. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πολύ ωραία. Περνάμε στην Ολομέλεια της Τετάρτης. Το ΕΛΚΑ ζήτησε η συζήτηση για τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Κομισιόν για τη σημασία της Ευρωπαϊκής ημέρας μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης να ολοκληρωθεί με ένα ψήφισμα το οποίο θα ψηφιστεί την Πέμπτη. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκάλερ για να παρουσιάσει το αίτημα του ΕΛΚ. Παρακαλώ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 Ντάλι θα κάνει μια δήλωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, θα ήθελα να τονίσω ότι διατηρούμε, θέλουμε να διατηρήσουμε τον τίτλο στην ε, Ολομέλεια ε, και δεύτερον, θα ήθελα στην ε, πρώτη ολομέλεια του Οκτωβρίου να έχουμε ψήφισμα, διότι είναι πολύ ευαίσθητο και σημαντικό θέμα. Θέλουμε αρκετό χρόνο να εκπονήσουμε ένα σωστό ψήφισμα. Ευχαριστώ. E πολύ ωραία. Θα ψηφίσουμε το αίτημα. Ακούσαμε τον κύριο Γκάλερ και τι μας είπε και τώρα θα ψηφίσουμε με ονομαστική κλίση. Πέρας της ψηφοφορίας. Θα διαβάσω εγώ, γιατί αλλιώς θα τα μπερδέψουμε όλα. Υπέρ, ψήφι υπέρ. Ή μάλλον, ψήφισαν 443 βουλευτές. Υπέρ 234, κατά 178, 31 αποχές. Επομένως, η πρόταση αυτή εγκρίνεται. τώρα, πάντα για την ε, Τετάρτη, την Ολομέλεια της Τετάρτης. Με βάση το άρθρο 314 της ε, Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ένωσης, προτείνω μετά από την παρουσίαση από το Συμβούλιο να γίνει μια πλήρη συζήτηση. Αυτό το λέω γιατί οι πράσινοι είχε κάνει ένα αίτημα, είχαν κάνει ένα αίτημα Η παρουσίαση από πλευράς του Συμβουλίου, δηλαδή, να αφορά το γενικό προϋπολογισμό, την άσκηση του 2020, αλλά προτείνω όχι μόνο να ακούσουμε την παρουσίαση του Συμβουλίου, να γίνει και μία πλήρη συζήτηση. Μία συζήτηση στην Ολομέλεια. Ναι, ασχοληθεί και η Ολομέλεια με αυτό το θέμα, δηλαδή, συζητώντας το παρατηρήσεις. Άρα εγκρίνεται. Αυτό. Ευχαριστώ. Σταματούμε εδώ, λοιπόν, περιμένοντας την επόμενη συζήτηση. Αλλάζει λοιπόν με τα όσα είπαμε ε, η ημερήσια διάταξη. Το πρώτο σημείο τώρα. Ακούμε τη δήλωση της Κομισιόν για την κατάσταση των ευρωπαϊκών δασών. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το λόγο έχει ο κύριος Αρίας Κανιέτη. Καλό τους συναδέλφους που θέλουν να βγουν, να βγουν ήσυχα. Ο Επίτροπος έχει το λόγο. Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να εκφράσει την αλληλεγγύη της απέναντι στους πληγέντες ε, μετά από τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν διάφορες περιοχές της Ισπανίας. Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου ε, απέναντι στι στις οικογένειες των πλημμυροπαθών και να σας ευχαριστήσω όλους. Επίτροπε, Επίτροπε διακόπτη πρόεδρος ζητώ συγγνώμη κύριε Επίτροπε. Θέλουμε να ακούσουμε αυτά που έχετε να πείτε. Παρακαλώ λοιπόν τους συναδέλφους να αποχωρήσουν ήσυχα από την αίθουσα. Κύριε Επίτροπε, να περιμένουμε ένα λεπτό καλύτερα. No, please, we'll hold. Please leave the chamber quietly, Σας παρακαλώ, αποχωρήστε ήσυχα από την αίθουσα, συνάδελφοι. Ξεκινάμε τη συζήτηση και ο Επίτροπος προσπαθούσε να μιλήσει. Επιτρέψτε μας να συνεχίσουμε. Ζητώ συγγνώμη κύριε Επίτροπε που σας διακόψαμε. Μπορείτε νομίζω να ξεκινήσετε πάλι από την αρχή. Παρακαλώ αποχωρήστε ήσυχα από την αίθουσα. Thank you. Thank you, Madam President. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελα να εκφράσει την αλληλεγγύη της απέναντι στους πλημμοπαθείς για τις πρόσφατες ε, πλημμύρες που έπληξαν διάφορες ισπανικές περιοχές. Θα ήθελα να διαβιβάσω στους, στις οικογένειες πλημμυροπαθών την αλληλεγγύη μας και να ευχαριστήσω τις αρχές, τους εθελοντές, τις σωστικές αρχές που δεν φύστηκαν κόπον για να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 support for the prevention of damage to forests caused by fires natural disasters and extreme events and for the restoration of production potential is also available to member states through the European Union. Ζητήματα που χρηματοδοτούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την περίοδο του 2014 έως το 2020 είχαμε μια, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό 9,7 ε, εκατομμύρια συγκεκριμένα για προστασία και ε, περαιτέρω για την ε, πρόληψη τέτοιων καταστροφών με ε, περαιτέρω κονδύλια σε ό,τι αφορά και την καλύτερη διαχείριση. Ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ε, Προστασία των Δασών παρέχει περαιτέρω υποστήριξη έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότερα μέσα στη διάθεσή μα για την αντιμετώπιση των ε, πυρκαγιών στα δάση. Και αυτό ο μηχανισμό έχει, για παράδειγμα, στραφεί προ τη δημιουργία και ενό αποθεματικού έτσι ώστε να υπάρχουν και περισσότερα ελικόπτερα πυρόσβεση. Επίση, ε, ε, επενδύουμε περισσότερο και στον τομέα τη έρευνα και τη καινοτομία, στον δασοκομικό τομέα και στον τομέα των δασών, ε, ιδιαίτερα εστιάζοντα στην προστασία των δασών και στην αύξηση τη ανθεκτικότητα των δασών. Και θεωρούμε πω ο προπολογισμό για αυτέ τι πρωτοβουλίε έρευνα και καινοτομία θα αυξηθεί σημαντικά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πολύ και περνάμε στον πρώτο ομιλητή των πολιτικών ομάδων, ο κύριος Πέτερ Λίσα από το ΕΛΚ. Δύο λεπτά. Εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τα δάση για μας εδώ στην Ευρώπη είναι σημαντικός προστάτης του κλίματος και αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν το διαχειριζόμαστε σωστά και ε, το ξύλο μπορεί να αντικαταστήσει άλλα προϊόντα όπως είναι ο χάλιβας και το τσιμέντο. Είναι επίσης σημαντικός οικονομικός τομέας και για την βιοπικιλότητα. Το δάσος σε πολλές χώρες της Ευρώπης βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Στη Τσεχία, τη Σλοβακία, τη Γαλλία, την ε, Γερμανία και τη Σκανδιναβία. Και αιτία είναι η ακραία ξηρασία των τελευταίων δύο ετών και η εξάπλωση βλαβερών οργανισμών όπως είναι ο βλαστοφάγος και βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω της αλλαγής του κλίματος ε, το δάσος ε, και γι' αυτό θα πρέπει ο καθένας ε, στο, στα διάφορα επίπεδα και στα κράτη-μέλη και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση όπου έχουμε αρμοδιότητες πρέπει να βοηθήσουμε. Πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της ε, οικονομικής υποστήριξης από, την ε, δεύτερη, από τον δεύτερο πυλώνα της ε, γεωργικής πολιτικής. Δεν μπορούμε όμως να μειώσουμε σημαντικά το, τα ποσά του δεύτερου πυλώνα. Χρειάζεται όμως επίσης να εκπονήσουμε κανόνες και στον τομέα του ανταγωνισμού και αλλού. Πρόκειται για μια καταστροφή, πρέπει όλοι να την συνειδητοποιήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να εκπονήσουμε κανόνες, αλλά όχι με γραφειοκρατικό τρόπο. Αγαπητοί συνάδελφοι, δυστυχώ ε, στην ημερήσια διάταξη έχουμε μόνο συζήτηση. Το ΕΛΚΙ ήθελε και ψήφισμα. Τι επόμενε ε, μέρε λοιπόν μπορούμε να συζητήσουμε ώστε να έχουμε και συγκεκριμένο αποτέλεσμα όπω ε, ένα ψήφισμα στην επόμενη Ολομέλεια. Πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι μας ενδιαφέρουν τα δάση και στηρίζουμε όλου όσου ενδιαφέρονται γι' αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αντριώ, ένα λεπτό από το S&D. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να μην κρυβόμαστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει ρόλο στην παγκόσμια αποδάσωση. Είμαστε εν μέρη υπεύθυνοι διότι εισάγουμε τεράστιες ποσότητες ξυλίας από όλο τον κόσμο. Καταναλώνουμε πολλά προϊόντα που περιέχουν φινικέλαιο. Κάποιες χώρες όπως η Γαλλία συνεχίζουν να προωθούν τα βιοκάψιμα και το φινικέλαιο παρά τις καταστροφικές συνέπειές τους. Ε, είναι πιο βλαβερά από το ντίζελ για το περιβάλλον. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε την κατάσταση, πρέπει να εκτιμήσουμε τους σπόρους από τα δάση. Πρέπει να έχουμε σαφείς κανόνες για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των δασών και μια προσωπική παρατήρηση. Θα ήμασταν πολύ πιο αξιόπιστοι εάν στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με τις χώρες Μερκοσούρ, για παράδειγμα, είχαμε δεσμευτικές ρήτρε ε, για το σεβασμό στο περιβάλλον. Ο κύριος Τόρβαλς. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε. Τα δάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μερικές φορές βρίσκονται σε καλή κατάσταση, άλλες φορές όχι. Και ο λόγος ε, γι' αυτό είναι ότι δεν έχουμε ένα γενικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δάση. Έχουμε δάση διαφορετικά και μερικά τα πάνε καλά, αλλά όχι τόσο. Και για να καταλάβουμε πού βρίσκεται το πρόβλημα, θα πρέπει να δούμε τι έγινε και στον Καναδά και στη Ρωσία. Και στις δύο αυτές χώρες ε, υπήρξαν εκτενείς πυρκαγιές και ε, η οικολογική ισορροπία των δασών ε, έχει ήδη καταστραφεί. Εάν έχουμε φυσικές ε, δασικές πυρκαγιές, δεν υπάρχει τρόπος να κατασβεστούν. Δεν υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό. Και γι' αυτό το πρόβλημα γίνεται μόνιμο. Στη Ρωσία τον Ιούλιο 4 εκατομμύρια εκταρίων καταστράφηκαν από πυρκαγιά και κανείς δεν είχε καν πρόσβαση στα μέρη αυτά. Χρειαζόμαστε σωστή διαχείριση των δασών. Ο Ντόναλτ Τραμπ είπε ότι θα πρέπει να ε, φροντίσουμε το υπέδαφος των δασών. Ε, αυτό δεν αποτελεί λύση. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και οι βλαβεροί οργανισμοί, όπως για παράδειγμα ο βλαστοφάγος, αποτελεί πρόβλημα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έιχαουτ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή για τα ευρωπαϊκά δάση. Συνήθως ε, μιλάμε για τα δάση εκτός της Ευρώπης, αλλά σημαντικό είναι να συζητήσουμε και την κατάσταση των ευρωπαϊκών δασών ιδιαίτερα διότι τα δάση είναι ζωτική σημασία για το κλίμα, είναι κατά βόθρα του άνθρακα και για την βιοπικιλότητα. Και στα δύο αυτά τα ευρωπαϊκά δάση δεν τα πάνε πολύ καλά. Ε, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 40% προέρχεται από βιομάζα. Και ε, στην ε, αναφέρεται ότι περιμένουμε μέχρι το 2030 να μειωθεί η καταβόθρα του διοξιδίου του άνθρακα, κάτι που έχει το ίδιο αποτέλεσμα με αύξηση των εκπομπών. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε το θέμα των δασών και της αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης, ο Οργανισμός Περιβάλλοντος ε, λέει ότι ε, στις περιοχές ε, Natura 2000 μόνο το 25% των δασών ε, βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τις καταβάθμιση του άνθρακα μέχρι το 2030 για να βελτιώσουμε τα δάση προς όφελος και του κλίματος και της βιοπικιλότητας. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά. Ο κύριος Χακαράινεν από την ομάδα ID. Micro, please. Thank you arvoisa puhemies Ευχαριστώ. Ο κύριο ε, Τόρβαλς ε, ξεκίνησε μια σκέψη την οποία θα ήθελα να συνεχίσω εγώ. Ε, στη Φιλανδία λοιπόν έχουμε επενδύσει στην δασοκομεία και γενικά στη διαχείριση των δασών εδώ και 100 χρόνια και ω συνέπεια αυτών των πρωτοβουλειών τα δάση μας αυξάνονται όλο και περισσότερο ακριβώς λόγω αυτών των πρωτοβουλίων που αναλάβαμε. Και ε, έχουμε για παράδειγμα κάποιες... Έχω ένα δικό δίκτυο μέσα στα δάση το οποίο βοηθάει στη διαχείρισή τους. Επίσης με αυτόν τον τρόπο είναι πιο εύκολο να καταπολεμήσουμε τυχόν πυρκαγιές. Βρισκόμαστε δηλαδή στο επίπεδο της σήμερα ημέρα της Σουηδίας, ε, ε, του Καναδά και της Ρωσίας. Στη Σουηδία υπήρξαν πρόσφατα πυρκαγιές δασικές. Αντιθέτως, εμείς στη Φιλανδία δεν είχαμε τέτοιου είδους ε, ε, είμαστε λοιπόν σε θέση να ε, φροντίσουμε τα δάση μας και να αναπτυχθούν. Ωστόσο τώρα ανησυχούμε πάρα πολύ για τα ευρωπαϊκά δάση. Όμως ελάτε στη Φιλανδία και δείτε, δείτε πώς φροντίζουμε τα δάση μας εμείς. Εγώ προσωπικά έχω εμπειρία σε αυτό το τομέα και όταν ήμουν 16 χρονών ξεκίνησα να εργάζομαι στα δάση. Και είδα με ποιον τρόπο τα φροντίζουμε, τα διαχειριζόμαστε τα καλλιεργούμε και τα αξιοποιούμε. Και γνωρίζω δηλαδή με ποιον τρόπο καταφέρνουμε να διατηρήσουμε εκεί την ε, βιοπικιλότητα. Οπότε σας προσκαλώ πραγματικά να έρθετε στη χώρα μου στη Φιλανδία και να δείτε πώς τα καταφέρνουμε εκεί. Μην προσπαθείτε λοιπόν να μας δώσετε συμβουλές ε, και να ορίσετε κανονισμούς ε, ως προς το τι θα πρέπει να κάνουμε, γιατί εσείς αντιμετωπίζετε προβλήματα, όχι εμείς στη Φιλανδία. Ευχαριστώ. Υπάρχει μπλε κάρτα. Υπάρχει μια μπλε κάρτα από τον κύριο Ρόλαντ. Αυτή είναι η σύνθεση διαδικασία. Περιμένετε λίγο. Κύριε, δέχεστε την μπλε κάρτα. Δέχεστε να σας υποβληθεί μια ερώτηση. Ναι. Ο κύριος Ρόλαντ τώρα μπορεί να υποβάλει την ερώτησή του. The, the question I had was... ναι, ήθελα να θέσω ένα ερώτημα ε, σε σχέση με αυτό που υπόθηκε. Ε, γιατί υπάρχει μια αντίφαση ε, ανάμεσα σε αυτά που θέλουμε εδώ να υποστηρίξουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα δάση, αφενός και από την άλλη με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το βιοντίζελ και τη βιομάζα. Δηλαδή θέλουμε και υποστηρίζουμε για παράδειγμα μια πολιτική η οποία καταστρέφει ε, τα τροπικά δάση, για παράδειγμα της Ινδονησίας ε, και αλλού ή καταστρέφει και τον βιότοπο ε, ζώων όπως ο ουρακοτάκη και ούτω καθεξής. Πρόεδρος, ε, αυτό που είπατε μόλις τώρα δεν ακούγεται ως ερώτημα αλλά ως παρέμβαση. Έχετε μόνο 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας κύριε Ρόλαντ για να θέσετε το ερώτημά σας. Μπορείτε να απαντήσετε αν θέλετε You are going to stand up and answer the question. I didn't. wasn't clear. Ε, ε, θα απαντήσετε στο ερώτημα. Θα πρέπει να σηκωθείτε και να απαντήσετε αν το επιθυμείτε. Πρόεδρε, μπορώ να απαντήσω μόνο σε ερωτήματα. Καλώ λέει πρόεδρο. Κύριε Ρόλαντ, λάβατε την απάντησή σα. Οπότε, επόμενο ομιλητή, η κυρία Βυσνεύσκα, για 1,5 λεπτό εκ μέρους του ECR. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, εξότιμη κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, πραγματικά η προστασία των δασών μας θα πρέπει να αποτελέσει μία από τις κύριες προτεραιότητες μας μέσα στην επόμενη δεκαετία. Κατά τελευταία χρόνια έχουμε βιώσει μαζικές καταστροφές των δασών μας λόγω για παράδειγμα παρασίτων όπως όπως ο βλαστοφάγος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλα αυτά τα πάει σχετικά ε, καλά ε, σε σύγκριση με κάποιες άλλες ε, περιοχές. Και στην Πολωνία, για παράδειγμα, η δασικές εξάσεις αυξάνονται σταθερά. Δηλαδή από 20% που καταλάβαιναν γύρω στο 1940 τη σήμερα ημέρα καταλαμβάνουν το 30% της συνολικής μας έκτασης ε, και η δική μας Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης των Δασών αποτελεί πραγματικά ένα φορέα με καλές πρακτικές οι οποίες θα έπρεπε να διαδοθούν και αλλού. Με αναδασώσεις ε, ενός εκατομμυρίου δέντρων κάθε χρόνο. Ε, βλέπουμε δηλαδή να λαμβάνει η χώρα ευρύτατη αναδάσωση, αλλά δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας υποστηρίζει σε αυτές τις ε, πρωτοβουλίε. Μια ενεργός λοιπόν δασοκομική πολιτική είναι εξαιρετική σημασία. Ε, και αφού έχουμε κάποιες βέντισες πρακτικές να μοιραστούμε με τους υπολείπου, καλό θα ήταν να αξιοποιηθούν. Ευχαριστώ. Καλώ προτού δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή να κάνω μια διευκρίνηση για τα νέα μέλη. Εδώ, όταν λέμε μπλε κάρτα, πρόκειται για ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να θέσει κάποιο στον ομιλητή που μόλι πήρε το λόγο για 30 δευτερόλεπτα. Ο κύριος Φερέρα ε, έχει τώρα το λόγο εκ μέρου τη Γκουέντζιελ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο ευάλωτο ε, χαρακτήρα ε, των ε, δασών διεφάνει και στο πλαίσιο των πυρκαγιών που διαπιστώσαμε, αλλά και με βάση τι εξωτικέ ασθένειε και του διάφορου επιβλομή οργανισμού. Και βλέπουμε ότι σε αυτό ο ευάλωτο χαρακτήρα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει, υπάρχουν ελλειπεί επενδύσει και δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό δυναμικό. Και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ασκηθεί κατάλληλε πολιτικέ και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιωτικό και αποδόμηση των δημοσίων υπηρεσιών, πράγμα που σημαίνει υποβάθμιση και της ε, δασική, των δασικών ε, περιοχών. Και αυτό και, για παράδειγμα και στη Μαδέρα, οι οποίοι ουσιαστικά δεν κατάφεραν να επιβιώσουν οικονομικά και αυτό οδήγησε με τη σειρά του βέβαια στην εγκατάλειψη των υπαίθριων περιοχών και στην εγκατάλειψη ευρύτερων περιοχών. Εδώ και πολύ καιρό λοιπόν υποστηρίζουμε την αύξηση των επενδύσεων στον δασικό τομέα και ε, υποστηρίζουμε την, μια ευρωπαϊκή προσέγγιση σε ό,τι αφορά τέτοιου είδου καταστροφέ με την απαραίτητη πυρκοδόπηση από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και προκειμένου να εφαρμόζονται στην πράξη αυτέ οι πολιτικέ. Δηλαδή, πέραν ε, τη ε, δασική πολιτική υπάρχουν και άλλε πολιτικέ αγροτικού χαρακτήρα σε ό,τι αφορά δηλαδή το, την υπαίθρια ανάπτυξη οι οποίε και αυτέ μπορούν να υποστηριχτούν μέσω δημοσίου κοντιλίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Παπαδάκη τώρα για ένα λεπτό. Η Ελλάδα έζησε πέρσι μεγάλη τραγωδία στο Μάτι με 102 νεκρούς και φέτος όπως κάθε χρόνο βίωσε μεγάλες πυρκαγιές σε Εύβοια, Ανατολική Αττική, Ζάκυνθο, Λουτράκη και αλλού οι κυβερνήσεις αλλάζουν αλλά ο ευρωνοσιακός σχεδιασμός μένει αυτός της εμπορευματοποίησης της γης της επιχειρηματικής δράσης στα δάση της εγκληματικής γύμνιας του κρατικού μηχανισμού με ένα ένα δις περικοπές την τελευταία δεκαετία στη δασοπυρόσβευση και δασοπροστασία. με το λεγόμενο resceu οι ελλείψεις σε μέσα προσωπικό υποδομές χρηματοδότηση σε κάθε κράτος μέλος όχι μόνο δεν καλύπτονται αντίθετα νομιμοποιούνται και διαιωνίζονται αυτό στηρίζεται στη δέσμευση μέρους των επιχειρησιακών ικανοτήτων του κράτους μέλους με τυράκι περιορισμένες χρηματοδοτήσεις για αγορές και επιδιορθώσεις αεροσκαφών οι οποίες θεωρούνται από την ευρωπαϊκή ένωση συνολικά κόστος ο μηχανισμός στέλνει δυνάμεις όπως ήδη αποδεικνύεται κατόπιν εορτής αν αυτές δεν απασχολούνται αλλού και μόνο σε εξαιρετικά κρίσιμες καταστάσεις. απαιτούμε εδώ και τώρα επαρκή κρατική χρηματοδότηση με μόνιμο προσωπικό με πλήρη δικαιώματα άρτιο εξοπλισμό σε κάθε χώρα για την κάλυψη όλων των πραγματικών αναγκών και καμιά επιχειρηματική δράση στα δάση. Ξέρετε κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, είναι έτσι όπως τα είπατε ε, κύριε Επίτροπε, δηλαδή η κατάσταση των δασών ε, πραγματικά είναι απειλητική τουλάχιστον εν μέρη. Ε, ο βλαστοφάγος δηλαδή ασχολείται, εξαπλώνεται όλο ένα και περισσότερο λόγω και της κλιματικής αλλαγής, αυξάνονται ταυτόχρονα και οι και τα καιρικά φαινόμενα και στη δική μου περιοχή το τελευταίο φθινόπωρο. Από την άλλη πλευρά όμως φυσικά και τα δάση μας και η ποικιλότητα παίζουν σημαντικό ρόλο. Ε, τα δάση μα δηλαδή αποτελούν τον, το πράσινο πνεύμονά μας ε, και για να τα προστατεύσουμε χρειαζόμαστε πράγματι μια βιώσιμη δασική πολιτική η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική. Ε, μπορούν να παίξουν το ρόλο που θέλουμε τα δάση σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή, μόνο εφόσον αξιοποιήσουμε με τέτοιο τρόπο τα δάση και την ξυλία που παράγουμε, έτσι ώστε να παράγουμε με τον κατάλληλο τρόπο τα προϊόντα μα αλλά και την ενέργειά μα. Ακούσαμε να λέγονται πολλά σε ό,τι αφορά την βιώσιμη δασική πολιτική, τη βιωσιμότητά τη και πράγματι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να διατηρήσουμε ζωντανά τα δάση μα αλλά και βιώσιμα ε, ε, με βάθο χρόνου δηλαδή έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, τα αξιοποιήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο και στον τρόπο τη αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Νομίζω πω μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό και μέσω του δεύτερου πυλώνα τη κοινή γεωρική πολιτική και σε σχέση με αυτό με ανησυχούν πάρα πολύ οι περικοπέ που έχουν προβλεφθεί στον προπολογισμό του δεύτερου πυλώνα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να λογιστούμε αν στο πλαίσιο τη συζήτηση που κάνουμε για την κλιματική αλλαγή κατά πόσο θα πρέπει να θεσπίσουμε νέα εργαλεία τα οποία θα επιτρέψουν να διατηρήσουμε ζωντανά τα δάση μας ε, προκειμένου να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Δύο λεπτά ο κύριος Δεκάστο. Επίτροπε, συνάδελφοι, πρόεδρε, η κατάσταση των δασών είναι και χειρότερη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει τον ηγετικό της ρόλο στον αγώνα αυτό. Έχουν ε, γίνει πολλά πράγματα. Πρέπει να τα επενθυμίσουμε και χάρη στην ευρωπαϊκή κοινή γεωργική πολιτική. Τα τελευταία 20 χρόνια αυξήθηκε η δασική επιφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ισούται ε, με την έκταση τη Πορτογαλία. Αυτό είναι το σήμα κατεθέν μια ευρωπαϊκή στρατηγική που πρέπει να βελτιωθεί βέβαια, αλλά που έφερε ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, αγαπητέ Επίτροπε, δεν μπορούμε να σταματήσουμε εδώ οι περικοπές που προβλέπονται στην ΚΑΠ, στην κοινή γεωργική πολιτική, με την πρόταση της Κομισιόν, σημαίνουν σε ορισμένε χώρες ότι θα υπάρξει δραστική μείωση των προγραμμάτων ανάπτυξη πέθρου. Σε αυτές τις ε, χώρες θα έχουμε 25% μείωση. Και αυτό αποτελεί βέβαια ένα βήμα προς τα πίσω που είναι παράδεκτο. Οι γεωργοί μα, οι δασοκόμοι μα θα πρέπει να είναι πρωταγωνιστές σε αυτόν τον αγώνα και να μπορέσουν να βοηθήσουν για να διορθωθούν τα προβλήματα στα δάση. Επίσης, παράλληλα, θα πρέπει να ε, δράσουμε σε επίπεδο μεγάλων ε, χωρών που εξάγουν ε, ξυλία με συγκεκριμένα προγράμματα, ούτως ώστε να ενεργοποιηθούν ρήτρε διασφάλισης. Βρισκόμαστε ενώπιον μια πραγματική κλιματική απειλή. Και μόνο μια δυνατή Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο μια ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει τις θαραλέες απαντήσεις που θέλουν οι πολίτες και δεν θα παραπέμπει το θέμα στις καλένδες ακόμα μια φορά. Ένα λεπτό, κύριο Στεφανούτα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, στη Ρουμανία Υπάρχουν πολλά δάση τα οποία πρέπει να προστατευθούν λόγω του σημαντικού τους ρόλου στη βιοπικιλότητα. Παρόλα αυτά βλέπουμε καταστροφή τους ε, και παραβίαση της οδηγίας ε, περί ε, βιοτόπων. Μέσα στα επόμενα έξι χρόνια υπολογίζεται ότι 3,6000 εκτάρια ε, θα καταστραφούν. 1,3 εκατομμύρια ε, κυβικά μέτρα ε, ξυλίας έχουν εξαχθεί. Και ο οργανισμός Earth and Green έχει υποβάλει αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσει η υλοτόμηση. Κύριε Επίτροπε, αυτά που βλέπουμε στα έγγραφα δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Θα πρέπει να εφαρμοστούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα στις διάφορες χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Η κυρία Ντεπαρνέ Γκρίνεμπεργκ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι το δάσος αναπτύσσεται πολύ αργά. Έτσι είναι η φυσική ρυθμή και βέβαια πρέπει στην Ευρώπη να ε, αναπτύξουμε περαιτέρω την, ε, ε, την δασοκομεία, θα πρέπει να κάνουμε πιο ανθεκτικά στα δάση μας, θα πρέπει να υπάρχει χώρος για τη φύση. Επίσης, θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε βιώσιμη παραγωγή του πολύτιμου αυτού υλικού του ξύλου. Ωστόσο, η το δάσος είναι ο μόνος τρόπος να αντισταθμιστούν κάποιες αρνητικές συνέπειες της ε, κοινωνίας μας ε, που βασίζεται στην όλο και μεγαλύτερη παραγωγή δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τα δάση μόνο κατά βόθρα διοξιδίου του άνθρακα, ούτε μπορούμε ε, να αλλάξουμε ε, την βιοπικιλότητα με άλλα μέτρα. Είναι λάθος η πολιτική αυτή και δεν μπορούμε να τα πετύχουμε όλα αυτά γρήγορα και ταυτόχρονα. Τα δάση αναπτύσσονται πολύ αργά. Τα παιδιά μας θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα που θα έχουμε πετύχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, κυρία Λίμε. Danke. In den Mitteilungen der Kommission στην, στις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπω τίτλους όπως είναι «Αποκατάσταση των δασών, μέτρα για την προστασία των δασών». Ε, μα δεν φοβάστε ότι γελιοποιείστε αυτή ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, με την ενεργειακή της μεταρρύθμιση συμβάλλει ε, στην καταστροφή των δασών. Και εάν δούμε τι γίνεται ε, στην Γερμανία που έχει πάνω από 33.000 αναμογεννήτριες, ε, πολλές βρίσκονται σε ε, βουνά με δάση. Δεν είναι... δεν είναι ο, ο σκολίτης, ο βλαστοφάγος, ο μεγαλύτερος καταστροφέας. Είναι ακριβώς η ενεργειακή μας μεταρρύθμιση και έχουμε γερμανικά δάση με δέντρα ηλικίας 800 ετών τα οποία καταστρέφονται. Ε, αφήστε στους ε, επιτόπου εμπειρογνώμονες ε, να καθορίσουν την πολιτική των δασών και όχι σε γραφειοκράτες από τις Βρυξέλλες. Ε, κυρία Λίμπερ, δέχεστε μία μπλε κάρτα από την κυρία Γραπίνη. Κυρία Γκραπίνη, παρακαλώ. 30 δευτερόλεπτα έχετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή αυτά που είπατε. Είπατε στην αρχή ότι είναι γελίο να μιλάμε για τα ευρωπαϊκά δάση. Όχι, νομίζω ότι είναι επίγον και σημαντικό εάν θέλουμε εσωτερική αγορά και ένωση κρατών που έχουν κοινού στόχου, θα πρέπει ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, δεν θα πρέπει από κοινού να αναλύσουμε την κατάσταση και να λάβουμε μέτρα για την προστασία των δασών. Νομίζω ότι δεν καταλάβατε τις παρατηρήσεις μας. Γελίο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ενεργειακή της μεταρρύθμιση ε, ε, που συμβάλλει στην καταστροφή να λέει ακριβώς ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα δάση. Mr. is our next for... Ο κύριος Τζαμπάσκι είναι ο επόμενος ομιλητής. Ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι πολύ επίκαιρη η συζήτηση αυτή. ιδιαίτερα μετά τις ε, τρομερές πυρκαγιές σε όλον τον κόσμο που κατέστρεψαν μεγάλες εκτάσεις. Ελπίζουμε ότι τα πράγματα δεν θα παραμείνουν στο επίπεδο της συζήτησης μόνο, όπως δυστυχώς συμβαίνει συχνά. Παρότι η δασοκομεία αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή στρατηγική ως σημείο αναφοράς. Η Ευρώπη ε, αντιπροσωπεύει το 5% των ε, δασών όλου του κόσμου. Τα ευρωπαϊκά δάση μπορεί σε παγκόσμιο επίπεδο να μην είναι πολύ σημαντικά, ωστόσο είναι αλήθεια ότι τα δάση είναι οι πνεύμονές μας. Είναι αλήθεια ότι όλοι συμφωνούμε όσον αφορά τη σημασία των δασών για την προστασία της βιοπικιλότητας και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ κύριο Σκάρθη, ένα λεπτό. Um, um, Κύριε Επίτροπε, η στρατηγική για τα δάση κανονικά θα πρέπει να είναι καλή για το περιβάλλον, καλή για τις τοπικές κοινότητες και καλή για την ε, οικονομία των αγροτικών περιοχών. Στην Ιρλανδία, στη δική μου χώρα, η κυβερνητική πολιτική έχει φροντίσει η πολιτική για τα δάση να μην κάνει τίποτα από όλα αυτά. Και γι' αυτό βέβαια δεν φταίνε ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θα ήθελα όμως από εσά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δέσμευση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα χρηματοδοτήσει αυτή την πολιτική και στρατηγική ε, με την οποία ε, έχουν ε, φυτευτεί δάση με ήδη μη αυτόχθονα ε, σε ε, τυρφώνες όπου πιο πολύ ζημιά κάνουν παρά όφελος προσφέρουν. Και επίσης θα ήθελα να μας πείτε, γιατί από τη μία μιλάτε για πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, για τα δάση, ενώ από την άλλη αφήνετε τη Βραζιλία να καίει χιλιάδες ε, εκτάρια ε, δασών που είναι πάρα πολύ σημαντικά για όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Ε, ε κύριε Κάρθη, αύριο έχουμε συζήτηση για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. μισή λεπτό η κυρία Πόλφιαρτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όλοι συμφωνούμε ότι παίζει τα δάση ρόλο κλειδί ε, στην αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Η κατάσταση των ευρωπαϊκών δασών είναι κακή ε, και λόγω της ξηρασίας. Θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας το θέμα αυτό και θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε στη συνέχεια. Η λύση όμως δεν είναι ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να διατηρήσουν την ε, αρμοδιότητα για τα δάση θα πρέπει να δει κάθε χώρα πώ θα συνεχίσει να διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δάση. Δύο πράγματα όμω μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρώτον, να εξυγχρονίσουμε και να επικαιροποιήσουμε τη στρατηγική για τα δάση του 2013. Διότι έχουν υπάρξει μεγάλε αλλαγέ στον κόσμο έκτοτε. Και επίση να φροντίσουμε η ευρωπαϊκή νομοθεσία να λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες που προσφέρουν τα δάση και τα προϊόντα των δασών. Ευχαριστώ. Thank you, Madam. Ευχαριστώ. Σπούρεκ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα δάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούνται από τα πιο πολύτιμα ε, φυσικά, φυσικές περιοχές, π.χ. τα Καρπάθια Όρη. Αυτό που συμβαίνει όμως τώρα ε, θέτει πολλά ερωτήματα. Το Πολωνικό Υπουργείο ε, Περιβάλλοντος αποφάσισε να κάνει μαζική ξύλευση δασών. Η πρωτοβουλία Άσπρα Καρπάθια, www. καλύπτει περιοχές του Natura 2000 και παραβιάζει αυτή η νέα απόφαση της, του Υπουργείου ε, διάφορες οδηγίες, ε, την οδηγία ενδιατεμάτων, οικοσυστημάτων κτλ. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να επιληφθούν του προβλήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μιούλερ, για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είχαμε ακραία ξηρασία τα τελευταία χρόνια, κάτι που έχει ε, βλάψει τα δάση μας και έτσι μπόρεσε να ε, επεκταθεί ε, με κρίτικους ρυθμούς ε, ο σκολίτης τα τελευταία 20 χρόνια. Έχουμε καταστρέψει δάση που είχαν καταστραφεί από τον σκολίτη και αυτό ήταν τεράστια οικονομική καταστροφή. Το δάσο, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, χάνει, είναι ο χαμένος από την αλλαγή του κλίματος. Για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στο μέλλον χρειαζόμαστε βιώσιμη διαχείριση των δασών ε, και χρειαζόμαστε ε, αηφόρο στρατηγική για τα καύσιμα, για την χρήση της ξυλίας σε όλους τους τομείς ε, της ζωής τα ε, η ξυλία που είχε καταστροφεί από ε, τον σκολίτη θα μπορούσε να προσφερθεί για ε, δημόσια κτίρια. Τα δάση αποθηκεύουν διοξείδιο του άνθρακα και προστατεύουν το κλίμα. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι μας. Κυρία Ριβαζή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τα δάση μας κινδυνεύουν και οι πυρκαγιές φέτος το καλοκαίρι μας αφυπνίζουν. Χάσαμε το ισοδύναμο 800 ε, γηπέδων ε, ποδοσφαίρου την ώρα με αυτές τις ε, πυρκαγιές. Η ανακοίνωσή σας κάνει πολύ σωστές διαπιστώσεις, κύριε Επίτροπε, αλλά δεν είναι πολύ αποφασιστική σε ό,τι αφορά τις προτάσεις. Προτείνει διάλογο και θελοντισμό, αλλά πολύ λίγα δεσμευτικά μέτρα. Να σας υποβάλω εγώ μερικές προτάσεις. Καταρχάς, για το θέμα ξύλο και ενέργεια. Θα πρέπει τώρα και όχι το 2023 να αποκλείσουμε αυτό το, το, ξύλο και το δάσος να χρησιμοποιείται για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, η, επίσης η έντονη γεωργία ε, οδηγεί σε αποδάσωση. Ε, επίσης ε, η καλλιέργεια του φινικέλεου ε, αποψηλώνει τα δάση της Αμαζονία. Θα πρέπει να δώσουμε τα, τη δυνατότητα στου αυτόχθονε πληθυσμού. την δυνατότητα να προστατεύσουν τα δάση τους, γιατί αυτοί είναι οι καλύτεροι θεματοφύλακες. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να γίνουμε, κύριε, ε, να, που να, μπορούν να γίνουν, κύριε Επίτροπε, και περιμένουμε και συγκεκριμένες προτάσεις. Πλάσκο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι δάση στην κεντρική Ευρώπη πεθαίνουν λόγω ενός συνδυασμού διαφόρων παραγόντων. Καταρχάς, ότι μας, ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρουν ε, υπερβολικά τα δάση ε, και οδήγησαν σε μια φοβερή ανάπτυξη του σκολίτη. Ε, δημιουργούμε αυτές τις ε, ζώνες μη παρέμβασης, ας πούμε, στα εθνικά δάση και ο σκολίτης είχε θαυμάσιο πεδίο για να πολλαπλασιαστεί. Γιατί δεν μπορούμε να να κόψουμε δέντρα σε αυτές τις ζώνες, ούτε καν τα, τα άρρωστα ζώνα. Κάποτε τα δάση μας ήταν υπέροχα και τώρα είναι κατεστραμμένα. Είναι ένα αξιολύπητο θέαμα αυτά τα άρρωστα δάση. Προτείνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει κατεπήγοντα μέτρα εναντίον της ανθρώπινης βλακείας και της ε, βλακείας των εμπειρογνωμόνων. Και καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσει αυτές τις, ε, ε, την, ε, τις πράσινες ζώνες, ζώνες ε, ανάσχεσης, όπου απαγορεύεται η, το να κόβουμε δέντρα. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Υπάρχει ε, ένα ερώτημα την κυρία Σόντεβα. Κυρία Μπλάσκο, το δέχεστε. Ναι, παρακαλώ. Ακούμε την ερώτηση. Θα ήθελα... Δεν θα ήθελα να κάνω μια τσέχο-τσεχική συζήτηση. Όμως, ο κύριος Μπλάσκο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει για να λύσει προβλήματα των κρατών μελών. Πιστεύετε ότι το Τσεχικό Υπουργείο Δασών ή ότι οι αρχές μας δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις. Θεωρείτε ότι κάποιος θα πρέπει να τους υποδείξει τι να κάνουν. Εγώ εμπιστεύομαι τους διαχειριστές των δασών, εμπιστεύομαι τους εμπειρογνώμονες, εμπιστεύομαι τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό το θέμα στη χώρα μου. Uh, Συνάδελφε, αντίθετα από εσά, εγώ συμμετείχα σε προσπάθειες ε, ξερίζωσης του σκολίτη και βλέπω τι γίνεται με τα δάση σε διάφορα βουνά μας. Έχετε πάει ποτέ σε αυτά τα υπέροχα κάποτε δάση, σε τι κατάσταση βρίσκονται σήμερα. Επειδή δεν ξέρουμε από μόνοι μας, χρειαζόμαστε εξωτερικές συμβουλές. Υπάρχουν τόσο πολλοί πυρογνώμονες επιτόπου Κοιτάξτε ποια είναι η κατάσταση στη Σούμοβα. Κοιτάξτε το αποτέλεσμα των εργασιών στην περιοχή αυτή. Τόματσιτς, ένα λεπτό. Τα δάση μας είναι ε, πάρα πολύ σημαντικά για το περιβάλλον, τη γεωργία μας, την ποιότητα του εδάφους, ε, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και την ενεργειακή μας αυτονομία. Αποτελούν ένα πολύ σημαντικό πόρο και Ευτυχώ εμεί στην Ευρώπη δεν πληττόμαστε από ε, παράνομη υλοτομία σε τεράστιο βαθμό. Και παρότι υπάρχει αύξηση των εκτάσεων, δεν σημαίνει ότι έχουμε διαχειριστεί σωστά τα δάση μα. Οι διαφορέ δηλαδή ανάμεσα στα εκάστοτε κράτη-μέλη είναι τεράστιε. Και εδώ δεν αναφέρομαι μόνο στην έκταση που καταλαμβάνουν τα δάση, αλλά και στην κυριότητα αυτών. Γιατί τα περισσότερα δάση βρίσκονται σε ιδιωτικά χέρια. Για παράδειγμα, στο, στην Κροατία το 80% των εδασών είναι δημόσιας ε, κυριότητα ε, και τη χάνουν διαχείριση από μια δημόσια υπηρεσία. Στο μέλλον θα πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε κοινού στόχου, Έχοντα όμω ταυτόχρονα υπόψη ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μα τι ιδιαιτερότητε του κάθε κράτου μέλου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Γεωργούλη τώρα για ένα λεπτό δεν είναι λογικό η ευρωπαϊκή ένωση να μην διαθέτει κοινή δασική πολιτική. τα δάση εκτό από φυσικό πλούτο μια χώρα είναι και ο πνεύμονα όλου του πλανήτη. δημιουργούν οξυγόνο για όλου του ανθρώπου αλλά και για τα ζώα. υπολογίζεται ότι το 43% τη έκταση τη ευρώπη αποτελείται από δάση τα οποία εκτό από τον πλούτο των οικοσυστημάτων και τη χρήσιμη πηγή ανανεώσιμη ενέργεια που προσφέρουν έχουν και την ικανότητα να απορροφούν εκπομπέ του διοξιδίου του άνθρακα. τα ευρωπαϊκά δάση απορροφούν το 10% των εκπομπών αυτών η ραγδαία υπερθέρμανση όμω οδηγεί σε φωνικέ πυρκαγιέ. Φέτο. ο μέσο όρο των πυρκαγιών στην ευρωπαϊκή ένωση τριπλασιάστηκε. ο Ευρωπαϊκό Νότο, η ελλάδα η ιταλία η ισπανία η πορτογαλία φλέγονται κυριολεκτικά κάθε καλοκαίρι από με σημαντικέ απώλειε σε φυσικό πλούτο ζώα αλλά και ανθρώπου. προβλέπεται επίση ότι αυτό ο, αριθμό θα αυξηθεί κατά 40 με 100% τα τελευταία χρόνια. δηλαδή δεν έχουμε δεν θα έχουμε δάση να προστατεύσουμε σε λίγο καιρό. γι' αυτό πρέπει να δράσουμε άμεσα και να... όσο έχουμε την πολυτέλεια. γιατί να μην ε, πάρουμε σαν παράδειγμα το μεγάλο πράσινο τείχος στην αφρική και να το ακολουθήσουμε. μεγαλώσαμε με το φόβο ότι η κλιματική αλλαγή θα είναι ένα πρόβλημα που θα απασχολούσε κάποια από τις επόμενες γενιές και τελικά η γενιά αυτή είμαστε εμείς. ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Άλβαρε Ζόιντε τώρα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε. Και καλή τύχη ενώπιον της Επιτροπής ε, κλίματο ε, και Περιβάλλοντος. Ελπίζω να τελεσφορήσει το, η συμφωνία του Παρισιού και να υλοποιηθούν οι φιλόδοξοι στόχοι ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. Είναι ένα μεγάλο θέμα, μεγάλος ε, σύμμαχος στα δάση που φιλτράνε τον αέρα, μας βοηθούν να καταπολεμήσουν ε, την κλιματική αλλαγή και παίζουν σημαντικό ρόλο, ειδικά στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Ε, το ξέρουμε πολύ καλά στην Ισπανία. Ε, είναι η δεύτερη χώρα σε, μεγαλύτερη, ε, σε έκταση δασική στην Ευρώπη. Και είναι Έχουμε 750 εκατομμύρια δάση ε, που απορροφούν 35% του διοξείδου του άνθρακα που εκπέμπουμε. Ε, και δεν υπάρχει τοπίο χωρίς δασικό τοπίο. Όμως για να διασώσουμε τα δάση μας αυτό εξαρτάται από τη σχέση που έχουν τα δάση με τι γεωργικέ κοινότητες και του γεωργικού πληθυσμούς. Τα δάση είναι ουσιαστικά για να καταπολεμήσουμε την αποψήλωση τη υπαίθρου. Ε, γεννούν οικονομικές ευκαιρίες ε, στα χωριά και στην αγροτική Ισπανία. Ε, παίζουν μεγάλο ρόλο στην βιοπικιλότητα, στη βιοενέργεια. Γι' αυτό ε, απορρίπτουμε τις περικοπές που προτείνει η Κομισιόν για τον προπολογισμό της ΚΑΠ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος ε, Γκονσάλες Καζάρες. Για ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ όπως υπόθηκε. Από τη μία πληρώνουμε για αγιορικά προϊόντα τα οποία μειώνουν τα δάση σε τρίτες χώρες και από την άλλη σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης ε, Έχουμε εγκατάλειψη των παραδοσιακών καλλιεργειών, έχουμε εκτεταμένη κτηνοτροφία και αυξάνονται βεβαίως οι δασικές πυρκαγιές. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την προοδευτική εξαφάνιση των δασών μας. Ειδικά ε, αυτά που είναι κοντά στη θάλασσα, στον Ατλαντικό και που είναι... Ε, απορροφούν το ε, διοξείδιο του άνθρακα. Στην Καλύφθη, ας πούμε, διπλασιάσαμε τις δασικές περιοχές. Απλώς δεν θέλουμε να τη χάνουν άτακτη διαχείριση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προχωρήσουμε με πολιτικέ ε, που, που φρενάρουν την αποψήλωση και να στηρίξουμε και διεθνεί εμπορικέ πολιτικέ τέτοιου τύπου. Εδώ στην Ευρώπη θα πρέπει να έχουμε μια βιώσιμη δασική διαχείριση, να προστατεύσουμε τα παραδοσιακά δάση, να καταπολεμήσουμε την αποψήλωση της υπαίθρου και να καταπολεμήσουμε την εντατική κτηνοτροφία με κονδύλια της ΚΑΠ για να κρατήσουμε τα δάση μας και τα οικοσυστήματα με το, στον πλέον υγιή, ε, στην πλέον υγιή κατάσταση. Ευχαριστώ. Ε, επόμενος, ο ο κύριος Χόισικ Μάρτιν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Ξιότιμε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. τα ευρωπαϊκά δάση απειλούνται και απειλούνται όχι μόνο στο πλαίσιο της κρίσης της κλιματικής αλλαγής αλλά και από την αύξηση της υποδομής ε, των ανθρώπων και από τα χημικά προϊόντα. Ε, και οι συνέπειες είναι καταστροφικές για το σύνολο της ε, κοινωνίας, για την κοινωνία μας. Αν θέλουμε λοιπόν μια εκπληρώσουμε τους στόχους μας και να διατηρήσουμε τη βιοποικιλότητά μας, τότε θα πρέπει να προστατεύσουμε τα δάση μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν κανόνες οι οποίοι θα επιτρέψουν ε, ή θα απαγορεύσουν μάλιστα τον ψεκασμό των δασών, θα ε, επιτρέψουν ε, την διατήρησή τους και φυσικά θα πρέπει ένα ελάχιστο ποσοστό 5% των δασών να παραμένουν ανέπαφα, χωρίς καμία ε, παρέμβαση. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση πολιτικού χαρακτήρα ή οικονομικού χαρακτήρα συμφέροντα να υπερισχύσουν ε, τη προστασία των δασών. Τα δάση είναι απολύτω απαραίτητα για την βιοποικιλότητα και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή στρατηγική προκειμένου να καθορίσουμε ε, το μέλλον. Ευχαριστώ η κυρία Σάστια Μπρικμόν τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν ξέρουμε ότι τα δάση συμμετέχουν ε, στην υλοποίηση των 9 από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξη μεταξύ των οποίων ε, παραγωγή τροφίμων, ανεφοδιασμό σε καθαρό νερό, ε, δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα, βιοπικιλότητα κτλ. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να είναι πιο ψηλά τα δάση στην πολιτική ατζέντα μας και γι' αυτό χαίρομαι για την προσπάθεια που κάνει η κυρία Φοντερ Λάιεν για να προωθήσει αυτό το θέμα. Υπάρχει πολιτική αναδάσωση, αλλά θέλω να κρατήσω μία φράση από την ανακοίνωσή σα. Τα δάση, τα οποία φυτέψαμε πρόσφατα, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα αρχαίγωνα δάση. Ε, όταν υπάρχει καταστροφή δεν μπορεί να υπάρξει αναδημιουργία. Καμία απώλεια δεν μπορεί να ξεπεραστεί. 43% του ευρωπαϊκού ε, τη Ευρωπαϊκή Επικράτεια ε, είναι δάση. Θα πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα μέσα. Υπάρχουν στην ΚΑΠ, ε, υποχρησιμοποιούνται τα μέσα. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει να κάνει μια έτσι, εκστρατεία για να γνωστοποιήσει στα κράτη-μέλη τι υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό. Επίση, η βιομάζα είναι πολύ σημαντική. Ε, υπάρχει μια υποκρισία όμω. Χρησιμοποιούμε τη βιομάζα ω ε, ανανεώσιμη ενέργεια, γιατί παράγεται από τα δάση. Καταστρέφουμε τα δάση για, την, με, να φτιάξουμε βιομάζα. Μπίγνη Ευτόρα Κουσνόκ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ζήτησα το λόγο στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης έτσι ώστε να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η χώρα μου αποτελεί έναν από τους προτεργάτες ένα από τα καλύτερα παραδείγματα που έχουμε σε ό,τι αφορά την άσκηση της σωστής δασοκομικής πολιτικής. Έχουμε διπλασιάσει δηλαδή ε, τον αριθμό της ε, ξυλίας ε, που παράγουμε στην Πολωνία, αλλά ταυτόχρονα τα δάση καταλαμβάνουν πάνω από το 30% της συνολικής έκτασης της χώρας μας. κατά συνέπεια, χαιρετίζουμε την απόφαση που έλαβαν Συμβούλιο και Κοινοβούλιο του 2018 να περιληφθούν τα δάση στην περιβαλλοντική μας πολιτική. Η συμβολή ε, των δασών, στην μείωση των αποπών διοξιδίου του άνθρακα, προφανώς θα ε, ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό ε, της μείωσης αυτών των εκπομπών, αλλά υπάρχουν εξερασίες, υπάρχουν χειμώνες όπου δεν μειώνονται αρκετά οι θερμοκρασίε και άλλα τέτοια ακραία φαινόμενα, τα οποία δημιουργούν περισσότερους κινδύνους και κατά συνέπεια χρειαζόμαστε περισσότερη υποστήριξη για τη διαχείρισή τους. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Υπάρχει μια μπλε κάρτα Κυρία μέρτιο, δέχεστε την μπλε κάρτα, παρακαλώ. Έχει το λόγο συνάδελφος που θέλει να θέσει το ερώτημα. Ευχαριστώ κύριε Κούσμα ε, που μου να θέσω το ερώτημα αυτό. Έχω ζήσει λοιπόν στην Πολωνία και γνωρίζω τη σημασία που έχουν τα δάση για εσάς. Ε, θα ήθελα ε, να μας πείτε τι νομίζετε ότι κάνει η δική σας κυβέρνηση προκειμένου να προστατεύσει τα δάση εκεί. Κύριε Γκούσμακ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το ερώτημα. Έχουν υπάρξει πολλές παρανοήσεις σε ό,τι αφορά την άσκηση της πολιτικής της πολωνικής κυβέρνησης, σε ό,τι αφορά τα δάση ειδικότερα δε σε ό,τι αφορά το σκολίτι. Αυτό τον επιβλαβή ε, οργανισμό και την εξάπλωσή του στο δάσος της ε, Βιέζα ε, στα ανατολικά της χώρας μας. Όμως υπάρχουν κάποια παραδείγματα που μπορώ να σας αναφέρω και τα οποία καταδεικνύουν ότι πραγματικά μπορούμε να αποτελέσουμε υπόδειγμα ως χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να υπενθυμίσω ότι είναι ένας αυτοχρηματοδοτούμενος τομέας αυτός η δασοκομεία στη χώρα. Η κυρία Σάντερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, συνάδελφοι, τα δάση ήταν εδώ πριν από τη... τους λαούς εδώ, ενώ ε, η έρημος ήρθε μετά τον άνθρωπο. Αυτό έλεγε ο Σατομπριό. Ε, και η φετινή πραγματικότητα μας ε, υπέδειξε ότι εμείς ε, είμαστε η εξαίρεση στην Ευρώπη. Γιατί ε, κάθε τέσσερα δευτερόλεπτα καταστρέφονται ένα μεγάλο κομμάτι του δάσους. Είναι μεγάλη η ευθύνη. έχουμε καύσονες έχουμε επιθέσει από παράσιτα και αρρώστιε των ε, δέντρων. Πρέπει να διπλασιάσουμε τι προσπάθειε ούτω ή άλλω να διαχειριζόμαστε σωστά το ευρωπαϊκό δάσο και να παίζει ένα οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό ρόλο όπω πρέπει. Το δυναμικό των ευρωπαϊκών δασών ε, για την υλοποίηση των στόχων του Παρισιού, ε, τη συμφωνία του Παρισιού είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει βεβαίω να μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε του πόρου μα, αλλά με σεβασμό τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη ανάπτυξη του δασικού πλούτου μας και της δασικής κληρονομιάς. Φυσικά δεν υπάρχει καμία κοινή δασική πολιτική, αλλά οι ευρωπαϊκές πολιτικές μπορούν να επηρεάσουν τις εθνικές πολιτικές για τα δάση. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό, Πρόεδρε, τα... οι του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ να διατηρηθούν και στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Είναι σημαντικό να στηρίξουμε του ιδιοκτήτε δασών στον τρόπο που διαχειρίζονται τα δάση, για να του διαχειρίζονται με βιώσιμο τρόπο. Επίση, τα ερευνητικά προγράμματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουμε την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Η κυρία Αρένα, Μαρία Αρένα. Ευχαριστώ. Στην πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία των Δασών, η Κομισιόν προβλέπει μέτρα, επιπλέον μέτρα ρύθμιση για να καταπολεμήσουμε την αποδάσωση και να προστατεύσουμε καλύτερα τα δάση. Δύο ερωτήσει. Καταρχά, θα, κάνετε, θα εισαγάγετε δεσμευτική νομοθεσία ούτω ώστε τα επικίνδυνα προϊόντα για τα δάση, παραδείγματο χάρη τα προϊόντα τη εντατική γεωργία ή τα προϊόντα ε, από την εκμετάλλευση των ορυχείων, να μην οδηγούν σε αποδάσωση ε, και επιπλέον να μην πηγαίνουν στην, και όλα τα προϊόντα τα οποία μπαίνουν στην δική μας αγορά να μην οδηγούν σε αποδάσωση. Δεύτερο θέμα, ούτως ώστε να, να χρησιμοποιήσουμε ως μοχλό τις εμπορικές συμφωνίες. Σκοπεύετε το κεφάλαιο για την αηφόρο ανάπτυξη να το καταστήσετε ε, υποχρεωτικό με ακυρώσει, δηλαδή από αυτή την ε, κινέζικη εταιρεία ε, ε, Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι ο, ο χρυσός ο οποίος εκμεταλλεύεται, παράγει αυτή η εταιρεία με την εξόριξη αυτή και που μια εταιρεία που καταστρέφει πάρα πολλά δέντρα, δεν θα μπαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νόρπερ Τελίνης, ένα μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Το δάσος είναι τόπος όπου ζει κανείς, είναι προστάτης του περιβάλλοντος, προστάτης κατά της ε, αλλαγής του κλίματος. Ε, η ζέστη, η ξηρασία, ε, οι σκολίτες και άλλα τα καταστρέφουν. Δεν θα πρέπει όμως να αφήσουμε τη μόνη μας ελπίδα για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Ε, το 10% ε, των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα αντιπροσωπεύει η καταστροφή των δασών. Το, τα δάση όμως αποθηκεύουν το διοξίδιο του άνθρακα και είναι σημαντικό να έχουμε υγιή δέντρα ώστε να έχουμε και την μεγαλύτερη δυνατή αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. Τα δάση όμως είναι και ευάλωτα ε, απέναντι στην αλλαγή του κλίματος. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε μία ενεργό και αποτελεσματική ε, διαχείριση των δασών. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους αυτούς, ε, χρειαζόμαστε Χρειαζόμαστε υγιή δάση και γι' αυτό μια καλή στρατηγική. Και πολύ θα ήθελα να συμμετάσχω στην εκπόνηση ε, προτάσεων. Κύριε η κυρία Μίλλερ έχει μπλε κάρτα. Κυρία Μίλλερ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λίνς, συμφωνείτε ότι όσον αφορά τους σχολίτες, ε, χρειαζόμαστε έρευνες αλλά και προγράμματα που να χρηματοδοτούνται ε, με ευρωπαϊκούς πόρους, όπως είναι το πρόγραμμα LIFE ή το ε, Horizon 2020 διότι ε, είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε βιολογικά μέσα για την καταπολέμηση των σκολητών, που θα πρέπει όμως να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Κύριε Λίνς. Ναι, μπορώ να απαντήσω πολύ σύντομα. Πιστεύω ότι αυτό είναι καλή ιδέα και πολύ καλό θα είναι να στηρίξει η Ευρώπη μια τέτοια προσπάθεια. Ευχαριστώ σας, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έρο όμα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, για να κάνουμε κάτι καλό για τα δάση μας, θα πρέπει να είναι σαφές ότι έχουμε πολλά διαφορετικά δάση, όχι ένα ενιαίο. Το 70% της επιφάνειας της Φιλανδίας καλύπτεται από δάση. Η Φιλανδία πάντα εκμεταλλευόταν τα δάση της, χωρίς να μειωθεί όμως η συνολική έκταση των δασών της τα τελευταία 100 χρόνια. Είναι σημαντικά ε, και ως καταβόθρος διοξιδίου το άνθρακα ε, και είναι απαραίτητο η διαχείριση των δασών στην Ευρώπη να είναι βιώσιμη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν σκέφτεται τι θέλει να κάνει στο δάσος, δεν θα πρέπει να τιμωρήσει τις χώρες που ε, έχουν κάνει καλή διαχείριση των δασών. Η κυρία Σιμώνε Μπάουερ από την Αυστρία, από την Πράσινη Στηρία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ευγενική εισαγωγή σας. Είναι αυστριακή είμαι. Ε, το 50% των εκτάσεών μας ε, αποτελείται από δάση και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικά για μας. Ε, ωστόσο, ε, προτού συζητήσουμε την κατάσταση των δασών στην Ευρώπη, θα ήθελα να τονίσω γιατί έχουν τόσο μεγάλη σημασία τα δάση. Στον αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος δεν έχουμε καλύτερο υποστηριχτή από δάση με σωστή διαχείριση, διότι αποθηκεύουν διοξίδιο του άνθρακα, αλλά μας προσφέρει και προϊόντα. Πρέπει λοιπόν Λοιπόν να ε, στηρίξουμε, ε, να προστατεύσουμε τα δάση. Επίσης, ε, τα δάση αντιπροσωπεύουν πολλές θέσεις εργασίας, 3 εκατομμύρια. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Το κλίμα αλλάζει, βλέπουμε ακραία καιρικά φαινόμενα και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσει και, οι ε, και, να προστατεύσει τους ιδιοκτήτες των δασών και το, συνολικό, ε, και το σύνολο του δασικού τομέα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ισχυρή πολιτική για τα δάση και δεν επιτρέπουμε ε, καμία μείωση του δεύτερου πυλώνα ε, του γεωργικού προπολογισμού. Μα Χρειαζόμαστε δημόσιου πόρου για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες αλλαγή του κλίματο ε, στα κράτη-μέλη μα. Γι' αυτό ε, Πιστεύω ότι πολύ καλή λύση θα είναι η χρήση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υποστηρίξουμε τους ιδιοκτήτες δασών. Μπορείτε να είσαστε στο μέλλον ο βασικός μας εταίρος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Σμιτ Ο κύριος Γιάρουμπας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι, τα δάση αποτελούν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο των οικοσυστημάτων μας ε, στην Ευρώπη και η καλή τους κατάσταση αποτελεί προϋπόθεση για την απορρόφηση ε, διοξιδίου του άνθρακα και ταυτόχρονα αποτελούν βέβαια ένα σημαντικό τομέα ε, οικονομίας ε, που δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας, ειδικότερα δε, σε τοπικό επίπεδο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη και τους κατόχους των δασικών εκτάσεων και τους διαχειριστές τους προκειμένου να τα προστατεύσουμε καλύτερα και να αντιμετωπίσουμε ε, τις επιπτώσεις ε, μεταξύ άλλων των ε, δασικών πυρκαγιών. Θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας γιατί κατακαιρματισμένοι δεν θα είμαστε το ίδιο αποτελεσματικοί. Αυτό βέβαια ε, ε, δεν σημαίνει ότι το εθνικό επίπεδο δεν είναι ε, το καλύτερο επίπεδο για την ανάληψη δράσης. Θα πρέπει όμως να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια που παρέχονται μέσω της κοινή γεωργικής πολιτικής, μέσω της έρευνας και της τενοτομίας, αλλά και μέσω της συμπερίληψης της κοινή δασικής πολιτικής στο Horizon Europe η αναδάσωση των δασικών εκτάσεων θα πρέπει να αποτελέσει ε, πολιτική μας και ταυτόχρονα θα πρέπει να στοχεύσουμε στην αύξηση της ανθεκτικότητας ε, των δασών απέναντι σε επιβλαβείς οργανισμούς. Και ε, θα πρέπει να τα καταστήσουμε και πιο ανθεκτικά στις ξηρασίες. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Άλβαρο Αμάρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι διάφορες ε, συμφωνίες ε, δεν αναφέρονται ρητά ε, στην, στον όρο δάση και γνωρίζουμε πως τα θεσμικά όργανα κατά τελευταία χρόνια έχουν παρόλα αυτά να λάβει περισσότερη δράση σε αυτό το τομέα. Το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, το Συμβούλιο. Παρόλα αυτά, τη σήμερα ημέρα θεωρώ πως παρά μάλλον τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα διαφορετικά ε, κράτη-μέλη, ήταν δυνατόν να χαράξουμε μια κοινή γεωργική πολιτική παρά όλες τις διαφορές που υπάρχουν στους ε, γεωργικούς τομείς των διαφόρων κρατών μελών. Με την ίδια λογική λοιπόν θα πρέπει να είναι δυνατόν να χαράξουμε μια κοινή δασική πολιτική για τα διάφορα κράτη-μέλη. Και ακριβώς για να επιτύχουμε και την καλύτερη οικολογική ισορροπία θα πρέπει πάντοτε σεβόμενοι ε, τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής να διατηρήσουμε ναι ε, την απαραίτητη βιομάζα αλλά ταυτόχρονα να προστατεύσουμε και την οικονομική αξία των δασών. Η οικονομική αξία των δασών τι σημαίνει όμω με τη σειρά τη αν λάβουμε υπόψη μα και αυτέ τι ε, οπτικέ γωνίες, ε, σε περισσότερου ανθρώπους αυτού ε, του και περισσότερο, δηλαδή περισσότερη ανάπτυξη, ισορροπημένη ανάπτυξη. και γι' αυτό θα ήθελα να υποστηρίξω αυτό που υπόθηκε από τη συνάδελφο, ότι δηλαδή περισσότερη πρικοδότηση και το Ταμείο αλληλεγγύη. Γιατί οι δασικέ πυρκαγιέ δεν καταπολεμούνται, οι δασικέ πυρκαγιέ προλαμβάνονται. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ένα ταμείο το οποίο θα υποστηρίξει την πρόληψη τέτοιων πυρκαγιών στα δάση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ένα Βίρκουνεν. Πρόεδρε, χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε αυτή τη συζήτηση για τα ευρωπαϊκά δάση. 40% της ε, επικράτειάς μας καλύπτεται από δάση. Και τα δάση είναι πολύ σημαντικά. Ειδικά όταν καταπολεμούμε ή θέλουμε να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν δύο τρόποι και τα δάση είναι σημαντική δεξαμενή του άνθρακα και είναι και βιώσιμη πηγή ε, φυσικών πόρων. Οτιδήποτε γίνεται από πετρέλαιο σήμερα, στο μέλλον θα γίνεται από ε, δάση, από ξύλο. Ε, είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τα δάση και να κάνουμε μια ενεργή διαχείριση των δασών. Αυτά τα δάση τα οποία τα διαχειριζόμαστε με ενεργό τρόπο δεν είναι τόσο πολύ ευαίσθητα σε πυρκαγιές, ε, παράσιτα, ξηρασία κτλ. Όταν ε, επέλθει η κλιματική αλλαγή θα έχουμε πολύ πιο έντονες ε, κατακλυσμιές βροχές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε μία ευρωπαϊκή δάση δεδομένων για, για το δασικό μας πλούτο θα μας βοηθήσει να συζητήσουμε και την κατάσταση των δασών. Γιατί δεν έχουμε επικαιροποιημένη πληροφορία για αυτό το θέμα τώρα. Και περνάμε έτσι στην διαδικασία Catch the Eye. Ήδη ζήτησαν αρκετοί το λόγο. Έχω τα ονόματά τους. Όπως γνωρίζετε υπάρχει ο κανόνας ότι μπορούμε να έχουμε πέντε λεπτά Catch the Eye μπορούμε ενδεχομένως να προσθέσουμε ε, και κάνα δύο λεπτά. Οχτώ άνθρωποι έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Χίτρεκη Πάλας, παρακαλώ. Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, συναδελφίζουμε σε έναν κόσμο πολύ βιαστικό και η ταπεινοφροσύνη ε, είναι πολύ σημαντική. Ε, οι πληθυσμοί κοντά στους δασ... δάση είναι αυτοί που προστατεύουν τα δάση και τα δάση είναι θεματοφύλακα τη βιοπικιλότητα. Επίση, οι άνθρωποι αυτοί δεν σκέφτονται με χρονικό οριζόντα ένα ή δύο χρόνια, αλλά 20 με 30 χρόνια. Ε, στα, προ, ε, πλαίσια του προγράμματος αναδάσωσης ε, της Ουγγαρίας 20 εκατομμύρια δάση φυτεύθηκαν από τους δασοφύλακες. Είναι καταφύγιο, είναι τροφή για χιλιάδες φυτά και ζώα τα δάση αλλά και συνεισφέρουν επίσης στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν γύρω-γύρω καθώς και στο γεωργικό πληθυσμό και στη διατήρηση του κλίματος γενικά. Ξέρουμε ότι τα δάση δεν είναι μόνο οικονομικός παράγοντας και περιβαλλοντικός παράγοντας. Όχι, είναι γωνιές που ο, Θεός τα έδωσε, τους έδωσε σε εμά για να τις διαφυλάξουμε. Γι' αυτό η Ουγγρική κυβέρνηση αποφάσισε να διατηρήσει και να διαφυλάξει αυτά τα δάση. Ο πρόεδρος έκοψε το μικρόφωνο του ομιλητή. Η κυρία μου Μικρόφωνο παρακαλώ. Θα τα καταφέρω, ε, θα το βρω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να πάρω το λόγο για να τονίσω ότι η προστασία των δασών είναι αδύναμη ακόμη στην Ήπειρό μας, νομίζω. Παράδειγμα, το σύστημα προστασίας των παρθένων και ημιπαρθένων δασών. Παρότι αυτά τα δάση είναι ένα πολύ μικρό κλάσμα Τη ε, δασική έκτασης στην Ευρώπη είναι αξιοθαύμαστα σε ό,τι αφορά την οικολογική ε, αξία τους. Όμως ε, όλο και περισσότερα άγρια δάση τα εκμεταλλευόμαστε στη Σλοβακία και στη Ρουμανία. Περίπου 10 εκατομμύρια δέντρα το χρόνο κόβονται παράνομα σε όλη τη Ρουμανία. Θα ήθελα να βρω ένα κατάλογο ευρωπαϊκό κάποια στιγμή για τα αρχαίγον αυτά δάση και να αναγνωρίσουμε την αξία τους που είναι πολύ αυξημένη. Αυτός ο κατάλογος θα πρέπει να απαριθμεί όλα τα δάση ε, και θα τα καταγράψει μια επιστημονική επιτροπή και να γίνει μια χαρτογράφηση. Επιμένω πολύ σε αυτόν τον κατάλογο αρχαίγωνων δασών. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Πόκοβιτ Φρανκ είναι ο επόμενος ομιλητής. Ε, ε, Ευχαριστώ για το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Σήμερα συζητούμε την κατάσταση των δασών στην Ευρώπη. Όλοι γνωρίζουμε ότι ε, τα δάση μας αποτελούν τους πνεύμονες μας, ε, αποτελούν δηλαδή ε, τους, τα σημεία όπου μπορούμε να αποθηκεύσουμε άνθρακα και υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα οποία κατασκευάζονται από ξυλία. Παρ' όλα αυτά, τα κράτη-μέλη βρίσκονται σε διαφορετική κατάσταση σε ό,τι αφορά τη διατήρηση των δασών τους. Στη δική μου χώρα, τη Σλοβενία, έχουμε πάρα πολλά δάση. Το 60% ε, των εκτάσεων μας ε, καλύπτεται από δάση. Και το εν λόγω ποσοστό αυξάνεται όλο και περισσότερο. Αλλά φυσικά και τα δικά μας δάση είναι ευάλωτα σε περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως για παράδειγμα ε, ο παγετός, οι πυρκαγιές αλλά και επιβλαβείς οργανισμοί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εργαστούμε περισσότερο και να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε επίπεδο συνεργειών μεταξύ προγραμμάτων Live, ε, Horizon και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να διαχειριστούμε καλύτερα τα δάση μας ε, στο ε, μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Εκαρίν Μάουρη έχει το λόγο. Μάικρο. Excuse me. In Venice, please. Arvoisa puheenjohtaja, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πέρσι, γύρω στα 15 εκτάρια ε, δασικών εκτάσεων κατακάθεται. Και αυτό ουσιαστικά αντιστοιχεί σε έκταση μεγαλύτερη από το σύνολο της έκτασης ε, διαφόρων ευρωπαϊκών χώρων. Ε, και πραγματικά είχαμε πάρα πολύ μεγάλες ε, συνέπειες ε, και σε ό,τι αφορά το ενεργειακό ε, επίπεδο αλλά και της παραγωγής. Ένας από τους λόγους που οδήγησαν σε όλες αυτές τις πυρκαγιές ήταν ότι υπάρχουν πάρα πολλά δάση τα οποία δεν είχαν τις κατάλληλες διαχείρισης. Όταν έχουμε λοιπόν δάση των οποίων η διαχείριση δεν γίνεται με το σωστό τρόπο, αυτά γίνονται αυτόματα πιο ευάλωτα στις πυρκαγιές. πριν από 60 ε, περίπου χρόνια 100.000 εκταρίων ε, κατακάηκαν στη Φιλανδία, αλλά έκτοτε ουσιαστικά έχουν μειωθεί πάρα πολύ και, είχα, και οι τελευταίες πυρκαγιές αντιστοιχούσαν μόνο σε χίλια εκτάρια στο σύνολό τους. Έχουμε λοιπόν μια δασοκομεία η οποία είναι ε, βιώσιμη και η οποία συμβάλλει στην αποτροπή των δασικών πυρκαγιών. Πράγμα το οποίο μας καθιστά πιο ασφαλής και απέναντι στη κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ. Αν έχει την καλοσύνη να τηρείτε το χρόνο σας, ε, υπάρχουν ε, κάποιοι κανόνες, θα παραμένουμε, θα παραμένουμε στο ένα λεπτό και αν ξεπερνάτε το ένα λεπτό θα είμαι αναγκασμένος να σας διακόψω. Αυτός είναι ο πρώτος κανόνας και ο δεύτερος κανόνας είναι ότι ε, δεν θα λαμβάνει κανείς το λόγο ε, ο οποίος ε, στην προηγούμενη συζήτηση ήδη έλαβε το λόγο μέσω του συστήματος Blue Card. Τα λέω απλά για να υπάρχει σαφήνεια για τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστούμε. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Wallace Mick. Προσφάτως η Ιρλανδική κυβέρνηση δημοσίευσε τους ε, σχετικούς στόχους οι οποίοι είναι 70% για κονοφόρα και 30% πλατήφυλλα. Ουσιαστικά έτσι θα διπλασιαστεί η υφιστάμενη εμπορική δασοκομεία, κάτι το οποίο αντιβαίνει σε κάθε αρχή της ε, βιοπικιλότητας, ε, καθώς έχουμε υπερβολική εξάρτηση από τα κονοφόρα. Δεν χρειαζόμαστε μόνο καλλιέργειες, χρειαζόμαστε τα κατάλληλα δέντρα στα κατάλληλα σημεία. 42% των ε, δέντρων αυτών στην Ιρλανδία πηγαίνει για ενέργεια, το υπόλοιπο για ξυλία. 57% είναι κονοφόρα, οπότε ουσιαστικά ένα μεγάλο ποσοστό των λανδικών δασών είναι δεσμευμένο ως βιομάζα και επιστρέφει στην ε, ατμόσφαιρα ως άνθρακας. Πρόκειται για μια τρελή αντιεπιστημονική πολιτική και θεωρούμε ότι η βιομάζα έχει μηδενικές εκπομπές. Θέλω η Κομισιόν να το ξαναδεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Frau Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ακούστηκαν πολλά και σημαντικά πράγματα. Ένα πράγμα πρέπει να είναι σαφές. Οπωσδήποτε δεν θα σώσουν τα ευρωπαϊκά δάση το παγκόσμιο κλίμα, αλλά σήμερα δείχνουμε ότι μιλάμε σοβαρά όταν μιλάμε για τα δάση στην Ευρώπη και αναζητούμε λύσεις. Γιατί όταν πεθαίνουν τα δάση βλέπετε ότι ε, χάνουμε όλοι και δεν δεσμεύουν άλλο διοξείδιο του άνθρακα πλέον. Γι' αυτό πρέπει το δάσος να το αντιληφθούμε ως μια θαυμάσια πρώτη ύλη και να το προστατεύσουμε αλλά και να το εκμεταλλευτούμε. Και τέλος θα ήθελα να ζητήσω να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φυτέψουμε εκατομμύρια νέα δέντρα στην Ευρώπη και να τους δώσουμε την ευκαιρία στα κράτη-μέλη, στο πλαίσιο της ε, στρατηγικής τους, ε, να το θέσουν αυτό ως πρώτη προτεραιότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Στάνισλαβ Πόλτσακ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε το λόγο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συζητάμε αυτό το σημαντικό θέμα σήμερα. Θα μπορούσαμε να έχουμε συζητήσει πολλά άλλα θέματα, όπως το Brexit, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα για να δείξουμε στους πολίτες ότι μας απασχολούν και αυτά τα ζητήματα. Δεν θα επαναλάβω όσα ήδη ακούστηκαν, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι έχουμε ένα μέσο εδώ πέρα για να προστατεύσουμε τα δάση, τα ευρωπαϊκά ταμεία δηλαδή. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την φύτευση δασών και δέντρων στα κράτη-μέλη εκείνα που υπάρχει ανάγκη. Και επίσης, να συνενωθούν τα αγροτεμάχια πρέπει να βοηθήσουμε περιφέρειες ε, και τις ενώσεις ιδιοκτητών γης. Υπάρχει μάλιστα στην ε, Τσεχία μια τέτοια ένωση και πρέπει να στηρίξουμε και την σχετική έρευνα για να αντιμετωπίσουμε τα ζυζάνια που βλάπτουν τα δάση. Έχουμε πολλά εργαλεία λοιπόν στη διάθεσή μας και εγώ θα στηρίξω το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Και τώρα περνάμε στον τελευταίο μιλητή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα δάση έχουν υποφέρει και είναι απόλυτα σαφές ότι η κατάσταση είναι τραγική, δεν υπάρχει απαραίτητη φροντίδα. Πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε και να λάβουμε σοβαρά μέτρα. Ε, το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα με τα δικά μας. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κάτι εδώ, ε, στις δικές μας τις χώρες. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου ότι η ε, ρήπανση δεν γνωρίζει όρια, ούτε και η κλιματική αλλαγή. η φύση δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς ανθρώπους, αλλά και οι άνθρωποι ε, δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς τη φύση. Γι' αυτό λοιπόν εγώ είμαι υπέρ του να εκταμνευτούν περισσότερα κονδύλια στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για την προστασία της φύσης, για την προστασία και τη διατήρηση των δασών. Αυτό είναι μια πολύ καλή επένδυση. Έκλεισε λοιπόν η ημερήσια διάταξη. Ε, τώρα θα δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Αρία κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές για τις ε, παρεμβάσεις τους ε, που κατέδειξαν το ενδιαφέρον που υπάρχει για τα δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι δεσμευμένη να προστατεύσει τα δάση που υπάρχουν, όπως αναφέρεται και στην πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τα δάση ανά την υφήλιο, γιατί έτσι μπορούμε να έχουμε καλύτερη αντίσταση στην ε, κλιματική αλλαγή, να ε, διαφυλάξουμε την βιοπικιλότητα και να προσφέρουμε βασικές υπηρεσίες ε, στην κοινωνία μας. Η κοινή γεωργική πολιτική με τη νέα ισορροπία των υπευθυνοτήτων των ευθυνών ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει στο να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη και μια σωστή στρατηγική. Αναγνωρίζεται ο ρόλος προς μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον, μια βιοοικονομία προστασία της βιοπικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Έχοντας κατά νου ε, τη δήλωση της κυρίας Φόντερ Λάιεν όσον αφορά στη βιοπικιλότητα και την αλλαγή, ε, νομίζω ότι μπορεί να, μπορούν να υπάρξουν και περαιτέρω μέτρα ε, στο πλαίσιο της μελλοντική βιοπικιλότητας για να προστατευτεί η ε, διατήρηση και η αντίσταση των ενωσιακών δασών. Η αποκατάσταση είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για το μέλλον. Αυτό βέβαια στο νέο στρατηγικό πλαίσιο για τα δάση μέχρι το 2020. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε λοιπόν τη συζήτηση για την κατάσταση των δασών ε, και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της σημερινή διάταξης ε, που ε, πρόκειται για μια προφορική ερώτηση που αφορά στη δυνατότητα κατοχήρωσης φυτών και κατ' ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα εύρεση τεχνίας από την Επιτροπή Γεωργίας. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στο συντάκτη της ερώτησης, τον κύριο Νόρμπερτ Λίντς. Παρακαλώ κύριε Λίντς, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, το να υπάρχει ε, δυνατότητα πρόσβασης ε, στο ε, υλικό που αφορά τα φυτά χωρίς καμία, κανένα εμπόδιο. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό για τη γενετική ποικιλομορφία των φυτών. Στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας στις 14 Σεπτεμβρίου όλοι συμφώνησαν ότι πράγματι έτσι είναι τα πράγματα. Υπάρχει μια απόφαση του Δεκεμβρίου του 2018 του Γραφείου Ευρεσιτεχνίας και δυστυχώς όμως απόφαση υπάρχουν πλέον προβλήματα στην απρόσκοπτη πρόσβαση. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε να εκπαιμφθεί ένα σημαντικό μήνυμα και εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας θα ήθελα να φέρω ε, και να εξηγήσω το γιατί κάνουμε αυτή την ερώτηση προς την Κομισιόν ε, σύμφωνα με το άρθρο 136. Το 2015 η ε, το τεχνικό εφετείο του ε, Γραφείου Διπλωμάτων Ευρυστοχνίας ε, αποφάσισε ότι βιολογικό υλικό, ε, όπως είναι αυτό που αφορά τα φυτά και τους σπόρους, πρέπει να κατοχυρώνονται. Και εκεί αναφέρθηκαν κυρίως μία ποικιλία ντομάτας και τον μπρόκολο. Το 2015 το Κοινοβούλιο δημοσίευσε μία απόφαση σχετικά με τα φυτά και αυτή κατ' ουσίαν ε, είναι ε, η Οδηγία 9844 η οποία προσφέρει την κατοχήρωση των φυτών. Ε, το 2016 η Κομισιόν είπε ότι ποτέ δεν ήταν ο στόχος τα διπλώματα έβρεση τεχνίας να δίδονται σε όλα τα φυτά μετά λοιπόν από αυτήν την απόφαση προέκυψε ε, μια αντιπαλότητα, μια αντιμαχία ανάμεσα σε διάφορες αρμόδιες υπηρεσίες. Ε, είχαμε την ε, διαφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γραφείο Ευρεσιτεχνίας. Και τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θα πρέπει να είναι δυνατή η κατοχήρωση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Το επόμενο βήμα ήταν στο ανώτατο, ε, στην ανώτατη βαθμίδα προσφυγών ε, του, του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και η απόφαση ήταν τελεσίδικη. Εκεί λοιπόν υπάρχουν ε, οι γραπτέ ερωτήσει που κατατίθενται. Η 1η Οκτωβρίου του 2019 ήταν η καταληκτική ημερομηνία. Η Επιτροπή Γεωργία σήμερα έχει δύο ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη ερώτηση είναι κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να καταθέσει μια γραπτή ερώτηση προς την τελευταία βαθμίδα προσφυγών του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία, έτσι ώστε να ε, μπορέσει να προστατεύσει το γενικότερο συμφέρον σχετικά με την κατοχήρωση των φυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερον ποια μέτρα θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι τα φυτά τα οποία προέρχονται από φυσικέ διεργασίε, τα φυτά αυτά δεν είναι δυνατόν να κατοχυρώνονται με διπλώματα ευρεσιτεχνία. Η δική μα η δωρητές, οι γεωργίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλου χρειάζονται την σαφήνεια για την καινοτομία που θα υπάρξει στο μέλλον. Σα ευχαριστώ πολύ. Η ερώτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την κυρία Μπιενκόφσκα. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ. Σα ευχαριστώ πολύ που θέτετε αυτό το ζήτημα που όπως ακούσαμε είναι πολύ σημαντικό να είναι ξεκάθαρο για όλους. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με το δεύτερο τμήμα της ερώτησής σας και η απάντηση εδώ είναι αρκετά απλή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει δράση για να διασφαλίσει ότι οι προϊόντα τα οποία προέρχονται από κατ' ουσίαν φυσικέ διαδικασίε ε, δεν κατοχυρώνονται με διπλώματα ευρεσιτεχνία. Είμαστε σε επαφή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο και με τι χώρε μέλη, αλλά και με τον κλάδο όσον αφορά το θέμα αυτό του δηλαδή να μην κατοχυρώνονται με ευρεσιτεχνία αυτά τα προϊόντα αναφέρθηκε και το Δεκέμβριο του 2015 στο ψήφισμά σα Το 2016 οθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωμα για κάποιο άρθρο τη οδηγία όσον αφορά τη νομική προστασία των ε, βιοτεχνολογικών εφευρέσεων. Σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκεί ότι προϊόντα φυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί από κατουσίαν ε, βιολογική διαδικασία ε, δεν κατοχυρώνονται από ευρεσιτεχνία και στη συνέχεια οι χώρες ε, μέλη προχώρησαν στην ε, ερμηνεία και στην πρακτική στις χώρες μέλη. Στις χώρες τους δηλαδή. Και τώρα έρχομαι στο δεύτερο τμήμα. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα είναι παρούσα στην διαδικασία που έχει ε, θέσει σε κίνηση η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνίας και η σύμβαση μεν δεν αποτελεί σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι όμως προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στη σύμβαση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Βρεσιτεχνίας και της δικιάς μας οδηγίας για τις ε, βιοτεχνολογίες. Έτσι λοιπόν θα δούμε πώς θα προχωρήσει το θέμα και εμείς θα επιμείνουμε για τα ζητήματα αυτά τα οποία αποκλείονται σύμφωνα με τη δικιά μας νομοθεσία από την ευρεσιτεχνία. Υπάρχει όμως η σύμβαση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνίας και όπως ε, το έχουμε σημειώσει ήδη από το 2016, οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, το Συμβούλιο και άλλες χώρες συμβαλόμενες έχουν συμφωνήσει με αυτό. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το συμφέρον του κλάδου και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των καταναλωτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε τώρα στην συζήτηση. Πρώτος που ζήτησε τον λόγο είναι η κυρία Σράιερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ. Ως Κοινοβούλιο απαιτήσαμε ξεκάθαρα το 2015 να παραμένουν ελεύθερα διαθέσιμα τα βιολογικά δεδομένα που αφορούν την ανάπτυξη νέων ειδών. Και αυτό αφορά ακριβώς και την κατοχύρωση των φυτών μέσω μιας διαδικασίας η οποία είναι κατ' ουσίαν βιολογική. Ε, από ό,τι φαίνεται όμως ε, στην παράγραφο 2 ε, της αποφάσεως έχουμε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεστεχνιών η οποία αντιβαίνει την απόφαση της ε, Κομισιόν καθώς είχαμε το Γραφείο Εφέσεων το οποίο στις 5 Δεκεμβρίου 2018 αποφάσισε ότι ο κανόνας αυτός ε, που είχε δημιουργηθεί είναι άκυρος. Δεν είναι δυνατόν όμως να προσπαθεί να επιλύσει μόνο του το ζήτημα αυτό ένας τεχνικός φορέας χωρίς να λαμβάνει υπόψη του συνομοθέτε μεταξύ των οποίων το Κοινοβούλιο. Από τη δήλωση τη Κομισιόν είναι σαφέ πω Κατά την κατάρτιση τη οδηγία περί ποτέ Κομισιόν, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο δεν είχαν ω στόχο να επιτρέψουν την κατοχήρωση διαδικασιών ε, οι οποίες είναι κατ' ουσίαν βιολογικές. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, είναι λοιπόν δημοκρατική ανάγκη η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση αυτή στο Συμβούλιο Εφέσεων της ε, Υπηρεσίας ε, Διπλωμάτων Τεχνίας. Και θα πρέπει να καταστεί αδύνατον η κατοχήρωση, να υπάρχει κατοχήρωση βιολογικών διεργασιών το συντομότερο δυνατόν. Θα πρέπει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε αντίστοιχη περίπτωση να προσφύγουν σε άλλα νομικά μέσα. Εν ολίγης, δεν μπορεί να υπάρχει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας επί της ζωής. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ανδρία... ο κύριος Ανδρία, με συγχωρείτε. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εμείς δεν θέλουμε τα προϊόντα τα οποία προέρχονται από βιολογική διαδικασία να κατοχυρώνονται με ευρεσιτεχνία είναι απόλυτα φυσιολογικό. Εμείς δεν θέλουμε οι πολυεθνικές ή πλούσιες ε, βιομηχανίες ε, αγροτροφίμων να επωφελούνται από κάτι τέτοιο. Και εμείς θα αγωνιστούμε υπέρ της καινοτομία. Είμαστε υπέρ της ποικιλομορφία των καλλιεργών. Και θα αγωνιστούμε προκειμένου υγεία των πολιτών να αποτελεί προτεραιότητα. Να μπορεί εύκολα κανείς να έχει πρόσβαση στα φυτά. Είναι πολύ βασικό αυτό για να υποφεληθεί από αυτό η καινοτομία του κλάδου, αλλά και ο διατροφικός τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν να απαγορεύουμε την χρήση των φυτών που βρίσκονται στη φύση για να δημιουργήσουν καινοτομία και να μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρους. Εγώ δεν θέλω μονοπόλια στη ζωή όταν οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ως μόνο στόχο το κέρδος και τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε. Η κυρία Χαϊτεμα. Ο κύριος Χαϊτεμα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, με το ψήφισμα αυτό θέλουμε οι έβρεση τεχνίες να κατοχυρώνονται. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Όμω, με τι αποφάσει του οδηγεί σε συζητήσει για το κατά πόσο επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται τεράστια αβεβαιότητα και από τους καλλιεργητές αλλά και από τους καταναλωτές. Ε, το θέμα της ντομάτας, της γεύσης της ή της πιπεριάς ή οτιδήποτε αυτά είναι πράγματα τα οποία βρίσκονται στη φύση. Είναι τρελό λοιπόν μια επιχείρηση να μπορεί να παίρνει δίπλωμα ευρωσιτεχνίας και να κατοχυρώνει τέτοια προϊόντα με ευρεσιτεχνία και επιτακηθικά αν το δούμε το θέμα. Επίσης είναι αυτό περίεργο. Πρέπει να δούμε και ποιες είναι οι συνέπειες αν ε, γίνει δυνατό κάτι τέτοιο. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες επιχειρήσεις θα έχουν όλα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ε, στα χέρια τους και θα αποφασίζουν ό,τι θέλουν για τα τρόφιμά μας και θα αποφασίζουν και ό,τι θέλουν για τις τιμές, το πόσο θα κοστίζουν τα τρόφιμά μας. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Εμείς δεν ε, θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλουμε ο καθένας να μπορεί να χρησιμοποιεί τους σπόρους για να φτιάχνει και καινούργια προϊόντα. Βέβαια με κάποια ασφάλεια. Δεν θα πρέπει να τίθονται σε κίνδυνο τα τρόφιμά μας κάθε φορά που έχουμε νέα προϊόντα και ίσως και νέες ε, αρρώστιες. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε την ε, εμπορία. Αυτό ναι, αλλά το να κατοχυρώνονται με βρεσιτεχνία τα φυτά, αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό είναι το όλο άκρο. Γι' αυτό λοιπόν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να στηρίξουμε την ε, πρόθεσή μας που δεν ήταν ποτέ στα φυσικά δημιουργούμενα φυτά να τα κατοχυρώσουμε με ευρεσιτεχνία. Ευχαριστώ για τους πράσινους ο κ. Μάρτιν Χόισλινγκ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι εξοργιστικό το ότι για τρίτη φορά συζητάμε αυτό το θέμα. Ήδη το 2012 είχαμε ψήφισμα, το 2015 και πάλι. Γιατί η υπηρεσία για την ευρεστεχνία αγνοεί αυτό το οποίο θέλουν οι πολιτικοί, δηλαδή να μην υπάρχει ευρεσιτεχνία επί της ζωής. Αυτό το οποίο λέμε εδώ πέρα, δηλαδή κατ' ουσίαν βιολογική διεργασία. Βεβαίω, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνία θέλει να εκδίδει διπλώματα ευρεσιτεχνία. Είναι προ το συμφέρον του. Αλλά εδώ πέρα πρέπει η πολιτική, εμεί, να ε, παίξουμε τον ε, ρόλο μας και η Κομισιόν ιδιαίτερα, γιατί δεν είναι δυνατόν ένα θεσμικό όργανο να ε, αγνοεί τις αποφάσεις του νομοθέτη αναφέραμε τον μπρόκολο και την ντομάτα, αλλά είναι ζήτημα αρχής. Εάν δεν προστατεύσουμε τώρα τους αγρότες, τους μικροκαλλιεργητές, να χρησιμοποιήσουν τους σπόρους τους, μακροπρόθεσμα και άλλες εταιρείες θα προσπαθήσουν ε, να κατοχυρώσουν διπλώματα ευρυστεχνίας, να διασφαλίσουν ε, δικαιώματα και αυτοί οι οποίοι τα χρειάζονται περισσότερο, οι μικροκαλλιεργητές και οι αγρότες θα χάσουν τα δικαιώματά τους. Γι' αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, να σταματήσει αυτό το οποίο κάνει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ωρές Σα ευχαριστώ και ο Ντάβιντ Ιβαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το να δίνονται διπλώματα ευρεσιτεχνίας για κάποια είδη ντομάτας ή μπρόκολου αντιβαίνει τη σύμβαση του ΟΗΕ περί βιοποικιλότητας και το πρωτόκολλο της Ναγκόγια στην σύμβαση αυτή και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και το σχετικό εκτελεστικό πρωτόκολλο. Τα συμβαλόμενα, μέρα, τα συμβαλόμενα μέλη με είναι ε, όλα μέλη και των ε, συνθήκων αυτών, αλλά και του Γραφείου Ευρεσιτεχνίας, ε, το οποίο υποτίθεται ότι επιλύει τις διαφωνίες. Γι' αυτό προτείνουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τους εκπροσώπους τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ε, Υπηρεσίας Περί Ευρεσιτεχνιών για να ακυρώσουν τις υφιστάμενες αυτές πατέντες για τα ίδια αυτά, τα φυτά αυτά, και το ίδιο και σε υπόλοιπε 200 περιπτώσει που εκκρεμούν. Σας ευχαριστώ. Ο κύριο Ράσιον, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι λάθος αυτό που κάνουμε. Δεν ξέρω πώ αλλιώ να προσδιορίσω το δρόμο που έχουμε πάρει όταν θέλουμε να κατοχυρώσουμε φυτά κατ' ουσίαν από βιολογική διαδικασία με διπλώματα ευρεσιτεχνία. Αυτό είναι λάθο και οδηγεί σε μονοπωλιακέ θέσει. Το τίμημα είναι ιδιαίτερα υψηλό, πάρα πολύ υψηλό πιστεύουμε εμείς. Διότι οι επιχειρήσεις που είναι φυτόρια για παράδειγμα χάνουν την ελεύθερη πρόσβαση σε γενετικό υλικό. Και αυτή η ελεύθερη πρόσβαση είναι πολύ βασική για να μπορούμε να δημιουργούμε νέα είδη. Έτσι λοιπόν ξέρω ότι υπάρχει εδώ ευρεία συνένεση. Οπότε αυτή τη βδομάδα να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνία για να του εξηγήσουμε ότι πρέπει να καταλήψουν αυτή την προσπάθεια και μάλιστα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Εννοείται φυσικά ότι πρέπει να προστατεύσουμε την πνευματική ιδιοκτησία επαρκώς. Αλλά γι' αυτό χρειάζεται ένα ισορροπημένο σύστημα. Ένα σύστημα δικαιωμάτων ε, διασταύρωσης και καλλιέργειας το να, να δίνουμε τέτοια ευρεσιτεχνία σε φυτά από φυσιολογική διαδικασία είναι λάθος. Τα φυτά ανήκουν σε όλους μας. Και θα μπορούσα να το πω κι αλλιώς. Αποτελούν δημιουργήματα του Θεού Δημιουργού. Και εμείς είμαστε εδώ για να τα διαχειριστούμε και μόνο. Ευχαριστώ. Thank you. Madame Η κυρία Σάντρα Περέρα. Δεν μπορεί κανείς ε, να κατοχυρώσει είδη τα οποία έχουν υποστεί μεταλλαγή, όμως ε, υπάρχουν αυθεντικά μονοπόλια τους ε, παραγωγούς. Οι πολυεθνικές εταιρείε ελέγχουν την αγορά και την του μεταξύ τους και δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Για τους μικρούς γεωργούς δεν είναι πλέον δυνατόν να επιτύχουν την ποικιλομορφία. Ε, οι μικροί γεωργοί εξαρτώνται από τις ε, πολυεθνικές εταιρείε. Ε, υπάρχει η μοριακή και η γενετική μετάλλαξη και αυτό πολύ το εκμεταλλεύουν. Τα προϊόντα τα οποία απορρέουν από αυτή τη τεχνολογία δεν είναι αποδεκτά. Υπάρχει και το δικαίωμα ε, του δημιουργού και δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ε, και για αυτούς τους οργανισμούς. Ε, τα προϊόντα τα οποία πορέουν από τέτοιου είδους διασταυρώσεις δεν είναι αποδεκτά. Παναλαμβάνω λοιπόν, υπάρχουν ολόκληρα γονίδια τα οποία χρησιμοποιούνται για τέτοιου είδους τεχνολογίες. Ο κύριος Μπούντα Ντάνιελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία, η έρευνα και η καινοτομία δεν μπορούν να μπλοκάρονται από διοικητικέ διαδικασίε, γιατί κυρίω η γεωργία εξαρτώνται από την έρευνα και την καινοτομία. Σήμερα υπάρχει μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να την αγνοούμε. Η δημογραφική αύξηση ε, περιορίζει του πόρου, που έτσι και αλλιώ είναι περιορισμένοι. Πρόβλημα είναι και η κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά μα αναγκάζουν στο να δραστηριοποιηθούμε. Χρειαζόμαστε πόρου, μηχανισμού ε, και διαδικασίε παραγωγή για τρόφιμα, τα οποία θα πρέπει να είναι και ποιοτικά και προσιτά. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι τα φυτά ε, τα οποία προκύπτουν από παραδοσιακές διαδικασίες ε, δεν είναι απαραίτητο να κατοχυρώνονται γιατί αυτό θα ήταν τραγικό και για τους ίδιους τους γεωργούς ε, το να είναι αναγκασμένοι να προβαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Τραγικό θα ήταν και για την έρευνα και σήμερα τη χρειαζόμαστε την έρευνα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους καταναλωτές. Αυτή είναι εκείνοι που θα κληθούν να πληρώσουν από πλευράς ε, κατάχρησης, αυτή την κατάχρηση από πλευράς του ε, Γραφείου ευρεστεχνιών Βεβαίως ε, δεν πρέπει την τελευταία στιγμή να προσπαθούμε να δραστηριοποιηθούμε και να σώσουμε την κατάσταση. Το αντίθετο πρέπει να ισχύει. Εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλουμε να εκπέμψουμε ένα σαφές μήνυμα. Οι φυσικές διαδικασίες δεν πρέπει να κατοχυρώνονται. Σας ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Παόλο Ντικάστρο. Sì. Presidente Commissario Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, τη στιγμή ε, που ε, έχουμε την κερδομία, έχουμε τα γονίδια των φυτών και είναι ο μόνος τρόπος για να ε, περιορίσουμε την επιδίνωση στην γεωργία, αυτό που αποφάσισε το Γραφείο Ευρωστεχνών είναι απαράδεκτο. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να περιοριστεί η καταχώρηση των φυτών. Δεν μπορεί να υπάρχει κίνδυνος για την έρευνα με πάρα πολλές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα της γεωργίας και επίσης και στην υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Επίτροπε σας καλούμε να παρέμβετε το στομότερο δυνατόν, να παρουσιάσετε τις απαραίτητες ε, δικές σας παρατηρήσεις γιατί αυτή η διαδικασία πηγαίνει αντίθετα με αυτό που επιθυμούν οι νομιθέτε. Να επαναφέρετε τη νομοθετική ε, σταθερότητα έτσι ώστε η Γεωργία να είναι όλο και πιο ε, στην προμετωπίδα της ε, ε, προόδου. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με φιλόδοξο τρόπο στα αιτήματα των εκατομμυρίων πολιτών. Η κυρία Μιλά. Κύριε Πρόεδρε, Κυρία Επίτροπε, η απόφαση της ε, του τεχνικού εφετείου του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνήσεων να δίδονται διπλώματα ευρεσιτεχνία για φυτά τα οποία έχουν προκύψει από την κλασική παραγωγή, κατά την άποψη των γεωργών δεν είναι σωστή. Ή για μένα ε, η ελεύθερη πρόσβαση είναι πολύ σημαντική έτσι ώστε να παραμείνει και αυτή η δυνατότητα των Ευρωπαίων καλλιεργητών. Εγώ λοιπόν θέλω να υπάρχει ποικιλομορφία των σπόρων στην Ευρώπη και θέλω και οι μικροί καλλιεργητές φυτών να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους γενετικούς σπόρους. Η ελεύθερη πρόσβαση στους σπόρους είναι καθοριστικό στοιχείο για να καλλιεργούνται νέες ποικιλίε οι θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις προκλήσεις τη κλιματική αλλαγή. Ελπίζω λοιπόν το μεγάλο άλλο το ανώτατο τεχνικό αυτό εφετείο του Γραφείου Ευρυστεχνιών να αναθεωρήσει την απόφαση έτσι ώστε το μέλλον να μην είναι απαραίτητο να κατοχυρώνονται τα φυτά. Παρακαλώ, κύριος Μπιτό. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η ομάδα των Πρασίνων πάντα ήταν κατά των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία στα φύτα, το ακούσαμε και πριν. Και μετά από όσο έχω ακούσει, τελικά νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Αλλά όσον αφορά τη διαδικασία, εκεί είναι το πιο σοβαρό, γιατί ποιο καθορίζει την νομοθεσία στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνία ή το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Εδώ και τόσα χρόνια παράνομες ευρεσιτεχνίες δίνονται για τα μπρόκολα και για άλλα φυτά και ακόμα και για ζώα, για το σολομό για παράδειγμα. Ε, μπορεί να μην είναι τέλειο το δικό μας σύστημα, αλλά επιτρέπει αν μη τι άλλο στους αγρότες να μπορούν να ρίξουν τους σπόρους τους και να καλλιεργήσουν όλα τα είδη. Εξάλλου ακριβώς επειδή είναι αποτελεσματική χρήση των σπόρων αυτών για την ε, επίκυλομορφία, την γενετική, Γι' αυτό τους το επιτρέψαμε και στην ε, συζήτηση που έχει γίνει φάνηκε ότι ήταν πολύ αποτελεσματική αυτή η μέθοδος. Οπότε σε διεθνές επίπεδο ε, παντού αυτό είναι το σωστό. Ενώ βέβαια οι πολυεθνικές πιέζουν και διακόπτεται ο μιλητής. Ε, ευχαριστούμε ο κύριος Λεμπρετόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το 2015 το Ευρωπαϊκό Γραφείο Βρεσιτεχνία είπε ότι είναι δυνατόν να δώσουμε βρεσιτεχνία σε τομάτες και μπρόκολα. Μετά άλλαξε θέση επειδή ακριβώ υπήρξαν πάρα πολλέ διαμαρτυρίες. Όμω, δυστυχώ, 18 Δεκεμβρίου του 2018 το Τεχνικό Συμβούλιο του γραφείου αυτού τροποποίησε τη θέση του. Και η Επιτροπή Γεωργίας, όπου είμαι και εγώ, ζητάει από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή να διαμαρτυρηθεί. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε τη θέση μας ότι είμαστε κατά της ευρεσιτεχνίας στη ζωή. Μπορεί να υπάρχουν πολύ ισχυρά λόμπι, αλλά περί αυτού πρόκειται τίποτα άλλο. Η διατήρηση λοιπόν τη βιοπικιλομορφία, η προστασία των καταναλωτών και των αγροτών μα είναι πράγματα που εξαρτώνται από εμά. Τέλο, Ήδη από το 1961 ε, υπάρχει νομική προστασία των σπόρων για την έρευνα. Πρόκειται δηλαδή για πιστοποιητικά, το οποίο είναι πολύ καλύτερα από ό,τι η ευρεσιτεχνία για τα δικαιώματα των ε, αγροτών και των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, Είμαι για πρώτη φορά εδώ, οπότε να ξέρουμε ότι 500 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθούν. Ο κύριος Αμπιλάρ είναι ο επόμενος. Η κυρία Αγγιλάρ. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ όλους για το ένα λεπτό σιγή για τα θύματα από τις πλημμύρες στην Ισπανία. Η συμφωνία μεταξύ μας δείχνει ότι επήγει το θέμα. Δεν είναι δυνατόν παρά το πνεύμα του νομοθέτη να ανοίγουμε την πόρτα στην κατοχύρωση φυτών με διπλώματα ευρεσιτεχνία. Έτσι καταστρέφονται και οι μικρές επιχειρήσεις αλλά και ολόκληρη η γεωργία. Κι όμως οι αποφάσεις του εφετείου, του γραφείου ευρεσιτεχνία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν άλοθη για να αλλάξουμε εμεί τη θέση μα και να μην προστατεύουμε το σύστημα που έχουμε σήμερα που λειτουργεί τόσο καλά και που προστατεύει όλου του ενδιαφερόμενους. Δεν είναι δυνατόν να αφισβητείτε ένα σύστημα ε, το οποίο στηρίζει την ανάπτυξη και λειτουργεί αποτελεσματικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Χάζεκα μέχρι τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λοιπόν, εδώ και 4 δισεκατομμύρια χρόνια έχουμε ζωή στη γη και αυτή η ζωή δεν ανήκει σε κανέναν, μα σε κανέναν και ούτε πρέπει να ανήκει σε κάποιον. Όλη αυτή η ιδέα, φυτά, ζώα και βιολογικέ διαδικασίε να κατοχυρώνονται από διπλώματα ευρεσιτεχνία είναι κάτι πολύ περίεργο. Δυστυχώ όμω αυτό ακριβώ συμβαίνει. Εξάλλου υπάρχει ήδη ευρεσιτεχνία για σολομούς και πέστροφες, τις οποίες ταΐζουν με φυτά έτσι ώστε να ανέβει το ποσοστό των κορεσμένων λοιπόν σε αυτά. Και τα έχει εφεύρει κανεί αυτού του ολομού και αυτέ τι πέστροφε. Και όμω. Λοιπόν, αυτού του είδου η ευρεσιτεχνία βοηθάει τα μονοπόλια και καταστρέφει του πολιτέ, του αγρότε. Εκεί είναι κάτι με το οποίο είμαστε αντίθετοι όλοι εμεί, αλλά και η Επιτροπή. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο. Παρ' όλα αυτά, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνία χορηγεί κατοχυρώσει στι πολυεθνικές τροφίμων. Είναι απαράδεκτο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλου θα πρέπει να αντισταθεί στην κατοχήρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνία για τη ζωή. Τέλο, στα δισεκατομμύρια επιχορηγήσεων για την αντατική κτηνοτροφία επίση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο τώρα έχει η κυρία Πιτσέρνο, τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ συμφωνώ με όλους εκείνους, ε, με όλους τους συναντέλφους που έχουν λάβει το λόγο και που έχουν ήδη εκφράσει την αντίθεσή τους ε, προς αυτήν την απόφαση που πραγματικά είναι κατανόητη. Είναι η απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΕΓΔΕ. Κατά τα άλλα, ε, όσον αφορά τη θέση του Κοινοβουλίου για τις για τα διπλώματα και την κατοχήρωση μέσα από φυσικές διαργασίες. Νομίζω ότι είναι σαφή η θέση μας, η θέση μας από το 2015, όταν εδώ, σε αυτή την αίθουσα, σας το επενθυμίζω, με καθαρή πλειοψηφία αποφανθήκαμε κατά αυτών των ε, διπλωμάτων. Με τον ίδιο τρόπο εκφράστηκε και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα δηλαδή εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την πολιτική βούληση του να μην είναι απαραίτητο να χωρίσουμε χορηγούνται διπλώματα βρεστεχνίας μέσα από, στα φυτά που έχουν προκύψει μέσα από φυσικές διεργασίες. Γι' αυτό, κυρία Επίτροπε, καλούμε εσά και καλούμε την Επιτροπή να εψώσει τη φωνή της έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η διαδικασία που έχει ξεκινήσει από το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία. Πρέπει να προστατεύει η διαδικασία της φυσικής επιλογής αλλά κυρίως ε, το γενικό συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην συνάδελφο Μελχιόρα από την ομάδα Ρινιού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το 2014 έγιναν εκλογές στην Δανία και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έγινε και ένα δημοψήφισμα για το εάν θα γινόμασταν μέλος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τις Τεχνίες. Ε, κερδίσαμε ε, και είπαμε να γίνουμε μέλο, αλλά επιμείναμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν διπλώματα βρυστεχνίες ε, σε φυτά και ζώα. Εάν δεν είναι αντιληπτό αυτό το μήνυμα, θα πρέπει να το πούμε πιο ξεκάθαρα στο γραφείο Ευρεστεχνία. Στην Τζαμαϊκά υπάρχει μια άγρια πίπεριά, η οποία αντιστέκεται στα διάφορα ζυζάνια, και τώρα κάποιος έβγαλε ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ε, επί του φυτού αυτού. Ένα ζήτημα το οποίο ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Πρέπει άρα ε, να ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους αγρότες, αλλά και για τη δημοκρατία μας. Να καταλήξουμε κάπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο έχει τώρα η κυρία Βίνερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι ντομάτες δεν είναι μηχανήματα, τα μπρόκολα δεν είναι τεχνικές διαδικασίες. Άρα δεν μπορεί να υπάρχουν διπλώματα βριστεχνίας. Με την ε, ερμηνεία αυτή λοιπόν εδώ πέρα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρυστεχνίας ε, διαφωνούμε πλήρως. Υπάρχει μεγάλος ε, κίνδυνος η καλλιεργητές και οι κτηνοτρόφοι ε, να μην έχουν πλέον πρόσβαση στα είδη τα οποία χρειάζονται. Ένα μονοπόλιο ολίγων παραγωγών σπόρων που θα σκέφτονται μόνο τα κέρδη τους πρέπει να εμποδιστεί. Είναι κάτι το παράδεκτο. Επίσης ε, είναι ξεκάθαρο ότι εδώ πέρα δεν εξυπηρετεί την πολιτική βούληση και το κοινό καλό το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνίας, αλλά κάποια οικονομικά συμφέροντα. Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα ότι ο Επίτροπος ο Αρμόδιος για τη Γεωργία, ο κύριος Βοητσικόφσκι, ως Ευρωβουλευτής ήταν σαφώς κατά των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας επιφυτών. Πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθούμε εδώ, να επιβάλλουμε τη θέληση του Κοινοβουλίου και να κάνουμε κάτι κατά αυτής της ε, απόφασης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Τον λόγο έχει ο κύριος ε, Ταραμπέλα τώρα, του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτες. Ε, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είναι μια επικίνδυνη διαδικασία. Οι επιχειρήσει σπόρων, οι πολυεθνικές, θέλουν να έχουν το μονοπόλιο στη ζωή και να ασχοληθούν μόνοι τους με την πρόοδο έτσι τουλάχιστον ε, υποστηρίζουν, θέλουν την πρόοδο στη ζωή. Είναι όμως η υποκρισία όλα αυτά. Τον Μάρτιο που μας πέρασε, πολλές κυβερνήσεις εκφράστηκαν στο Συμβούλιο στηρίζοντας το ερμηνευτικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2016... που λέει ότι φυτά τα οποία είναι κατουσία από βιολογική διαδικασία δεν πρέπει να κατοχυρώνονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Αυτό το κατ' από βιολογική διαδικασία όντως δεν πρέπει να κατοχυρώνεται από ευρεσιτεχνία και αυτή είναι η καλύτερη εγγύηση για τους αγρότες μας αλλά και για τον κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γκυλέρα έχει τώρα το λόγο εκ μέρους των σοσιαλιστών, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ολοκληρώνεται η συζήτηση και πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ με την ομοφωνία που ακούστηκε εδώ στο σώμα από όλες τις πολιτικές ομάδες και από όλους τους συναδέρφους. Υπάρχει μια ομοφωνία η οποία εκφράζεται και στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην κυρία Βινκόφσκα, να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα ξεκάθαρο και αναφεσβήτητο από την Επιτροπή Γεωργίας και από εδώ, ότι δηλαδή δεν είναι δυνατόν να κατοχυρώνονται διπλώματα ευρεσιτεχνία σε φυτά από κατ' βιολογική διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή έχουμε χρόνο μέχρι την 1η Οκτωβρίου, γι' αυτό το ψηφισμά μας, γι' αυτό και η προφορική ερώτηση. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα, το οποίο δείχνει ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο γραφείο ευρεσιτεχνίας. Είναι θέμα συμφέροντος του κόσμου γενικά και να το πούμε ξεκάθαρα ότι δεν θέλουμε τέτοιε κατοχυρώσει. Είναι σαφέστατη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζουμε να σταθεί στο ύψο των περιστάσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώνει εδώ πέρα η συζήτηση και ήρθε η ώρα του ΚΕΤΣΤΙΑΗ. Τρία αιτήματα έχω λάβει. Να δώσω τον λόγο στην κυρία Σόιντροβα. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον την Επίτροπο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χαίρομαι για το ότι όλοι συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ευρεστεχνία επιφυτών και ζώων. Είναι ανοησία. Αλλά φαίνεται ότι διαφωνεί μαζί μας ε, το γραφείο περί γιατί φαίνεται ότι έχει πέσει θύμα του λόμπι της ε, βιομηχανίας. Ε, θα πρέπει λοιπόν εδώ πέρα ε, η Κομισιόν να ακολουθήσει αυτά τα οποία λέει το Συμβούλιο, το οποίο συμφωνεί μαζί μας. Επαφείται πλέον στα κράτη-μέλη να επιβάλλουν την θέλησή τους, όπως είχαμε διαπραγματευτεί, να περάσουν τη θέλησή τους λοιπόν εντός του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνιών. Οπότε εγώ θα ήμουν υπέρ του να συνεχίσουμε αυτήν την πρωτοβουλία, να συνεργαστούμε με Κομισιόν και κράτη-μέλη και ελπίζω ότι αν κάνουμε κάτι τέτοιο θα καταφέρουμε να ξεμπερδέψουμε αυτές τις ανοησίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως, τώρα τον λόγο στον κύριο Wallace. Κυρία Πρόεδρε, είναι αστείο να θεωρεί το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υπηρεσία ότι μπορεί να εκδώσει διπλώματα ευρεσιτεχνία επί φυτών. Έχουμε φυσικές ποικιλίε της ντομάτα και του μπρόκολου που κατοχυρώνονται. Δηλαδή, πού τα βρίσκουν. Οι πολυεθνικές ήδη έχουν αρνητική επίπτωση στη ζωή μας και θα ήταν τρέλα να του επιτρέψουμε να έχουν μονοπόλιο στην ζωή να ασκούν πίεση στους αγρότες και να εμπορευματοποιούν κάθε πτυχή της ζωής μας. Το κάνουν ήδη με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που δεν πρέπει επίση να ανεχτούμε. Πρέπει να απαιτήσετε να σεβαστούν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που αποκλείει του ζωντανού οργανισμού. τους φυσικούς οργανισμούς. Είναι κάτι το αδιανόητο, έχει τρελαθεί ο καπιταλισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κύριος Ντόρφμαν, τελευταίος. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Εγώ νομίζω στην Ευρώπη μερικές φορές πιστεύουμε ότι οι καλλιεργητές φυτών απλά είναι ένα θέμα που αφορά τις πολυεθνικές. Δεν είναι όμως αλήθεια αυτό γιατί έχουμε πάρα πολλούς μικρούς παραγωγούς, ερευνητικούς φορείς που ασχολούνται με την καλλιέργεια και ακριβώς αυτοί οι μικροί χρειάζονται την ανεμπόδιστη πρόσβαση στο γενετικό υλικό. Ε, ως εκ τούτου πρέπει το γενετικό υλικό που υπάρχει υπάρχει ανά τον κόσμο να προσφέρεται έτσι ώστε οι καλλιεργητές να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ε, ποικιλίε αυτές δίθεν να τις κατοχυρώνουμε, αυτό να το εμποδίσουμε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που διακομματικά συμφωνούμε όλοι από αυτού. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε η ζωή ε, και τα φυτά να μην πρέπει να κατοχυρώνονται ε, κυρίω ε, όσον αφορά την φυσική τους παραγωγή. Τώρα για τα γενετικά δροποποιημένα προϊόντα, εκεί έτσι κι ισχύουν ξεχωριστέ διαδικασίες και νομοθετικές διατάξεις. Ε, θα ήθελα λοιπόν να δώσω τώρα το λόγο στην Επιτροπή για να κλείσει τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, χαίρομαι που βρισκόμαστε όλοι σε αυτή την θέση. Συμφωνούμε όλοι μας και νομίζω ότι ήταν απόλυτα σαφές ευθύς εξ αρχής ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εκπέμψει το μήνυμα ότι τα φυτά τα οποία προκύπτουν από φυσικές διεργασίες δεν θα πρέπει απαραίτητα να κατοχυρώνονται. Ε, Πράγματι θα προσπαθήσω να συνεχίσω τη συζήτηση με το Γραφείο περιστεχνιών ε, να είμαστε ενεργοί, να επαναφέρουμε την νομική ασφάλεια, γιατί ξέρουμε ότι αυτή είναι πολύ σημαντική για τους ενδιαφερόμενους. Και βεβαίως ε, θα παρουσιάσουμε και τα συμφέροντα των καλλιεργητών, των πολιτών. Θα προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε και τον κοινό νου, τη λογική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, γιατί νομίζω ότι μας έδωσε το οδηγό βήμα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για το μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείνει λοιπόν η συζήτηση για το θέμα αυτό και πάμε στο επόμενο θέμα της ε, ημερήσιας διάταξης. Ε, είναι μια δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής, είπα της εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, πρόκειται για την κατάσταση στο Χονγκ Κόνγκ. Όμως πριν από τη συζήτηση, ε, σας παρακαλώ να βάλετε ακουστικά σας όλοι, να με ακούσετε γιατί θα ήθελα να πω κάτι σχετικά με την Ολομέλεια αυτής της εβδομάδας. Θα δοκιμάσουμε ένα νέο σύστημα που αφορά στη διαδικασία του Catch the Eye και τις μπλε κάρτες. Θα δοκιμάσουμε λοιπόν ένα σύστημα που θα είναι ε, να μας ε, ενημερώνεται ηλεκτρονικά όλοι οι ευρωβουλευτές έχουν ενημερωθεί με email, με ηλεκτρονικό μήνυμα. Αν θέλετε να λάβετε το λόγο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική σας κάρτα. Και γι' αυτό σας ερωτώ το εξής. Αν θέλετε να λάβετε το λόγο στη διαδικασία Catch the Eye ή να ρωτήσετε κάτι με το σύστημα της μπλε κάρτας, μπορείτε να το κάνετε με την ηλεκτρονική σας κάρτα, να την έχετε μαζί σας. Αυτή βέβαια θα είναι μια δοκιμαστική περίοδος. Ε, προφανώς και μπορείτε αν θέλετε να σηκώνετε το χέρι σας, αλλά θα θέλαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και στο μέλλον να χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και μόνο το ηλεκτρονικό σύστημα. Λοιπόν, θα το δοκιμάσουμε το ηλεκτρονικό σύστημα κατά την επόμενη συζήτηση που σημαίνει ότι αν θέλετε να λάβετε λόγο στο πλαίσιο της διαδικασίας Catch the Eye ή μέσω μιας μπλε κάρτας να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική σας κάρτα. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μπιανκόφσκα για να μας μιλήσει για την κατάσταση στο Hong Kong. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Να σας κάνω μια αρχική παρουσίαση της κατάστασης στο Hong Kong εξ ονόματος της ΥΠΑ της εκπροσώπου της κυρίας Μογκερίνη. Τον τελευταίο μήνα ο λαό Χονγκ Κόγκ έχει ασκήσει το θεμελιώδες ε, δικαίωμα του για ειρηνική διαδήλωση, για την αυτονομία και τα δικαιώματα της ελεύθερη έκφρασης και του συνέρχεστε. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ζητήσαμε από όλε τι πλευρές να αποκηρύξουν την βία και να αποκλιμακώσουν την κατάσταση. Υπ' αυτήν την έννοια, η απόσυρση του νόμου περί έκδοσης στην υπηρετική Κίνα είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Ο λαός του Χονγκ κατέβηκε στους δρόμους μαζικότατα και έδειξε την αποφασιστικότητά του. 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους στις 18 Αυγούστου. Τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η κατάσταση κλιμακώθηκε, είχαμε σοβαρά κρούσματα βίας από την Τριάδα, την Κινέζικη Μαφία, επιθέσεις ε, παρισταμένων, αναφορές για υπερβολική βία από την αστυνομία, κοκτέιλ μολότοφ ε, και βανδαλισμούς. Όλη αυτή η βία είναι απαράδεκτη. Παρ' όλα αυτά, οι διαμαρτυρίες ήταν κατά κύριο λόγο ειρηνικές και συνεχίζουν να έχουν τη στήριξη του λαού του Χονγκ Κόνγκ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στηρίξει την αρχή «Μία χώρα, δύο συστήματα» μια αρχή η οποία ε, υπάρχει στον θεμελιώδη νόμο του Χονγκ Κονγκ και είναι και διεθνής υποχρέωση της ε, Κίνας ε, με βάση και την σύμβαση με την Μεγάλη Βρετανία την οποία έχει κυρώσει το, η Εθνοσυνέλευση της Κίνας και η οποία εγγυάται τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του λαού του Χονγκ Κονγκ. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και για την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων στο Χονγκ που παραμένει ένα πάρα πολύ σημαντικό οικονομικό κέντρο και κόμβος μεταφορών. Η αρχή μια χώρα, δύο συστήματα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να συνεχίσει το Χονγκ να παίζει τον στρατηγικό οικονομικό του ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την διατήρηση των ελευθεριών των πολιτών του Χονγκ και τον υψηλό βαθμό αυτονομίας αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την ευημερία του Χονγκ Κόνγκ, αλλά επίση και τη υπηρετική κίνα. Ο σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τι ελευθερίε και την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Επίση έχουν κέρια σημασία για την ανάπτυξη του Χονγκ Κόνγκ και για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων εκεί. Και θα πρέπει βεβαίω ε, να τηρηθεί ο θεμελιώδη νόμο και οι διεθνεί δεσμεύσει τη Κίνα. Στι 18 Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζήτησε αυτά τα θέματα σε κατεπίγουσα συζήτηση και ενέκρινε ένα ψήφισμα. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράσης ε, δημοσίευσε τρεις δηλώσεις και στις 17 ε, Αυγούστου η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος έκανε μια επίσημη δήλωση που ενέκριναν όλα τα κρατημέλη, η οποία απέριπτε την βία και καλούσε σε διάλογο όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο συζήτησε την κατάσταση με πολλούς διεθνείς εταίρους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και εξέδωσε μια κοινή δήλωση με το Υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά. Το Hong Kong ε, συζητήθηκε και από τους Υπουργούς Εξωτερικών στο Ελσίνκι στο τέλος Αυγούστου έκτοτε. Η Κάρι Λαμ, η διοικητή του Χονγκ Κόνγκ, ανακοίνωσε στι 4 Σεπτεμβρίου πω ο νόμο ο οποίο θα επέτρεπε έκδοση στην υπηρετική Κίνα θα αποσυρθεί. Η καλοδεχόμενη αυτή κίνηση των ε, αρχών δίνει ένα περιθώριο για να μεταβούμε σε μια ειρηνική επίλυση της κατάστασης η οποία παραμένει τεταμένη. Μας ανησυχεί η βία που υπάρχει ακόμα και θεωρούμε ότι όλες οι πλευρές ε, θα πρέπει να απέχουν από την βία και να αναζητήσουν λύση μέσω ενός πραγματικού και επικοδομητικού διαλόγου. Για να συμβεί αυτό πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνουν τολμηρά βήματα για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη δεύτερον. Βλέπουμε ότι η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των επενδυτών επίσης επηρεάζεται. Το Hong Kong είναι μια γέφυρα μεταξύ της κινέζικης και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Έχουμε πολλές επιχειρήσεις που παίζουν θετικό ρόλο και στον διάλογο για να βρεθεί μια μόνιμη και διαρκής λύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην κυρία Σόιντροβα. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Όπως είπε η Επίτροπος, η κατάσταση στο Χονγκ δεν είναι απλή και συνεχίζονται τα προβλήματα εκεί. Όταν εγώ είδα τους χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους, στις διαδηλώσεις υπέρ της ειρήνης, αυτό μου θύμισε ιστορία 30 χρόνια πίσω στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Αλλά τότε η δικτατορία πάει, δεν υπάρχει πια. Ενώ εδώ βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση προσπάθειες που κάνει η Κίνα να επανισάγει διάφορα στοιχεία δικτατορίας. Έπειτα σκέφτομαι και τις χριστιανικές αξίες. Οι διαδηλωτές φώναζαν αλληλούια και προσπαθούσαν να αποφύγουν την σύγκρουση και τη βία. Αξίζουν τη στήριξή μας λοιπόν. Υπάρχουν ε, άνθρωποι οι οποίοι εκεί φοβούνται να χάσουν τα δικαιώματά τους και για εβδομάδες διαδήλωναν και κατάφεραν να κάνουν ε, τις αρχές να ανακαλέσουν τα επίμαχα νομοσχέδια. Όμως συνεχίσουν τους διαδηλώσεις γιατί ζητούν και άλλα. Θυμάμαι ότι είχαμε και τις απαγωγές των ε, πέντε ε, βιβλιο... υπαλλήλων σε βιβλιοπολία βιβλιοπολών ε, απήχθησαν εξαφανίστηκαν ορισμένοι, έχουν χαθεί τα ίχνη τους, οπότε διαδηλώνουν για την απελευθέρωσή τους οι άνθρωποι στο Χοκόγκ. Η Κίνα πρέπει να γνωρίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν προϋπόθεση για οποιοδήποτε εμπορική συνεργασία. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ρένα έχει τώρα το λόγο εκ των Σοσιαλδημοκρατών. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται στο Χοκόγκ παρόλο που οι, Κινες, αρχές του Χονγκ Κόγκ απέσυραν το νομοσχέδιο το σχετικό με τις εκδόσεις. Όμως αυτό καλύπτει μία μόνο διεκδίκηση των ε, ακτιβιστών και διαδηλωτών εκεί. Εκατομμύρια άνθρωποι εδώ και τρεις μήνες κατεβαίνουν στους δρόμους και αξίζουν τη στήριξή μας, ε, την ε, στήριξη της Ευρώπης, το δικαίωμα στη διαδήλωση, το δικαίωμα σε ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αυτά τα πράγματα πρέπει να ισχύουν αν θέλουμε να έχουμε ένα δημοκρατικό σύστημα. Αυτά που κάνει η Κίνα σε βάρος των διαδηλωτών του Χονγκ Κόνγκ είναι δυσανάλογα, υπερβολική βία, κάτι το οποίο παραβιάζει τι διεθνεί συμφωνίε και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και εμεί δεν μπορούμε να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίζει πάντα όσου υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτο δικαίου ειρηνικά. Φαίνεται όμω ότι κάποιε χώρε μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πουλήσει τεχνολογικό υλικό το οποίο οδηγεί σε καταστολή σε βάρο των διαδηλωτών, κυρίω υλικό παρακολούθηση αλλά και δακρυγόνα. Το άλλο ψηφισμό μα το 2019 ζητούσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα μηχανισμό ελέγχου των εξαγωγών προ την Κίνα, ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και η τεχνολογία του να μην αποτελούν συνένοχο τελικά τέτοιων παραβιάσεων. Ένα μήνα αργότερα που βρισκόμαστε. Οι τελευταίες ακροάσεις που είχαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μα ε, έδειξαν μαρτυρίε από τους ακτιβιστές που φοβούνται όχι μόνο μην χάσουν την ελευθερία τους αλλά και την ίδια τη ζωή τους. Ποιο είναι το μήνυμα που μπορούμε να του στείλουμε λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε κυρία έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ, από το Renew. Χωρίς μικρόφωνο, κύριε Βάτμαντς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πέντε εβδομάδες. Τόσο καιρό κρατάνε τώρα οι μαζικές διαδηλώσεις στο Χονγκ Κόνγκ. Με εκατομμύρια ανθρώπους, εκατομμύρια διαδηλωτές που τολμούν να κατέβουν στους δρόμους και να ζητήσουν δημοκρατία και περισσότερο σεβασμό στα δικαιώματά τους, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι πριν από μένα. Και εμείς τι απαντάμε. Η απάντηση που παίρνουν είναι δακρυγόνα, είναι πλαστικές σφαίρες, υπερβολική βία από πλευράς της αστυνομίας και εκφοβισμός, ε, συλλήψεις, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν είναι δυνατόν εμείς να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και αδιάφοροι. Μία χώρα, δύο συστήματα. Είναι καλό που αποσέρθηκε το νομοσχέδιο, αλλά οι διαδηλωτές ζητούν περισσότερα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί και το Χοκόγκο να μην ακολουθήσει δρόμο που αποκλίνει από τη δημοκρατία δεν πρόκειται για μια εσωτερική πια υπόθεση τη στιγμή που πρόκειται για τα οικουμενικά δικαιώματα τα οποία παραβιάζονται εκεί. Οπότε ρωτάω συγκεκριμένα την Επιτροπή πώς πάει ο διάλογος με την Κίνα, πόσο θα ξεκαθαρίσετε ότι εμείς θέλουμε να έχουν ελευθερία οι διαδηλωτές και πώς θα ζητήσετε να υπάρχει πραγματική ανεξαρτησία και όχι υπερβολική βία. Θα πρέπει ειρηνικά να μπορούν οι διαδηλωτέ να διαδηλώνουν και να μην φοβούνται για τη ζωή του. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Επόμενος ο κύριος επόμενο ομιλητή είναι ο κύριο Μπιτικόφα. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από δύο εβδομάδε επισκέφτηκα το Χονγκ Κονγκ και μίλησα με διάφορου ε, άμεσα ενδιαφερόμενου και επέστρεψα πισμένος ακόμα περισσότερο ότι το Κοινοβούλιο έκανε το σωστό όταν πριν από το καλοκαίρι δήλωσε ότι εμεί στηρίζουμε το λαό του Χονγκ Κονγκ. Το κίνημα για την δημοκρατία και την ειρήνη στο Χονγκ Κονγκ εξακολουθεί να υπάρχει και εξακολουθεί να αξίζει την αμέριστη υποστήριξή μας. Μία χώρα, δύο συστήματα. Αυτό δεν πρέπει να υπονομεύεται με παρεμβάσεις του Πεκίνου ή επιβάλλοντας αποφάσεις για κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ε, δεν αρκεί να αποσυρθεί αυτός ο νόμος περί έκδοσης υπόπτων στην Κίνα. Οι άνθρωποι θέλουν περισσότερα θέλουν μια ανεξάρτητη έρευνα για τη βία που ασκείται κυρίως από την αστυνομία και θέλουν και καθολικό δικαίωμα ψήφου το οποίο τους το υποσχέθηκαν πριν από 22 χρόνια στο Σύνταγμα αλλά αυτή η υπόσχεση δεν έχει τηρηθεί. Το Πεκίνο πρέπει να τηρήσει αυτή την υπόσχεσή του. Εμείς ως πράσινοι στηρίζουμε αυτόν τον αγώνα για το καθολικό δικαίωμα ψήφου στο Χονγκ Κονγκ. Πρέπει να νικήσει η δημοκρατία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Ριβιέρ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι δραστήριο προκειμένου να σέβεται η Κίνα τη δημοκρατία. Πολύ καλό βέβαια, η επιλογή των λαών ε, προέχει και δεν πρέπει να υπάρχει ε, βία. Το να κοιτάμε τι γίνεται στην Κίνα είναι καλό, το να κοιτάμε τι γίνεται και στην Ευρώπη είναι ακόμα καλύτερα. Εδώ το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε κυρίαρχα να αποχωρήσει και εμείς δεν το αφήνουμε. Στην Ιταλία πάλι ε, παραφύσει η διαδικασία για να αποφύγουμε αυτά τα οποία επιθυμούν οι Ιταλοί. Και στη Γαλλία ε, στηρίζεται ο πρόεδρος από ένα κοινοβούλιο το οποίο δεν ε, είναι πια όπως ήταν όταν το στήριξε. Είναι όλα αυτά πρόσφατα παραδείγματα. Εμείς πρέπει να καταδικάζουμε αυτές τις πρακτικές. Αν δεν το κάνουμε, είμαστε αναξιόπιστοι αν συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο, απομακρυνόμαστε ακόμα περισσότερο από τους λαούς και έτσι ακριβώς πεθαίνει η δημοκρατία. Ευχαριστούμε κυρία Φωτίγκα, Άννα Φωτίγκα, εκ μέρους του ECR. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εμείς ε, στηρίζουμε τον λαό του Hong Kong. Αυτή είναι η απαρέγκλητη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τότε που πρώτο ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες και εμφανίστηκαν οι πρώτες ε, διαφωνίες. Οι πολίτες του Χονγκ Κόνγκ επιθυμούν να αποσυρθεί ο νόμος περί εκδόσεως υπόπτων. Τώρα όμως όλα τα κόμμα θα πρέπει να σεβαστούν ε, την δήλωση του 1984 και κυρίως το Πεκίνο δεν θα πρέπει να προσπαθεί να παρεμβαίνει, δεν θα πρέπει να προκαλεί. Όπως σας είπα, εμείς εξακολουθούμε να στηρίζουμε το λαό του Χονγκ Κόνγκ. Ευχαριστούμε πολύ. από την Είναι η πέμπτη εβδομάδα από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις στο Χονγκ Κόνγκ, 15η εβδομάδα. Και πού βρισκόμαστε σήμερα βία. Είδαμε και χτες νέες σκηνές βίας, όπου η αστυνομία ε, με δακρυγόνα και με κανόνια νερού επιτίθεται κατά των διαδηλωτών. Εμεί θέλουμε να γίνεται σεβαστό, γιατί είναι θεμελιώδε το δικαίωμα στη διαδήλωση και να γίνεται σεβαστό παντού στον κόσμο και στο Χονγκ Κόνγκ. Πώ αλλιώ. Οπότε εμεί συζητάμε να ερευνηθούν οι δράσει τη αστυνομία, να απελευθερωθούν οι ειρηνικοί διαδηλωτέ. Τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά και αδιέρετα. συνεπώ θέλουμε να καταδικάσουμε εδώ τη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν παρακολουθούν τι γίνεται σε άλλες ε, χώρες, αλλά δεν κοιτάει τι γίνεται μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τελικά οι διάφορες χώρες μέλη έχουν μεγάλες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επιτέλους να αποκτήσει ένα στρατηγική σημασία σε σχέδιο όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Κίνα. Θέλουμε διάλογο, θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις συνομιλίες που έχει με την Κίνα να φροντίσει να σεβόμαστε παντού τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί αυτό είναι το μόνο που μπορεί να οδηγήσει σε κάτι θετικό γεωπολιτικά στον 21ο αιώνα. Ευχαριστούμε. Τενό τώρα. Παρακαλώ. Μη γραμμένος. Με το μικροφωνό σας παρακαλώ.

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είτε πιστεύουμε στη δημοκρατία και την ελευθερία, είτε δεν πιστεύουμε. Γιατί αν δεν πιστεύουμε, τότε αυτή η συζήτηση είναι περιττή. Εάν όμως πιστεύουμε, τότε είναι μια αρχή που ξεπερνάει τα εθνικά σύνορα και μάλιστα ξεπερνάει τα ευρωπαϊκά σύνορα. Είναι μια οικουμενική αρχή. Βία από το κράτος εις βάρος των ε, διαδηλωτών είναι απαράδεκτο. Η βία από τους διαδηλωτές και αυτή δεν είναι κάτι αυτονόητο. Όμως ε, το θέμα είναι πάρα πολύ απλό σε τελική ανάλυση. Ποιος θα αποφασίσει ποιος ε, κυβερνάει το Χονγκ Κονγκ. Ξεχάστε τον, την πολιτική του 19ου αιώνα, γιατί αυτή εξακολουθεί να επηρεάζει τον 21ο αιώνα. Η απάντηση πρέπει να είναι ότι οι άνθρωποι, ο λαός του Χονγκ Κόνγκ έχει το ίδιο δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, όπως και όλα τα υπόλοιπα ανθρώπινα όντα. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, κυρία Σάντος από τους Σοσιαλδημοκράτες, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ο αγώνας ε, των ε, τελευταίων μηνών και οι, οι ειρηνικέ διαδηλώσει στο Χονγκ Κονγκ. Αυτό είναι ένα αγώνα για την ελευθερία τη έκφραση γνώμη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Η, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί απλά να παρακολουθεί δρανείς ε, πρέπει να δραστηριοποιηθεί, να κάνει κάτι ε, απέναντι στις ε, τοπικές και τις κινέζικες αρχές. Δεν πρέπει να κλιμακωθεί περαιτέρω η βία εις βάρος των διαδηλωτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για να παρεμποδίσει τη βία και να πει με απόλυτη σαφία στις αρχές της Κίνας ότι η βία εις βάρος των διαδηλωτών δεν μπορεί να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει υπάρξει μια ειρηνική λύση να διευθετηθεί ειρηνικά το θέμα. Εμείς χαιρετίζουμε αυτά που είπαν οι επικεφαλής των διαδηλώσεων, ότι οι διαδηλώσεις θα παραμείνουν ειρηνικέ και πρέπει να πούμε στην κινέζικη κυβέρνηση ότι δεν αρκεί να προβαίνει σε, προθέσεις, σε δηλώσεις προθέσεων. Πρέπει να ε, γίνουν συγκεκριμένα πράγματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του συνέρχεστε. Ο κύριος Γκέτα από το Ρινιού. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θάρρος, αποφασιστικότητα και αγώνας για τη δημοκρατία. Αυτά χαρακτηρίζουν ε, τις διαδηλώσεις στο Χονγκ Κόνγκ. Δεν ε, αντέδρασαν οι κινέζικες αρχές ε, στην Τιαναμέν, τώρα απέσυραν το νομοσχέδιό τους. Πρέπει λοιπόν να χειροκροτήσουμε τους διαδηλωτέ στο Χονγκ Κόνγκ και να χαρούμε για την νίκη τους, γιατί κάθε υποχώρηση από ένα καθεστώς που τυρανά τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα βήμα προς τη δημοκρατία για όλους. Δεν φτάνει. Πρέπει να στηρίξουμε τον ε, αγώνα προκειμένου η Κίνα να γίνει πιο δημοκρατική δεδομένου ότι είναι εμπορικό μα εταίρο. Έχουμε την ηθική υποχρέωση. Έχουμε επίση την υποχρέωση, επειδή μπορούμε να το κάνουμε και μπορούμε να το κάνουμε, γιατί σε αυτήν την δελκιστίδα με τον Τραμπ οι κινέζικε αρχές δεν μπορούν να επιτρέψουν στον εαυτό τους να απομακρυνθούν από την Ευρώπη. τι χρειάζονται. Και εμείς, ευρωβουλευτές, μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο το οποίο είναι ισχυρό, ανεξάρτητο και μπορεί να αντιμετωπίσει ένα καθεστώς που έγινε η πιο, σύγχρο... το πιο σύγχρονη, η πιο μεγάλη και η πιο περίπλοκη δικτατορία. Μπορούμε αυτό να το πούμε πολύ σύντομα, ελπίζω, και ελπίζω να το ζητήσουν αυτό όλες οι πολιτικές ομάδες δίνοντας το βραβείο Ζαχάροφ σε έναν αντιφρονούντα Κινέζο, στον κύριο Λακωτή, ο οποίος είναι ακτιβιστής, είναι φυλακισμένος από τους Ιγούρους και αποτελεί μια μεγάλη προσωπικότητα. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ρόβετ από τους Πράσινους. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Επί Βρετανικής Αυτοκρατορίας η Βρετανία θεωρούσε ότι είναι η μητέρα των ελεύθερων ανθρώπων. Πού κατέληξε όμως αυτή η αυτοκρατορία. Χτες οι διαδηλωτές κρατούσαν βρετανικές σημαίες και διαδήλωναν έξω από το βρετανικό προξενείο στο Χονγκ Κονγκ και δικαίως γιατί η Βρετανία έχει καθήκον να υπερασπιστεί την ελευθερία τους από την ε, κοινή δήλωση του 1984. Η πρόσφατη απάντηση από την Βρετανίδα πρέσβυρα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων μοιάζει πάρα πολύ ήρεμη. Γιατί η απόσυρση του νομοθεσίου δεν μπορεί να επιλύσει τις ανησυχίες. Εάν η ίδια η Βρετανία δεν αμφισβητήσει την Κίνα, τότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί να είμαστε εμεί αυτοί οι οποίοι θα υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρί σύνορα και να υπερασπιστούμε το δικαίωμα του εκλέγην των ανθρώπων του Χονγκ γίνουμε εμεί η μητέρα των ελεύθερων ανθρώπων και αυτό να μην γίνει με το να οικοδομήσουμε μια αυτοκρατορία, αλλά με το να αμφισβητήσουμε τον υπεριαλισμό. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπονφρίσκο κατόπιν από το ID. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης μας ενώνουν όλους στις απαραβίαστες αρχές του κατζουκαίου και της δημοκρατίας. Βλέπουμε από την άλλη πως προσπαθεί η Κίνα να αγνοήσει τους πάντες και τα Ηνωμένα Έθνη αγνοώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεωρώντας ότι το κράτος έχει πρώτο καθεδρία ε, όταν, ακόμα και όταν διαμαρτύρονται οι άνθρωποι για τις ελευθερίες τους. Ε, η Δε Κέρι Λάμ λέει πως οι διαδηλωτές είναι μια μικρή μειονότητα βιαίων διαδηλωτών που δεν έχουν ανταπόκριση στην κοινωνία, οι οποίοι προκαλούν χάος και αναταρχές χειρότερες και από την οικονομική κρίση. Πρόκειται για κάτι λάθος και αντιδημοκρατικό. Η δράση της αστυνομίας και των αρχών του Χονγκ Κονγκ που βρίσκονται υπό τον αυστηρό έλεγχο των κινέζικων αρχών είναι εν ολίγης ε, απάνθρωπες. Σε όλα αυτά θα πρέπει να απαντήσουμε χωρίς φόβο με μια ξεκάθαρη πολιτική δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα του καθεστώτος του Χονγκ Κονγκ και θα καθορίζει τις μελλοντικές μας σχέσεις με την Κίνα έξω ονόματος του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Μίσλαβ Κουλάκουτσης έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα στο κοινοβούλιο αυτό να συζητάμε τις αρχές αυτές περί κράτους δικαίου και δημοκρατία σε τρίτες χώρες, αλλά θα ήθελα να σκεφτείτε το θέμα του κράτους δικαίου στην Κροατία όπου ένα 94% των ανθρώπων σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πιστεύουν ότι ε, το καθεστώ είναι διεφθαρμένο. 76% των Κροατών θεωρούν ότι έχουμε ε, κακή έως πολύ κακή δικαιοσύνη. Δυστυχώς η παρακολούθηση την οποία είχαμε ε, μέχρι την στιγμή της ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επαρκούσε. Πολύ απλά Έχω εργαστεί στην ε, κροατική δικαιοσύνη, ήμουν δικαστής επί 21 έτη, 9 έτη στα εμπορικά δικαστήρια. Ε, Εκπήρας λοιπόν λέω πως είναι εξόχως διεφθαρμένη η κροατική κοινωνία και πρώτα απ' όλα πρέπει να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εμπλακούν, πρέπει να δούμε τα ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και την διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα έχουμε δικαίωμα να κάνουμε μαθήματα και σε άλλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Νίνα Γκίλ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους του Χονγκ Κονγκ για να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά. Η αντίδραση ήταν κτηνοδία, πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα. Πολλοί τραυματίστηκαν. Το μόνο τους έγκλημα ήταν ότι ζητούσαν δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Οι αξίες τους είναι οι αξίες μας και πραγματικά κινδυνεύουν, ε, κινδυνεύει η ζωή τους. Η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση πρέπει να εξετάσουν όλα τα μέτρα για να στηρίξουν τους ανθρώπους του Χονγκ Κονγκ που ε, προσβλέπουν ε, από εμάς να τους στηρίξουμε. Έχουμε ένα μοχλό πίεση. Παραδείγματος χάρη Μήπως να αποσύρουμε το καθεστώς του Χονγκ Κονγκ ε, για την ισοδυναμία τρίτης χώρας ε, στα χρηματοπιστωτικά. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους Κινέζους ε, τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την αρχή «Μια χώρα, δύο συστήματα» στην οποία περιλαμβάνεται η προστασία αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων, την οποία έχουν συνυπογράψει τη στιγμή της μεταβίβασης ε, κυριαρχίας από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1997. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μια ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους του Χονγκ Κονγκ. Πρέπει να τους προστατεύσουμε ε, να βρουν καταφύγιο στην Ευρώπη εάν συνεχίσουν να αποτελούν στόχο διώξεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπέργκ από το ID. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα μιλάμε για το Χονγκ Κονγκ και νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι αυτή η αρχή, μία χώρα, δύο ε, συστήματα, ε, την αρχή αυτή τη στηρίζουμε για τη μορφή διακυβέρνηση ε, του Χονγκ Κονγκ. Όλοι γνωρίζουμε αυτά που είπε, είπατε εκπρόσωπο και ο Καναδό, οι οποίοι κάλεσαν τι αρχέ τη Κίνα να σέβονται το Χονγκ Κονγκ, να εφαρμόζουν το Σύνταγμα και του νόμου και να έχουν υπόψη του ότι μόνο ένα ουσιαστικό διάλογο μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα πρόβλημα. Τα αιτήματα, το να υπάρχει μια ανεξάρτητη έρευνα για την άσκηση βία από πλευρά αστυνομία, κάτι το οποίο έχει προτείνει τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτή είναι μια δυνατότητα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η κινέζικη κυβέρνηση δεν πρέπει να εγκλωβίζεται όλο και περισσότερο στην επιθετικότητα, να ασχοληθεί με τα προβλήματα που επισημαίνονται από τη διεθνή κοινότητα, μια στρατηγική στρατηγική διπλωματία που θα επιτρέψει ε, στην κινέζικη πλευρά να διαφυλάξει το κύρος της και έτσι ίσως επιτύχουμε τα αποτελέσματα τα οποία διεκδικούν οι πολίτες του Χονγκ Κονγκ. Να μπορέσουμε να παρεμποδίσουμε ενδεχόμενο καταστροφής όπως έγινε στην πλατεία Τιένα Μεν. Να μην υπάρξει κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος ε, Πίκουλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πολύ. Πάρα πολύ. Πέρασαν 100 μέρες από όταν ξεκινήσαν οι διαδηλώσεις στο Χονγκ Κόνγκ. Είναι η μεγαλύτερη κρίση που έχει υπάρξει στις ε, σχέσεις ε, του Χονγκ Κόνγκ με την υπηρετική Κίνα από το 1987. Παρά το ότι το σχετικό νομοσχέδιο του μεταξύ αποσύρθηκε, οι διαδηλωτές συνεχίζουν ε, με τα αιτήματά τους και διαδηλώνουν με μεγαλύτερη ένταση. Θέλουν περισσότερες δημοκρατικές ελευθερίες και ζητούν την απελευθέρωση των κρατουμένων διαδηλωτών. Η κλιμάκωση της βίας στους δρόμους του Χονγκ Κόνγκ είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Η δικαιοσύνη του Χονγκ Κόνγκ θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Και η Κίνα όταν ε, εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις της, αλλά και παγκοσμίω ε, έχει επιλέξει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει υπογράψει σχετικές ε, συμφωνίες. Οπότε υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να σταματήσει η βία και να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ των διαφόρων μέρων. Αυτή είναι η μόνη εγγύηση για να υλοποιηθούν αυτές οι δεσμεύσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη. Ε, Θέλετε να κάνετε μπλε κάρτα. Θέλετε να κάνετε ερώτηση με την μπλε κάρτα. Μπλε κάρτα. Κύριε Πίκουλο, δέχεστε μία ερώτηση από τον συνάδελφο, ναι. Έχετε 30 δευτερόλεπτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε συνάδελφε, περιγράψατε πάρα πολύ καλά την κατάσταση στο Χονγκ Kong, κάνατε και μια σύντομη ιστορική αναδρομή όμως, ε, δεδομένου του ζητήματος και τη σημασία της Κίνας ως εμπορικού εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε πόσο μεγάλες είναι και οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κροατία Πώς βλέπετε την ε, σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας ε, δεδομένων όλων των προβλημάτων που αναφέρατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μπορέσουμε όλοι να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό από κοινού για το πώς ε, δηλαδή θα έχουμε σχέσεις με χώρες όπου οι δημοκρατικές αρχές ε, δεν ε, τηρούνται στο έπακρο. Θα επικρατήσει το κίνητρο του κέρδους ή οι αιώνιες αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω να επιτύχουμε την σωστή ισορροπία και να βελτιωθεί η κατάσταση ε, στις χώρες αυτές ε, όπου δεν γίνονται σεβαστές αυτές οι αρχές. Ε, πρέπει να επιλέξουμε προτεραιότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα περνάμε στη διαδικασία και Πέντε βουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο. Τρεις το ζήτησαν ηλεκτρονικά. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουν όλοι τις ε, κάρτες τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος είναι ο πρώτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, εγώ είμαι ένας από εκείνους ε, που ζήτησα το λόγο ηλεκτρονικά, για να το ξέρετε. Κατά τη δική μου άποψη θα πρέπει να στηρίξουμε τις ειρηνικές διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ. Ε, Κατό ημέρες ε, ταρακούνησαν το Χονγκ Κονγκ και ταρακούνησαν και την εμπιστοσύνη μας στο διάλογο ανάμεσα στις άμεσα ενδιαφερόμενες πλευρές. Οι διαδηλωτές διεκδικούν το δικαίωμα αυτονομίας, το δικαίωμα του συνέρχεστε. Αυτά έχουν κατοχυρωθεί το Σύνταγμα του Χονγκ Κονγκ. Χαίρομαι πάρα πολύ ε, που έχει αποσυρθεί ο νόμος περί εκδόσεως υπόπτων, αλλά νομίζω ότι ο ρόλος μας είναι να στηρίξουμε τους διαδηλωτές στο Χονγκ Κονγκ. Έχει διαχυθεί η βία, Είναι επικίνδυνο αυτό και νομίζω πραγματικά πρέπει να στηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται κάποιο τίμημα. Οφείλουμε να επαναφέρουμε το θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων οποτεδήποτε αντιπροσωπεί μας πάνε στην Κίνα. ποιο άλλο θα το κάνει, το κάνουμε εμείς. Και να μην διαπραγματευτούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα με οποιοδήποτε οικονομικό όφελος. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος, μαζί και με άλλους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ε, μαζί με ακτιβιστές. Εγώ υπέγραψα μια ανοιχτή επιστολή εκφράζοντας την αλληλεγγύη μου για να συνεχιστεί ο αγώνας στο Χόγκ. Εμείς στηρίζουμε την ε, αντίσταση των πολιτών στο Χονγκ Κόνγκ για την επίθεση που δέχονται στα δικαιώματά τους. Στηρίζουμε τα πέντε αιτήματα του κινήματος για να μην υπάρχει καταποίηση, να ληφθούν σοβαρά μέτρα για να αντιμετωπιστεί το αστυνομικό κράτος, να υπάρχει δημοκρατία και μια κυβέρνηση που θα εκλέγεται ε, μέσα από το καθολικό δικαίωμα ψήφου. Καλούμε το εργατικό κίνημα σε ολόκληρο τον κόσμο να οργανώσει την πολιτική και πρακτική αλληλεγγύη με το Χονγκ Κονγκ και στον αγώνα για τη δημοκρατία. Στηρίζουμε τις οργανώσεις ανεξάρτητων εργατών και φοιτητών που εμπλέκονται στον αγώνα ε, και επαναλαμβάνουμε ε, αυτό που έχουμε ήδη πει ότι πρέπει να στηρίξουμε το εργατικό κίνημα να υπάρξουν ε, και υπάρξει υποστήριξη για τον Τζέρεμι Ταμ Πρέπει λοιπόν να στηριχθούν όλοι οι εργαζόμενοι, κυρίως οι μετανάστες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όλα αυτά είναι άρρηκτα συνδεμένα με τον αγώνα των αδελφών μας ε, στο Χονγκ Κονγκ. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Wallace. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτή τη συζήτηση, γιατί πρέπει να πω ότι δεν ήταν όλες οι ε, διαμαρτύρες ειρηνικές. Υπάρχουν σχέσεις και με την άκρα δεξιά και υπάρχει και μεγάλη παραπληροφόρηση. Πολλά εκατομμύρια από τις Ηνωμένε Πολιτείες έχουν διοχετευτεί για να αλλάξει η δημοκρατία ε, υπάρχουν πολλοί που βρίσκονται μπλεγμένοι μέσα από το κίνημα και υπάρχουν και διαμαρτυρίες εκείνων που συναντήθηκαν με τους Αμερικανούς στο Χονγκ Κόνγκ. Οι νέοι που βρίσκονται στους δρόμους πράγματι νόμιμα διαδηλώνουν, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και σχέσεις με τον φιλελεύθερο κίνημα. Οι ολιγάρχες είναι εκείνοι που επικυριαρχούν. Η Κίνα βεβαίως και πρέπει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει όμως να εμπλέκεται στις υποθέσεις της Κίνας και ας μην έχουμε παροπίδες όσον αφορά αυτά τα θέματα. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά που συζητάμε για το Χονγκ Κόνγκ και για την υπεράσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Χονγκ Κόνγκ και όλα αυτά που είπαμε για την Κίνα. Λυπάμαι όμως ότι ξεχνάμε όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα κάτι άλλο και αυτό είναι ένα παράδοξο. Πριν από μία εβδομάδα μόνο η κυρία Μογκερίνη ήταν στην Κούβα. Όταν ακριβώς στο νησί της Κούβας υπήρξε κύμα καταστολής όσο λίγα στο παρελθόν. Και η κυρία Μογκερίνη εκεί μιλούσε για μια υπέροχη Κούβα, για μια Κούβα γέφυρα ε, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λατινική Αμερική. Μα είναι ένα σκάνδαλο αυτά που είπε στην Αβάνα η κυρία Μογκερίνη δείχνοντας συνενοχή με τη δικτατορία της Κούβας που 70 χρόνια τώρα καταπιέζει τους Κουβανούς και προσπαθεί να στηρίξει και, άλλες, ε, και άλλα τυρενικά καθεστώτα όπως εκείνο της ε, ε, Βενεζουέλας. Παρακαλώ να υπάρχει κάποια συνέπεια σε αυτά που λέμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ε, τελευταία στη διαδικασία του Κατσδιά είναι η κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ πολύ. Καταδικάζουμε και πρέπει να καταδικάζουμε τη βία οπουδήποτε και αν αυτή ασκείται. Αλλά εμείς είμαστε επιλεκτικοί στη συζήτηση αυτή που κάνουμε όσον αφορά τις διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ και με την κάλυψη που δίνεται στην Ευρώπη γι' αυτό. Γιατί εμφανίζεται ε, σαν κάτι πολύ απλό. Από τη μια έχουμε την αυταρχική Κίνα και από την άλλη μεριά έχουμε την δημοκρατία και τα δικαιώματα. Μα είναι τεράστια απλοποίηση αυτή που κάνουμε. Εδώ πέρα έχουμε εξωτερική ανάμιξη, διότι το κόστος ζωής στο Χονγκ Κόνγκ είναι τεράστιο και τα νίκια είναι πάρα πολύ ακριβά. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πάμε από την άλλη μεριά του κόσμου για να βρούμε αστυνομική καταστολή ή για να στηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ, στην Γαλλία, με τεράστια καταστολή, με εκατοντάδες ανθρώπους τραυματισμένους. Δεν λέμε όμως τίποτα για αυτή την καταστολή ή για τους πολιτικούς κρατούμενους στην Ισπανία που κανονικά είναι συνάδελφοί μας και θα έπρεπε να βρισκόντουσαν εδώ. Αλλά μιλάμε για την απελευθέρωση των κρατουμένων στο Χονγκ Κόνγκ. Ναι, συμφωνώ να το κάνουμε εκεί αλλά να το κάνουμε και στην Ευρώπη, στην Ισπανία, στη Γαλλία και όλες τις άλλες χώρες που κινδυνεύουν από τέτοιες πρακτικές. Ευχαριστούμε πολύ. Θα απαντήσει η Επίτροπος η κυρία Μπιακόφσκα. Παρακαλώ κύριε Μπιακόφσκα. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις παρεμβάσεις σας. Υπήρξε νομίζω ομοφωνία ε, λίγο πολύ για το πώς βλέπουμε ε, τι συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στο Χονγκ Κόνγκ. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν που έχετε το θέμα αυτό ψηλά στην ημερήσια διαταξή σας. Αναφέρθηκαν τα οικουμενικά δικαιώματα αρκετές φορές και σας υπενθυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στηρίζει το κράτος δικαίου τα οικουμενικά αυτά δικαιώματα και τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται παντού. Όλοι οι πολιτικοί εταίροι πρέπει να συμφωνούν και στο Χονγκ και στο Πεκίνο, πράγματι. Είχαμε και τον Ιούλιο ανταλλαγή απόψεων για το ίδιο θέμα και βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει στο Κονκόκ, για την ε, ευημερία εκεί. Και το πιο σημαντικό ενδιαφέρεται για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση από κοντά, τι γίνεται με τους ε, κατοίκους στο Χοκόγγ αλλά και με τους εταίρους που έχουν οικονομικά συμφέροντα εκεί. Θα έπρεπε να μην υπάρχουν πια εντάσεις εκεί γιατί αυτό θα είναι προς όφελος του Χοκόγγ των πολιτών του και όσων έχουν συμφέροντα σε αυτόν τον οικονομικό κόμβο. Η είπατη εκπρόσωπος, η κυρία Μογκερίνη, μου ζήτησε να εκφράσω την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι έχετε ψηλά στην ημερήσια διάταξη αυτό το θέμα και θα επαναλάβω ότι είμαστε υπέρ των οικουμενικών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θα συνεχίσουμε να τα στηρίζουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώνεται έτσι αυτή η συζήτηση. Και περνάμε στο τελευταίο θέμα για σήμερα στην ημερήσια διάταξη, που είναι οι παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού και πρώτος ο κύριος Σόκολ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, πριν από 30 περίπου χρόνια κατέρευσε το κομμουνιστικό καθεστώς ε, στο Βερολίνο προέκυψαν νέες προοπτικές για το σύνολο της Ευρώπης, κυρίως όμως για την Ανατολική Ευρώπη η διεύρυνση της Ευρώπης προς Ανατολάς, μπορούμε ενδεχομένως να πούμε ότι ήταν ε, επιτυχής. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια, η πολιτική συνοχή με βάση την αλληλεγγύη συνέβαλαν προς αυτή την κατεύθυνση σε μεγάλο βαθμό και έτσι λοιπόν κατέστη δυνατόν για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης να αλλάξουν και να μπορέσουν να ε, φτάσουν να πλησιάσουν τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Τώρα όμως δυστυχώς βρισκόμαστε και πάλι σε μια κατάσταση όπου διαφορές ε, ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση επιτείνονται. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το, αυτή την πολιτική. Πιστεύω ότι η πολιτική συνοχή είναι επιτυχημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμα και οι λιγότερο αναπτυγμένοι μπορούν να έχουν ικανοποιητικά κονδύλια, ίσες ευκαιρίες για να ανταγωνιστούν τους ε, πιο πλούσιους και νομίζω ότι αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Το να αρνούμε θα την ε, πολιτική ε, συνοχή. Σε αυτό νομίζω ότι επιτείνει την ανισότητα στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενος... Ο κύριος Αγγιλάρ, ευχαριστώ πολύ. Τώρα το καλοκαίρι το 2019, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, είχαμε τεράστιες πυρκαγιές στο νησί που γεννήθηκα και κατοικώ, τα Κανάρια. Το κόστος βέβαια είναι δυνατόν να εκτιμηθεί, αλλά η καταστροφή στα δάση είναι τεράστια. Πρόκειται για ένα ε, μέρος το οποίο είναι προστατευμένο. 10.000 εκτάρια κάηκαν, 6.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Και έχουμε πρόσφατα τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Αντίδρασης Προστασίας των Πολιτών ακριβώς για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπου έχει προσφέρει και η Ισπανία δύο αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα τελικά διατέθηκαν. Η Ισπανική κυβέρνηση κινητοποίησε τον μηχανισμό κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά η ευρωπαϊκή απάντηση πρέπει να είναι περισσότερο ευέλικτη, ώστε να μπορεί να κινητοποιηθεί και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης και πάνω απ' όλα, ήδη από το 2002 ζητάμε να υπάρξει αναθεώρηση έτσι ώστε να μπορεί έγκαιρα να δοθεί η έκτακτη αυτή βοήθεια από την Ευρώπη όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις καταστροφών όπως είχαμε το καλοκαίρι στην Ισπανία. Ευχαριστούμε πολύ. Γκροσέ από το Ρινιού. Ευχαριστώ πολύ. με εντατικές ε, προσπάθειες ε, της ε, Κομισιόν και της Επιτρόπου Διεύνησης για να ξεπεραστούν οι εντάσεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Και όμως έχουμε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Η θεσμική κρίση στην Βοσνία Ερζεγοβίνη και η πάρα πολύ ε, μεγάλη δασμή που επέβαλε η Σερβία στα προϊόντα κοσφοπεδίου ε, δεν βοηθούν καθόλου. Πρέπει να αναζητηθεί μία μόνιμη λύση καθώς ε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το μέλλον της περιοχής. Θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσει να βρει μια λύση αποδεκτή και από τις δύο πλευρές για να καταργηθούν αυτοί οι δασμοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αλφόνση έχει το λόγο. Εκ μέρους των Πρασίνων. Από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει έκθεση για τις γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ψηφίζοντας ε, το, την έκθεση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να γίνουν πράγματα, αλλά ελάχιστα έχουν να κάνει. Η πολυγλωσία δεν αναφέρεται σαν αποστολή σε κανέναν από τους αποσταλμένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όμως πρέπει να ευνοηθεί η τύχη των γλωσσών αυτών. Έξι χρόνια μετά η χάρτα για τις γλώσσες αυτές δεν έχει ακόμα εγκριθεί. Και ο αρμόδιος υπουργό, ο κύριος Μπλανκέρ της κυβέρνησης Μακρόν, έχει ξεκινήσει μια ανοιχτή πολιτική για τις γλώσσες μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε διάφορες χώρες. Αλλά ο σεβασμός της πολιτιστικής κληρονομιάς, της γλώσσας που είναι βασικό στοιχείο της κληρονομιάς αυτής είναι κάτι που πρέπει να προωθήσουμε. Ζητώ λοιπόν και από τη Γαλλία αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υλοποιήσει αυτό που έχουν ζητήσει από το 2013 οι ευρωβουλευτές, έτσι ώστε η ευρωπαϊκή κληρονομιά να μην κινδυνεύει από αφανισμό. Ευχαριστούμε. Κύριος Μπένιε, η κυρία Μπένιε από το Μπενιέ, Αγαπητοί συνάδελφοι, έκθεση της Ένωσης Γενιές του Μέλλοντος μιλάει για επικίνδυνη χρήση φυτοφαρμάκων στην Ευρώπη και η έκθεση αυτή υπογραμμίζει ότι η χρήση των φυτοφαρμάκων δεν λαμβάνει υπόψη την επιστημονική γνώση. Οι πολίτες και οι καταναλωτές αυτέ δυστυχώς μπερδεύονται Υπάρχει και σύγχυση γιατί υπάρχουν και αντιφατικές ε, μελέτες. Οπότε δεν μπορεί να ξέρει κανείς αν ε, τις έχουν ζητήσει τις διάφορε έρευνε, οι ε, του κλάδου ή όχι. Πρέπει να υπάρχει έρευνα ανεξάρτητη από κάθε οικονομικό συμφέρον για να μπορεί να καταλαβαίνει τι γίνεται ο και να είναι καλά ενημερωμένο. Μια τέτοια μελέτη πρέπει να είναι εκτενέστατη και να διευρύνει βέβαια το θέμα και στους ανδροκρινικούς διαταράκτες. Ευχαριστούμε από το ECR. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στις 2 ε, Ιανουαρίου 2019 άλλαξαν οι κανόνες για τη χορήγηση βίζας ε, στους υπήκοους ε, Λευκορωσίας. Τώρα μπορεί κάποιος να πάρει τουριστική βίζα. Αυτό μεταξύ άλλων οδήγησε στην αύξηση των αριθμ... του... στη μείωση, του αριθμού υπηκών ε, Λευκορωσίας που επισκέπτονταν την χώρα. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει ξανά η δυνατότητα είτε μια απλής διαδικασίας είτε κάποιο είδους βίζας που θα επιτρέπει το εμπόριο στις μεθοριακές περιοχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Overgaard. μετά από την ε, ψήφο 17,4 εκατομμυρίων Βρετανών για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είπαν πως ε, θα έπρεπε να μην είναι επιτυχές στο Brexit. Μήπως γιατί εάν έφευγε η Βρετανία θα ακολουθούσαν κι άλλο. Εάν ρωτούσαμε τους πολίτες Ευρώπης εάν ήθελαν συμφωνία ελευθερία εμπορίου ή ένα υπερκράτος θα ήταν υπέρ ε, μιας εμπορικής συμφωνίας. Αλλά γιατί να ακούσουμε τους λαούς τη δημοκρατία την ακούμε μόνο όταν ε, λέει αυτό που θέμε. Κοιτάξτε, ο πατέρας μου στο δεύτερο παγκόσμιο ήταν αντάρτης ε, επί τέσσερα χρόνια και άκουγε τον ε, Μόντι, τον Άγγλο στρατηγό, όταν μπήκε στην χώρα μας και εγώ είχα κατεβεί σε διαδηλώσεις κατά της συνθήκης του Μάστριχτ. Οπότε δεν θα σκύψω το κεφάλι σε κανέναν. Πιστεύω στην ελευθερία, τη δημοκρατία και την αυτοδιάθεση. Θα ήθελα λοιπόν να σα παρακαλέσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ανταποκριθεί στον αρχικό του σκοπό να είναι ο δημοκρατικός φάρος τη Ευρωπαϊκή Ένωση να σεβαστεί τον Βρετανικό λαό, αλλά και αυτού που είναι πέρα από την φούσκα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα... Τον λόγο έχει ο κύριος Πόλτσακ για το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο ένα λεπτό αυτό θα ήθελα να αναφέρω μια τεράστια σύγκρουση συμφερόντων του Τσέχου Πρωθυπουργού με το ελεγκτικό συνέδριο. Όπως ξέρετε, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, ο Τσέχος Πρωθυπουργό είναι ιδιοκτήτης μιας εταιρείας η οποία λαμβάνει ευρωπαϊκά κονδύλια από διάφορα προγράμματα. Πέρσι το Δεκέμβριο, ο Επίτροπος Έτιγκερ έκανε κάποιες ε, παρατηρήσεις και σημείωσε ότι η εταιρεία συνεχίζει να λαμβάνει ευρωπαϊκά κονδύλια και εξακολουθεί να είναι ιδιοκτησία του Τσέχου Πρωθυπουργού. Οι ελεγκτέ Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωσης βρήκαν αυτού τους δεσμούς με τον Τσέχο Πρωθυπουργό και διάφορα προβλήματα όσον αφορά την άντληση των κονδυλίων. Δυστυχώ, τα προκατακτικά ευρήματα δεν δημοσιεύονται από το τσεχικό κράτο. και θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να δημοσιεύσει τα τελικά συμπεράσματα των ελέγχων αυτών για την ιδιοκτησία της εταιρείας αυτής και τον Τσέχο Πρωθυπουργό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Πάλμερ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ε, ευχαριστώ. Οι χαμηλοεισοδηματίες ε, θα επηρεαστούν δυσανάλογα από την αύξηση της τιμής των τροφίμων. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Αυτά τα λέει το σενάριο της κυβέρνησης για ένα Brexit χωρίς συμφωνία. Είχα πάει λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα σε μια τράπεζα τροφίμων, όπου μας λένε ότι η ζήτηση αυξάνεται μήνα με το μήνα. Συζητήσαμε το ότι τα παιδιά δεν λάμβαναν αρκετά, αρκετό φαγητό επειδή είχαν κλείσει τα σχολεία. Αυτά δεν είναι τρομοκρατία, είναι η πραγματικότητα. Ο Πρωθυπουργό, ο κ. Τζόνσον, μπορεί να έφαγε μια χαρά στο Λουξεμβούργο σήμερα, αλλά οι φτωχές οικογένειες στην Βρετανία που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα θα δυσκολευτούν πάρα πολύ έτσι όπως κουτρουβαλάει προς ένα Brexit ο κύριος Τζόνσον. Θα βρεθούν και άλλα παιδιά κάτω από το όριο της φτώχειας. Πηγαίνουν οι γονείς να ζητιανέψουν φαΐ. Δεν μπορούμε λοιπόν να επιτρέψουμε Brexit χωρίς συμφωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μπότος από το Renew Europe. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το μοναδικό εγχείρημα κατά την άποψή μου είναι το καλύτερο που συνέβη ποτέ σε αυτήν την Ήπειρο. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Αυτό το λένε πολύ συχνά, αλλά παρόλα αυτά τα σημαντικότερα μέτρα για την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας δεν έχουν ληφθεί. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να υπάρξουν λύσεις. Οι λύσεις όμως ε, είναι εμβαλωματικές. Ε, ε, υπάρχουν οι ειδικοί οι οποίοι θα ήθελαν να εργαστούν, έχουν εμπειρία στην προστασία του περιβάλλοντος και έχουν και εμπειρία σε επιτυχημένα προγράμματα τα οποία τα έχουν εφαρμόσει από κοινού με άλλα κράτη-μέλη. Γιατί λοιπόν ε, περιμένουμε τόσο πολύ, δεν μπορούμε να περιμένουμε ε, να συσταθεί ένας ειδικό οργανισμός, ως εκ τούτου χρειαζόμαστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οικονομική Υποστήριξη για να μπορούν αυτοί οι ειδικοί, όπως σας είπα, να πιάσουν δουλειά. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, θα πρέπει να διοχετευτούν τα κονδύλια το συντομότερο δυνατόν για να καταρτιστούν προγράμματα και για να στηρίζονται με τον ίδιο τρόπο όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για την προστασία του περιβάλλοντος. Χρειαζόμαστε περισσότερες συζητήσεις και περισσότερες ε, πράξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενος ε, ομιλητής από τους πράσινους παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, για πάνω από 30 χρόνια η Ιαπωνία ε, τώρα πλέον έχει αρχίσει ε, την, το εμπόριο της φώκιας ε, το οποίο διαταράσει τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Το κοινοβούλιο αυτό έχει καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απευθυνθεί στην Ιαπωνία με στόχο να πάψει αυτή την πρακτική και είναι ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την Ιαπωνία δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις για το εμπόριο της φάλαινας. Όμως δεν μπορούμε να είμαστε αδρανείς, δεν μπορούμε να επιτρέπουμε την σφαγή των φαλενών για καθαρά ε, κερδοσκοπικούς ε, λόγους. Έτσι λοιπόν εμείς ε, γράψαμε μία επιστολή στον Επίτροπο Εμπορίου ε, ερωτώντας κατά πόσον όλα αυτά είναι συμβατά με την Εμπορική Συμφωνία περί βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, γι' αυτό λοιπόν καλούμε να εφαρμοστεί άμεσα μία διαδικασία να σταματήσουμε να εφαρμόζουμε εμπορικές συμφωνίες όταν αυτές παραβιάζουν ακόμα και τις ε, καλύτερες περιοριστικές μας ε, πρακτικές. Πολύ ωραία. Επόμενος ο ο κύριος Γκίντο ε, Ρέιλ. Κύριε Πρόεδρε, είμαι νέος εδώ και εκπλήσωμαι για πάρα πολλά και με εκπλήσει κυρίως αυτό που βρήκα στο διαμέρισμά μου, ενώ το διαμέρισμα στις Ξέρετε τι, μια λάμπα. Ε, θα θυμάστε πολλοί από εσά, ε, πριν από 10 χρόνια απαγορεύτηκε αυτό το είδο τη ε, λάμπα. Πριν από 100 χρόνια βέβαια μα φώτισε. Με τώρα όμω την έχουμε απαγορεύσει. Γιατί? Για να εξοικονομηθεί ενέργεια. Μέσα στη λάμπα υπάρχει υδράργυρος και επειδή τους Βρυξελιώτες του συμπαθώ, πρέπει να σου πω ότι οι Βρυξελιώτες ε, δεν πολύ ενδιαφέρονται για αυτές τις απαγορεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό και αυτό, γιατί στην Ευρώπη έχουμε ε, πολίτες ε, οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν μόνοι τους τι θα αγοράζουν και πώς θα ζουν. Είναι όριμοι και ενήλικες. Ευχαριστούμε κύριο Τζαμπάνσκι. ECR. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, Έχουμε εδώ πέρα μια κατάσταση στην ε, Τουρκία η οποία δεν εφαρμόζει την ε, συμφωνία και απειλεί την Ευρώπη με παράνομους ε, μετανάστες. Και στην Τουρκία αυτή θέλει η Volkswagen να φτιάξει και ένα δεύτερο εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων. Αυτό είναι άδικο. Δεν είναι δυνατόν να γίνει. Λοιπόν, ερωτώ τον Πρωθυπουργό της Κάτω Σαξονίας. Ε, πότε λέτε την αλήθεια, όταν μιλάτε σε εμά ε, ή όταν μεταφέρετε την παραγωγή σε χώρες ε, όπου δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα μια απάντηση και από την κυρία Φόντερ για το θέμα αυτό δεν είναι δυνατόν να επιβραβεύουμε το καθεστώς Ερντογάν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τόμακ είναι ο επόμενος ομιλητής. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα συζητάμε για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό εγώ ήθελα σήμερα να μιλήσω για ανθρώπινα δικαιώματα που δεν τηρούνται στην υπερνηστερία, που είναι λιγότερο από 100 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ρουμάνοι χάνουν την αξιοπιστία τους. Εγώ έχω πάει αρκετές φορές και δεν έχω μπορέσει να μπω στην ε, Ρωσία εξαιτία των πολιτικών μου απόψεων. Μου το απαγορεύουν αυτοί που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα καταπατούν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν που είναι υπέρ της ε, δημοκρατίας δεν μπορεί να εγκαταλείψει την ε, περιοχή και τους πολίτες της. Γι' αυτό και ζητάω από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να εκπονήσει έκθεση όσον αφορά την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην υπερδνηστερία που αποτελεί μέρος της δημοκρατίας της Μολδαβίας και ε, βρίσκεται υπό παράνομη κατοχή από τη Ρωσία. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Άβραμα έχει τώρα το λόγο και μέρος των ε, ε, Δημοκρατών. Συνάδελφοι, τώρα που μιλάμε για την βιωσιμότητα, την αηφορία και την βιοπικιλότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει ότι εξαφανίζονται κάποια είδη και ένα από αυτά είναι ο ξύριχος, το ψάρι στον ε, Δούναβη. Έχει επιζήσει από τους δεινόσαυρους, όμως τώρα εξαφανίζεται σιγά σιγά γιατί υπάρχει υπερβολική αλίευση από τους Ουκρανούς ε, αλείς που δεν σέβονται την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και έτσι κινδυνεύει το κλίμα επίσης. Από τα είδη που υπάρχουν στην Ρουμανία, δύο έχουν ήδη εξαφανιστεί και για τα υπόλοιπα είδη υπάρχουν ελάχιστα είδη, για κάποιο είδος μόνο εννέα ε, αρσενικά και κανένα θηλυκό. Υπάρχουν σχετικές συμβάσεις που όμως δεν λειτουργούν ε, η οικονομική ζημιά επίσης είναι τεράστια. Γι' αυτό ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να πάρει μέτρα προκειμένου να σώσει τον οξύριχο. Εμείς ζητούμε χρηματοδότηση πριν εξαφανιστούν αυτά τα είδη. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Στεφανούτα έχει τώρα το λόγο από το Ρινιού. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής εξαρτάται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις χώρες μέλη, προκειμένου να τηρούν τους κανόνες. Ε, θα σας δώσω παραδείγματα όπου δεν τηρείται το άρθρο 11 της συνθήκης που μιλάει για γενική συμμόρφωση από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να λάβει υπόψη της στα μέτρα που υιοθετεί την κλιματική αλλαγή. Έχουμε πρώτα απ' όλα το πακέτο κινητικότητας το οποίο θα ε, οδηγήσει και μάλιστα η ρύθμιση αυτή προβλέπει ότι τα φορτικά πρέπει να επιστρέφουν στην έδρα τους. Αυτό σημαίνει ότι θα επιστρέφουν άδεια πάρα πολλά φορτηγά και θα κυκλοφορούν άδεια στους δρόμους μας. Με αύξηση βέβαια των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ως συνέπεια. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και ένα δεύτερο παράδειγμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει την πρόσβαση στην δικαιοσύνη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αυτό παραβιάζει μάλλον τη συνθήκη του αρχού στο σημείο 9. Αν θέλουμε λοιπόν να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, πρέπει να κοιτάξουμε τι κάνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν μιλήσουμε για τους άλλους. Ευχαριστούμε πολύ. Η επόμενη είναι η κυρία Ρίμπα η Χινέρ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, υπάρχουν νέοι που βρίσκονται στην φυλακή πολλές μέρες επειδή ανακατεύτηκαν σε έναν καυγά στην Ισπανία όπου συμμετείχαν και χωροφύλακες εκτός ορών υπηρεσίας. Ε, πρόκειτο, είπε το δικαστήριο, για τρομοκρατική ενέργεια και ενώ το δικαστήριο τους κατηγόρησε και τους επέβαλε ποινές 2 με 8 χρόνια. Και όμως το 2017 διάφοροι ευρωβουλευτές ζήτησαν να παρέμβει ο πρόεδρος Γιούγκερ. Και ο αντιπρόεδρος Τίμερμαν είπε ότι παρακολουθεί από κοντά την περίπτωση. Αναφέρεται ο κίνδυνος να εκλαμβάνεται λάθος ε, το περί Εδώ γίνεται μια διάκριση σε βάρος των κατηγορούμενων εξαιτία της ιδεολογίας τους. Υπάρχει δίκη πάλι σε τρεις μέρες. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει την υπόθεση αυτή και να υιοθετήσει ό,τι μέτρα χρειάζονται προκειμένου να μην υπάρχουν παραβιάσεις από το Ισπανικό κράτος, παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Η κυρία Σαρδόνε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους σας. Ε, θα ήθελα να απευθυνθώ στον Πρόεδρο κύριο Σασόλη ε, με την ιδιότητά του του Προέδρου του Κοινοβουλίου. Τώρα βέβαια δεν είναι εδώ στην αίθουσα. Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπε όταν ανέλαβε το αξίωμά του και θέλω να σας πω ότι άκουσα να έχει μία έμονη ιδέα με τη μετανάστευση. Είπα προηγουμένως ότι είμαι υπέρ των ΜΚΟ, αλλά βεβαίω ε, δεν ξεχνάω ότι διευκολύνουν τις αποβάσεις, αποβιβάσεις ε, των μεταναστών, αλλά θα πρέπει να έχουμε και κατά ότι περισσότεροι από αυτούς που μπαίνουν στην Ιταλία είναι παράνομοι και δεν έχουν δικαίωμα να ε, αποβιβάζονται. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, όπου η Ιταλία χάρη της αριστεράς ε, έγινε ο καταβλισμός ε, της Ευρώπης, θα περίμενα από τον πρόεδρο να είναι λιγάκι πιο μετριοπαθής. Όχι να είναι ο παντός των μεταναστών χωρίς καμία συστολή. Έχω ακούσει κενά λόγια πάρα πολλά μετά από όλα αυτά τα χρόνια, όπου δεν έγινε τίποτα απολύτως από πλευρά τη Ευρώπη. Εμεί θέλουμε μια Ευρώπη που να μην είναι τόσο εστιασμένη στο να μιλάει για την ενσωμάτωση, αλλά να προσπαθεί να προστατεύει τα δικά τη ε, τα σύνορα. Θέλω λοιπόν να πω ότι κουραστήκαμε πια από μια Ευρώπη η οποία επικρίνει την Ιταλία και η οποία όμω δεν έχει βοηθήσει καθόλου, μα κατά το ελάχιστον, ούτε κατά το ελάχιστον, τη δική μα τη χώρα. Ευχαριστούμε. ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύμφωνα με το άρθρο 172, κατά τη διάρκεια των ομιλιών του ενός λεπτού, ε, δεν μπορεί να γίνει ερώτηση με μπλε κάρτα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τέλτς από το ECR είναι ο επόμενος, αλλά δεν τον βλέπω. Οπότε περνάμε στον κύριο Μπασέσκου από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευστήσω την προσοχή σας σε κάτι το οποίο είναι γνωστό σε όλους μας αλλά δεν το συζητάμε. Αναφέρομαι στο ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όλο και λιγότερη σημασία στην παγκόσμια σκηνή, στην εξωτερική πολιτική. Θα ήθελα να γίνει μια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο στην Επιτροπή Εξωτερικών και στην Κομισιόν για να βρεθούν κάποιες λύσεις έτσι ώστε Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ένας πόλος παγκόσμιας ισχύω όπως η ΕΠΑ, η Κίνα και η Ρωσική Ομοσπονδία. Αν δεν έχουμε έναν τέτοιο στόχο, κινδυνεύουμε να γίνουμε ένας πολιτικός και οικονομικός χώρος ο οποίος ε, θα υφίσταται την παγκοσμιοποίηση και δεν θα την ε, διαμορφώνει. Ε, εκ μέρους των 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Γι' αυτό θεωρώ ότι είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε, να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και να συμμετέχουμε και εμείς αποφάσεις που θα διαμορφώσουν την παγκοσμιοποίηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο έχει η κυρία Γκραπίνη. Σας ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να μιλήσω για την διακίνηση ανθρώπων, ανηλίκων, γυναικών. Υπάρχουν διασυνοριακά δίκτυα, γι' αυτό συνέταξα και μια επιστολή προς τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, αλλά θα ήθελα να ζητήσω και από την Κομισιόν να κάνει μια έρευνα σε όλα τα κράτη-μέλη, μέσω της Europol, παραδείγματος χάρη. Γιατί μια χώρα δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα αυτό μόνη της. Να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ασφάλεια για τους πολίτες, δικαιώματα για τους πολίτες. Και αυτό σημαίνει ασφάλεια. Να σας δώσω ένα παράδειγμα στη Φιλανδία. Τα παιδιά που είναι στα ιδρύματα δεν έχουν δικαίωμα να εκφράσουν άποψη παρά το ότι στα 12 χρόνια σύμφωνα με τον νόμο μπορούν να εμφανίζονται στο δικαστήριο. Ε, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο την οικονομική ανάπτυξη αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τις ανατολικές χώρες αλλά και τις ε, δυτικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. κυρία Γιάρο Κακάνο, κατόπιν από το ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στην 30η επέτειο του τη στιγμή εκείνη πριν από 30 χρόνια ενό πικνίκ ε, που ήταν σύμβολο ελευθερίας και ειρήνης. Ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι είχαμε ενότητα τότε και ε, δυστυχώς όλα αυτά ξεχνιούνται και η Ευρωπαϊκή Ένωση Όχι, Υπάρχουν 120 εκατομμύρια φτωχοί άνθρωποι που δεν έχουν τα βασικά της υγιεινής ε, στο σπίτι τους. Πρέπει λοιπόν ε, να δούμε αυτό το θέμα στο πρόγραμμα των 100 ημερών της Νέας Κομισιόν. Αν δεν βρεθεί μια λύση για τη φτώχεια, οι δημοκρατίες μας ε, θα παραμείνουν χωρίς ουσία και δεν θα μπορούν να επιβάλλουν τα βασικά δικαιώματα των πολιτών τους και βλάπτει και την ευρωπαϊκή οικονομία. Σας παρακαλώ να κάνετε κάτι το οποίο θα είναι αντάξιο των όσων έγιναν πριν από 30 χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Κυρία Σπουρακ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα έχετε ακούσει τη βρώμικη εκστρατεία κατά δικαστών που επικρίνουν την πολωνική κυβέρνηση. Πρόκειται για το σκάνδαλο Πίμπιακ. Και ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης ε, παρετήθηκε μετά από διάφορες ανακοινώσεις και διάφορα ψεύτικα μηνύματα. Πρόκειται για εκστρατεία εκφοβισμού που συντονίζεται από το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατά δικαστών που θέλουν να επιβληθούν στην πολωνική δικαιοσύνη. Ο Γενικός Συγγελέας είναι συγχρόνος και Υπουργός Δικαιοσύνης και επιβλέπει αυτές τις διαδικασίες. Οπότε ήρθε η ώρα να υπάρξει μια δική εξεταστική επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διασφαλίσει ανεξαρτησία στις σχετικές διαδικασίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Άλβαρες. Ευχαριστώ. Η Ισπανία επέστη μια από τις χειρότερες πλημμύρες της ε, ιστορίας της. Η Ανδαλουσία, η Μούρσια, η Καστίγια Λαμάντσα υπέφεραν αυτοκινητόδρομοι, κόπηκαν εντελώς. Ε, καταστράφηκαν υλικά 18 ετών και πολλές καλλιέργειες και ο κόσμος αναγκάστηκε να φύγει από τα σπίτια του. Χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές. Τώρα είναι που η Ευρώπη πρέπει να δείξει την αλληλεγγύη της με τους χιλιάδες Ισπανούς που υπεφέρουν από τις συνέπειες των πλημμυρών αυτών. Και θέλω να υποφεληθώ από αυτή την ευκαιρία για να πω ότι θέλουμε να βοηθήσουμε. Θέλω να αναγνωρίσω επίσης την βοήθεια όλων των υπηρεσιών που την προσέφεραν. Η Ευρώπη πρέπει να συνεισφέρει λοιπόν με όλα τα μέσα που διαθέτει για να βοηθήσει να αποκατασταθούν οι ζημιές και να βοηθήσει επίσης ώστε να επανέλθει η κανονικότητα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Καρσία Νταμπλάνκο, ε, Σοσιαλδημοκράτης. Ευχαριστώ η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι κάτι που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από αυτό εξαρτάται και η επιβίωσή μας. Όμως, δεν θα πρέπει να βοηθήσουν μόνο κάποιες ε, περιοχές της Ευρώπης. Οι περισσότερες χώρες κάνουν πράγματα, επιταχύνουν τις ε, διαδικασίες και πολλές από αυτές τις χώρες έχουν προχωρήσει και στην οικονομική μετάβαση των περιοχών αυτών. Σε πολλές δεν έχουν πετύχει όμως τα πράγματα. Ήρθε η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει περισσότερο τις εθνικές κυβερνήσεις και να προσφέρει κονδύλια, όχι μόνο οικονομική όμως στήριξη, να προσφέρει και πραγματογνωμοσύνη και τεχνική αρρωγή. Έφτασε η στιγμή στις ε, μελλοντικές ε, δημοσιονομικές προοπτικές να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη εκβιομηχανοποιήθηκε με τον άνθρακα. Γενιές και γενιές Ευρωπαίοι έχασαν την υγεία τους ή τη ζωή τους στα ορυχή άνθρακα. Τώρα χρειάζεται κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και δικαιοσύνη απέναντι στην ιστορία. Ο κύριος Χάισελ από τους Σοσιαλδημοκράτες, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε ότι πρέπει να είναι απολύτως σαφές ε, ότι δεν υπάρχει κανένας μοιραίος πόλεμος η Ευρώπη εκτέθηκε στον πόλεμο και αυτό ήταν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Οι Ναζί επιτέθηκαν στην Πολωνία το 41, το Σεπτέμβριο του 41 και αυτή, αυτή ήταν η έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όμως πόλεμοι υπήρχαν και αλλού κατά το παρελθόν. Δεν αναφέρεται αυτό συχνά Αλλά ας μην ξεχνάμε τη συνθήκη Ριμπεντόφ Μόλοτοφ. Αυτό πρέπει να το αναφέρουμε. Πολλοί το ξεχνούν. Και ας μην ξεχνάμε και τη συνθήκη του μονάχου ένα χρόνο πριν συνήθει αυτή την επίθεση στην Πολωνία. λόγω αυτής της ε, διαδικασίας η Μεγάλη Βρετανία και, και ο Χίτλερ επέτρεψαν στον ε, Χίτλερ να ε, διεχοτομήσει την Τσεχοσλοβακία και να υφαρπάξει ένα κομμάτι της Σλοβακίας. Αυτό λοιπόν το βήμα επέτρεψε στο Χίτλερ να μετακινηθεί προς Ανατολάς, Drang nach Osten. Θέλω να πω ότι ο πόλεμος σήμερα δεν είναι κερδοφόρος και ως εκ τούτου οφείλουμε να αγωνιζόμαστε για την ειρήνη. Ο κύριος Νικολάου τώρα. Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Πρόεδρε, οι κυβερνήσει προχωρούν σε αντιδραστικέ αλλαγέ στου νόμου για τη λειτουργία των εργατικών συνδικάτων. Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να επιβάλλει συνδικαλιστικό νόμο, ο οποίο περιλαμβάνει ηλεκτρονικά μητρώα στα συνδικάτα, φακέλωμα των εργαζομένων. Καταστρατηγεί τα καταστατικά του εισάγει την ηλεκτρονική ψηφοφορία για την απεργία χτυπώντα τι συλλογικέ ζωντανέ διαδικασίε φέρνοντα την κατάργηση του απεργιακού δικαιώματο συνεχίζοντα την αντιλαϊκή πολιτική τη προηγούμενη κυβέρνηση που άνοιξε το δρόμο με εμπόδια στην απεργία. παρόμοια μέτρα εφαρμόζονται σε άλλα κράτη μέλη τη ευρωπαϊκή ένωση όπω είναι η ιταλία η βρετανία το βέλγιο η σουηδία. η ευρωπαϊκή ένωση το κεφάλαιο οι κυβερνήσει του δυναμώνουν την αντεργατική επίθεση ανησυχούν για το ενδεχόμενο μια νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση προετοιμάζονται δυναμώνοντα την καταστολή εργατικών αγώνων υπονομεύοντα τα συνδικάτα και τι αγωνιστικέ διεκδικήσει προσπαθώντα να περάσουν τον επικίνδυνο για του εργαζόμενου κοινωνικό εταιρισμό. Οι εργαζόμενοι αντιστέκονται σε αυτέ τι αντεργατικέ μεθοδεύσει, οργανώνουν την πάλη του, όπω γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αντιπαρατίθενται μαζικά με την κυβερνητική πολιτική. Παλεύουν για αγωνιστικά συνδικάτα που θα υπερασπίζονται τα εργατικά δικαιώματα και θα συγκρούονται με τις δυνάμεις του κεφαλαίου και την εξουσία τους. Ευχαριστούμε.